Πολύ καλή σας μέρα, αξιότιμοι συνάδελφοι. Κυρίσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, μέρα πέμπτη. Έχω μια ανακοίνωση να σας κάνω. Οι αρμόδιες ισπανικές αρχές ε, κατέθεσαν ε, στον πρόεδρο ε, έτοιμα ε, άρση ασυλίας και κυρίας Κάραπος Άρντεδιός για να ξεκινήσει ποινική διαδικασία. Σύμφωνα με το κανονισμό θα ε, διαβιβαστεί το αίτημα αυτό στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου. Ερχόμαστε λοιπόν στο πρώτο θέμα στη μέση διάταξη, προφορική ερώτηση ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο, ο ρόλο των γεωργών στις αγροτικές περιοχές. Γνωρίζετε ότι μπορείτε να ζητήσετε αυθόρμητα το λόγο και ε, με τις γαλάζιες κάρτες και με τον παραδοσιακό τρόπο και με τον ηλεκτρονικό. θα δώσω το λόγο στο συντάκτη της ερώτησης πρώτα, τον συνάδελφο κύριο Λιντ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επιτροπέ, η Γεωργία σημαίνει πάθος. Δεν είναι απλώς έτσι, ένα επάγγελμα όπως όλα. Όπως πας και κάνεις τη δουλειά σου, πας στο γραφείο και φέρνεις και τίποτα λεφτά στο σπίτι για να ζήσεις την οικογένειά σου. Δεν είναι αυτό η γεωργία. Οι αγρότες έχουν αποστολή. Θέλουν να παράγουν τα καλύτερα, ε, υψηλότερης ποιότητας βιώσιμα τρόφιμα. Και το κάνουν ήδη από σήμερα θέλουν να εφοδιάζουν τους καταναλωτές, άνδρες και γυναίκες, με τα καλύτερα τρόφιμα. Και θέλουν να αναπτύσσουν και την επιχείρησή τους, την εκμετάλλευσή τους, έτσι ώστε να μπορούν κάποια στιγμή να τη μεταβιβάσουν στην επόμενη γενιά. Συχνά ακούμε ιστορίες γενεών αιώνων όπου οι άνθρωποι ζουν στις ίδιες εκμεταλλεύσεις και παραδίδουν τη γη τους στην επόμενη και στη μεθεπόμενη γενιά. Θέλω να σας αναφέρω για την προσωπική μου ιστορία. Είμαι 42 ετών, γι' αυτό σας μιλάω για πάθος. Πάνω από 30 χρόνια δουλεύω. Για ποιο λόγο? Διότι έχω εργαστεί ε, μαζί με τους γονείς μας ε, στην οικογενειακή μας εκμετάλλευση από μικρό παιδί. Ε, ετάιζα τα μοσχάρια, άρμεγα τις αγελάδες, έπιανα και το δίκρανο και τους έβαζα σανό ε, και έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου από μικρό αγόρι για να συνεχιστεί αυτή η δραστηριότητα και να μπορέσουμε να παράγουμε τα καλύτερα τρόφιμα. Και σας λέγω ότι καμιά φορά ήταν δύσκολο αυτό όταν οι άλλοι το καλοκαίρι πήγαιναν στην πισίνα ας πούμε και εγώ έπρεπε να βοηθήσω στο, ε, αγρότημα, στο αγρόκτημα. Αλλά αυτό το έκανα όχι μόνο γιατί είχα αυτό το πάθος, αλλά γιατί υπήρχε και αναγνώριση, εκτίμηση έπιανε τόπο η δουλειά μας. Μας σεβότανε ο κόσμος στο χωριό για όλα αυτά που κάναμε και για όλα αυτά που έκανε η δική μας οικογενειακή εκμετάλλευση. Αυτός ο σεβασμός λοιπόν, η εκτίμηση, η αναγνώριση όλο και περισσότερο φθήνει και εξαφανίζεται και θα πρέπει να προσέξουμε ε, κάνουμε διάφορες συζητήσεις ε, ε, για τη γεωργία. Δεν θα πρέπει να καθίζουμε τους αγρότες στο εδόλιο ότι ρηπαίνουν το περιβάλλον, δηλητηριάζουν τον κόσμο. Θα πρέπει να του πούμε ότι κάνετε καταπληκτική δουλειά, αλλά θα πρέπει ακόμα καλύτερα να γίνει. Θα πρέπει να τους βοηθήσουμε να γίνει καλύτερη η δουλειά τους. Και να μην αρχίσουμε τους επόμενους μήνες ένα όργιο απαγορεύσεων, ένα όργιο ρυθμίσεων. Θα πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα για περισσότερη προστασία του κλίματος. Να μπορούν οι αγρότες, ας πούμε, να ε, παράγουν βιολογικό ε, λίπασμα ε, με λιγότερα φυτοκτόνα, με λιγότερα φυτοφάρμακα, αλλά με κίνητρα, όχι με απαγορεύσεις, όχι με φόβητρα. Στην Ευρώπη έχουμε πολύ υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα Πώς προστατεύουμε τους αγρότες μας πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα καταφέρουμε κύριε Επίτροπε οι άλλοι να μας ακολουθήσουν παγκοσμίω, να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας, τις εμπορικές συμφωνίες. Θα πρέπει να τις μετεξελίξουμε. Δεν θα πρέπει να έχουμε πρότυπα προϊόντος, αλλά πρότυπα παραγωγής. Και επίση θα πρέπει να κυριαρχήσει άλλο ένα ζήτημα σε αυτή τη συζήτηση και τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο ή από το δίκρανο στο πυρούνι. Ε, πρέπει να παίζουν και οι καταναλωτέ αυτό το παιχνίδι. Χρειάζεται ε, αλλαγή νοοτροπία των καταναλωτών. Στη χώρα μου το 72% των καταναλωτών λέγουν ότι είμαι πρόθυμος ε, για περισσότερη προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος να πληρώσω κάτι παραπάνω αλλά αυτά τα λένε ε, στη θεωρία, αλλά όταν φτάνουν στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, μόνο το 16% είναι πρόθυμο να πληρώσει περισσότερο. Θα πρέπει λοιπόν και οι καταναλωτές να αλλάξουν λογική και νοοτροπία και να βάλουν το χέρι πιο βαθιά στη τσέπη. Σε συνεργασία ε, με τους αγρότες θα πρέπει να δράσουμε. Το περασμένο Σαββατοκύριακο είχα πέντε εκδηλώσεις με αγρότες και κύριε Επίτροπε έχουν θορυβηθεί πάρα πολύ, ανησυχούν πάρα πολύ ε, ότι τους παραγωνίζουμε, ότι αποφασίζουμε ρήμην του. Θα πρέπει να τους πούμε στη συζήτηση αυτή ότι δεν είστε τμήμα του προβλήματο αλλά τη λύση. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση εδώ στο Κοινοβούλιο ε, σε, χώρα, σε ώρα μάλλον υψηλής ακροματικότητας, 9 το πρωί, στο κέντρο της συζήτησης είναι ο αγρότης, πριν ε, αρχίζει να υλοποιείται η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο και πριν καν δημοσιευθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ο ε, Επίτροπος κύριος Βοητσεχόφσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο Λίντς και τους ευρωβουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας που οργάνωσαν αυτήν την τόσο σημαντική συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που εκτιμούν πολύ και που ανέμεναν οι αγρότες μας. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω για την στρατηγική αυτή από το χωράφι στο πιάτο. Να ξέρετε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Τον Μάρτιο θα ξέρουμε περισσότερα πράγματα. Δεν ανακοινώθηκε η Πράσινη Συμφωνία στο μεταξύ και πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο για βιώσιμη παραγωγή τροφίμων. Οι Ευρωπαίοι αγρότες παίρνουν μεγάλη σημασία μέσα σε αυτή τη στρατηγική. Το σχέδιο θα προτείνει διάφορα φιλόδοξα προγράμματα όσον αφορά την χρήση φυτοφαρμάκων για παράδειγμα, ε, παρασιτοκτόνων αλλά και αντιβιωτικών που πρέπει να χρησιμοποιούνται πολύ λιγότερο από ό,τι μέχρι τώρα. Θα υπάρξουν περισσότερες διευκρινήσεις επίσης για την βιολογική γεωργία που θα προωθηθεί. Θα δώσουμε μεγάλη σημασία επίσης στην ποιότητα ε, του δάφους των υδάτων και του αέρα ακόμα. Οι αγρότες θα πρέπει να παράγουν με περισσότερο βιώσιμο τρόπο και θα προωθούν την ανθρώπινη υγεία περισσότερο και θα φροντίσουν για την άμβληση της κλιματικής αλλαγής. Δεν είναι δυνατόν να ξεχάσουμε τους αγρότες, να τους αφήσουμε πίσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει και όλοι μας πρέπει να τους βοηθήσουμε. 10 εκατομμύρια Πολωνοί αγρότες προσφέρουν τρόφιμα με ασφάλεια στην ε, Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να τους ευχαριστούμε πραγματικά σε καθημερινή βάση για την προσπάθειά τους, για την βούλησή τους να αντιμετωπίσουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα ζώα, με το έδαφος, με τη γη. Να ξέρετε ότι δεν το κάνουν όλοι. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα επίσης με την διαδοχή, δηλαδή πώ θα αντικατασταθούν οι αγρότε οι οποίοι εγκαταλείπουν τη δραστηριότητά του. Η επισητιστική ασφάλεια και η ασφάλεια των τροφίμων είναι κάτι εξίσου σημαντικό όπως είναι η άμυνα ή όπως είναι η ενέργεια. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει προστασία, ότι υπάρχει ασφάλεια, πρέπει να νοιαζόμαστε για τους αγρότες μας και να τους προσφέρουμε καλές συνθήκες εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό και για τη γεωργική πολιτική αλλά και για άλλες πολιτικές. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις ερωτήσεις που υποβάλλατε σε αυτή την ερώτηση. Ε, ρωτάτε πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει ότι ο κόσμος στην Ήπεθρο και οι αγρότες θα εξακολουθούν να έχουν σημασία και πώς οι μελλοντικέ φιλοδοξίες και στόχοι μας θα ληφθούν υπόψη, όπως επίσης και οι προκλήσεις. Πώς θα διασφαλίσουμε επίσης ικανοποιητικά έσοδα για τους αγρότες και καλές συνθήκες πρέπει να αλλάξουν πολιτικές στρατηγικές. Όντω και οι ίδιοι αγρότε αναρωτιούνται για όλα αυτά. Πρόσφατα συναντήθηκα με πολλού από αυτού στην Κροατία, στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Πολωνία επίση. Και πολύ σύντομα θα πάω και στη Γαλλία να συναντηθώ με αγρότε, αλλά και σε άλλε χώρε. Συναντήθηκα επίσης με εκπροσώπους Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών Αγροτών και αντιλαμβάνονται ότι η βιώσιμη παραγωγή τροφίμων είναι κάτι αναγκαίο. Συνεπώς, αν τώρα δεν έχουμε βιωσιμότητα, αν δηλαδή υπάρχει υπερβολική συγκέντρωση της παραγωγής τροφίμων, δεν είναι επειδή το θέλουν, αλλά έχει να κάνει με τις οικονομικές συγκυρίες. Αναγκάστηκαν για να μπορέσουν να κερδίσουν τα προστοζήν. Οι αγρότες λοιπόν πρέπει να συμμετέχουν σε πιο εντατική παραγωγή. Αυτό πρέπει να αλλάξει και πρέπει να τους βοηθήσουμε να το αλλάξουν και η γεωργία να αλλάξει. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο δεν πρόκειται να επιβληθούν με το ζόρι. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Λίντς. Χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεται δηλαδή ο κατάλληλος προϋπολογισμός ε, στην ε, ΚΑΠ, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, να έχουμε έναν ισχυρό, έναν δίκαιο προϋπολογισμό με δίκαια κατανομή. Και χαίρομαι που υπάρχει συνειδητοποίηση για τον προπολογισμό αυτό και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στις χώρες μέλη. Τρεις υπουργοί, κύριε από τη Γερμανία, η από τη Γαλλία, και επίσης ε, Σπανός υπουργό Γεωργίας δήλωσαν πράγματα που έχουν μεγάλη σημασία για μένα. Και τι είπαν, είπαν ότι χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα, περισσότερα κονδύλια για την ε, ΚΑΠ. Και στο τέλος ε, Ιανουαρίου στην Σύνοδο Υπουργών Γεωργίας και άλλοι υπουργοί εξέφρασαν την ίδια άποψη. Και εγώ τη στηρίζω επίσης. Πράγματι χρειαζόμαστε έναν άνετο προπολογισμό για την ΚΑΠ που να είναι δίκαια κατανεμημένος. Έχουμε φιλόδοξους στόχους στην ε, πράσινη αυτή συμφωνία και στην ε, στρατηγική μας από το χωράφι στο πιάτο και πρέπει να πολεμήσουμε για αυτούς. Χρειαζόμαστε επίσης χρήματα και για οικολογικά προγράμματα στον πρώτο πυλώνα. Κυρίως στις χώρες εκείνες που είναι χαμηλές οι άμεσες ενισχύσεις. Επίσης πρέπει να κάνουμε κάτι και για την προστασία των ζώων και για το περιβάλλον στο δεύτερο πυλώνα. Και αυτά είναι σημαντικά για κάποια άλλη ομάδα χωρών. Θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι αγρότες αντιλαμβάνονται την ανάγκη για βιώσιμες πρακτικές. Να έχουμε λιγότερο εντατική δηλαδή γεωργία και να έχουμε σε εθελοντική βάση εισαγωγή μέτρων για προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων. Να ξέρετε ότι θα λάβουμε πολύ σημαντικές αποφάσεις όταν αποφασίσουμε για το δημοσιονομικό πλαίσιο της επόμενης περίοδου. Πρέπει επίσης να μην ξεχνάμε ότι οι αγρότες δεν είναι το πρόβλημα. Πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε θετικά. Είναι εκείνοι είναι οι εταίροι μας και θα μας βοηθήσουν να εφαρμόσουμε ε, τη στρατηγική μας και τα μέτρα που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Πρέπει λοιπόν να έχουν την πλήρη στήριξή μας και να τους βοηθήσουμε στις αλλαγές που προβλέπονται. Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Γεωργία πρέπει να είναι βιώσιμη, πρέπει να είναι οικολογική, πρέπει να είναι φιλική προς το περιβάλλον αλλά για να το πετύχουμε αυτό, η γεωργική πολιτική πρέπει να είναι φιλική και προς τους αγρότες, να είναι φιλόδοξη αλλά και δίκαια συγχρόνως. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε πίτροπε. Ακολουθεί η συζήτηση. Πρώτα εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων και ο Ντόρφμαν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμε κύριε Επίτροπε, καλό είναι το γεγονός ότι γίνεται σήμερα αυτή η συζήτηση και χρειάστηκε να αγωνιστούμε γι' αυτό. Έχω την εντύπωση ότι ορισμένοι πιστεύουν αυτή η στρατηγική από το αγρότημα στο πιάτο μπορεί να γίνει ερήμην των αγροτών ή ακόμα και απέναντι στους αγρότες. Ε, και χαίρομαι που σας βλέπω εδώ. Αλλά πού είναι ο κύριος Τίμερμανς, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φαίνεται ότι αυτή η νοοτροπία επικρατεί ακόμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τολμώ να προχωρήσω και σε μία πρόβλεψη. Αν δεν ε, ε, συμμετέχουν ενεργά οι αγρότες σε αυτή τη στρατηγική θα ε, αποτύχει παταγωδός. Τώρα φαίνεται φταίνε για όλα οι αγρότες, για την κλιματική αλλαγή, ε, τα χημικά, την απώλεια της βιοπικιλότητας, για τα αντιβιωτικά. Μα είναι τελείως διαφορετική η πρακτική. Η περισσότερη συντριπτική πλειονότητα των αγροτών ε, αγωνίζονται να επιβιώσει η εκμετάλλευσή τους οικονομικά, να βρουν ε, διαδόχους και πολλές φορές σκέφτονται με πολύ μεγαλύτερη αγωνία για τη βιωσιμότητα. Οι καταναλωτές συνέχεια θέλουν πιο βιώσιμα προϊόντα, πιο υγιεινά και πιο δεν ξέρω εγώ τι και πάνε ε, ε, στο σούπερ μάρκετ και ψάχνουν την προσφορά που θα πληρώσουν ένα προϊόν και θα πάρουν τρία. Ε, πολλά χωράνε ε, εδώ ως βελτιώσεις. Μπορούμε να σκεφτούμε τη φυτοπροστασία, να σκεφτούμε τα λοιπάσματα, αλλά πώς θα γίνει αυτό να δίνουμε και μια ελπίδα ε, στους αγρότες για πρόοδο, για καινοτομία, για έρευνα, για περισσότερη γνώση. Μόνο έτσι τελικώς θα ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Γενικά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μια συμμαχία με τους αγρότες, να είναι στο πλευρό μας. Όχι απέναντι. Η δική μου πολιτική ομάδα αυτό το δρόμο θέλει να ακολουθήσει, θέλει να χαράξει αυτή τη στρατηγική μαζί με τους αγρότες, όχι εναντίον τους. Ευχαριστώ κύριε Ντόρφμαν ο συνάδελφος Δεκάστρο από την Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλδημοκρατών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, χωρί την ενεργή συμμετοχή των γεωργών μα, οποιαδήποτε προοπτική μετριασμού των κλιματικών αλλαγών τελικά θα είναι ανέφικτη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια κοινή προσέγγιση στον καθορισμό της μελλοντική γεωργικής πολιτικής, η οποία θα πρέπει να παραμείνει ευρωπαϊκή πολιτική. Και το Κοινοβούλιο μας, κύριε Επίτροπε, δεν μπορεί να χάσει την ευκαιρία να ενσωματώσει σημαντικά στοιχεία της στρατηγικής από το αγρόκτημα στο πιάτο σε μια κοινή γεωργική πολιτική που θα καθοδηγήσει την μελλοντική ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική για την επόμενη δεκαετία. Ο αγροδιατροφικός τομέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να παράσχει περισσότερες υπηρεσίες προκειμένου να πετύχουμε μια οδετερότητα σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. οι προσπάθειες αυτές δεν θα πρέπει να διέπονται μόνο από κίνητρα οικονομικά στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής, αλλά θα πρέπει να έχουμε και καινοτόμε παραγωγικές τεχνικές, όπως για παράδειγμα η βελτίωση των ποικιλιών που θα μας έπαιτρε ως τεχνική να αντικαταστήσουμε τον χημικό τομέα, τις χημικές τεχνικές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε βιωσιμότητα γεωργική, βιωσιμότητα περιβαλλοντική, αν δεν έχουμε οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει στο τομέα αυτό μια ανανεωμένη ηγετική στάση. Ευχαριστώ κύριε Τεκάστρο. Στη συνέχεια από την ομάδα Renew Europe το λόγο έχει ο κύριος Τσόλος. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, χθες εδώ, στην Ολομέλεια, συζητήσαμε για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είπαμε ότι θα πρέπει να είναι αναλογικό, να ανταποκρίνεται πραγματικά στις προτεραιότητες και τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαμε ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής ότι δεν θα πρέπει στι νέε αυτέ προτεραιότητε να αντιτάσσουμε παραδοσιακέ πολιτικέ όπω η κοινή γεωργική πολιτική. Δεν θα πρέπει να έρθει η κοινή γεωργική πολιτική σε αντίθεση και σε αντιπαράθεση με νέε ιδέε όπω για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Τα ζητήματα τα οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι σαφώ επίκαιρα, Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε αρκετά θαραλέοι, προκειμένου να δούμε πώς θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στι πραγματικέ ανάγκες και προσδοκίες τόσο των γεωργών όσο και των σημερινών καταναλωτών. Διότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ευοδοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πρόκειται να στεφθεί με επιτυχία αν δεν συμμετέχει και ο γεωργικό τομέα. Ο γεωργικό τομέα αντίθετα μπορεί να συμβάλλει προκειμένου να αποκριθούμε καλύτερα στι προσδοκίε των πολιτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πλαίσια τη πολιτική αυτή να εξασφαλίσουμε σωστά εισοδήματα για του γεωργού. Θα πρέπει οι δημόσιε υπηρεσίε να υφίστανται προκειμένου να έχουμε την καλύτερη δυνατή διαχείριση των φυσικών πόρων. Και θα πρέπει να βρούμε λύσει προκειμένου να έχουμε ένα αξιοπρεπέ εισόδημα για του γεωργού. Πέρα όμω από την κοινή γεωργική πολιτική, θα πρέπει να έχουμε και μια επενδυτική πολιτική για τον τομέα της γεωργίας. Θεωρώ ότι η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο δεν μπορεί να εφαρμοστεί ούτε θα επιτύχει αν μεμονωμένα σκεφτόμαστε μόνο κάποιου τομεί, όπω τα φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα κτλ. Η στρατηγική από το, πρόγραμμα, από το αγρόκτημα στο πιάτο θα πρέπει να αποτελεί ένα new deal, μια νέα συμφωνία για του ίδιου του γεωργού. Αυτό θα πρέπει να είναι το σημείο κίνηση. Α δούμε ποιε είναι και απαιτήσει που έχουν οι πολίτε από τη γεωργία, πώ μπορούμε να έχουμε τρόφιμα υψηλότερη ποιότητα και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλου του απαραίτητου πόρου και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της τεχνολογικής μετάβασης προκειμένου να συμβαδίζουν περισσότερο οι γεωργικέ τεχνικέ με τι προσδοκίε των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ κύριε Τσόλο. Συνεχίζουμε. Ο κύριος Ντάβιτ από την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ετοιμάζουμε μία βάση δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία για τους Ευρωπαίους αγρότες, για τους λιανικούς ε, πολιτές και το κόστος θα το επομιστούν οι χώρες μέλη, αλλά και οι ίδιοι αγρότες. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι καταλήγουμε σε μια κρίση και θα είμαστε λιγότερο ανταγωνιστικοί. Από την άλλη μεριά, ετοιμάζουμε από το διεθνές εμπόριο μία δίωδο, ένα τρόπο δηλαδή να έχουμε εισαγωγέ από τρίτες χώρες χωρίς έλεγχο και χωρίς δασμούς. Σε αυτές τις χώρες κανείς δεν θα πρέπει να συμμορφώνεται με αυτούς τους αυστηρούς κανόνες που έχουμε εμείς. Για παράδειγμα, το βόλιο κρέας, ε, τα ζώα από τα οποία προέρχονται προέρχεται το κρέας αυτό, δεν θα έχουν κανένα έλεγχο και όλο και περισσότερα τρόφιμα μας έρχονται από τρίτες χώρες. Οι αγρότες όμως πολύ σωστά έχουν κάποιες απαιτήσεις. πρώτα απ' όλα για τις τιμές που πληρώνουν. Δεν είναι δυνατόν να εισάγουμε από χώρες από τις οποίες δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις ίδιες συνθήκες παραγωγής όπως έχουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι απαράδεκτο αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Βίνερ από τους Πρασίνους Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε Βοητσεχόφσκι. Χαίρομαι που σήμερα συζητούμε για τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο ή από το δίκρανο στο πυρούνι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε τεράστια προβλήματα. Αλλιώ δεν θα βρισκόμασταν όλοι εδώ. Αποτελεί λοιπόν ιστορική ευκαιρία η στρατηγική αυτή ε, για ε, να είναι η κοινή γεωργική πολιτική πιο φιλική προς το κλίμα, να σταματήσουν να πεθαίνουν τα οικοσυστήματα, να επιστρέψει η υγεία των ζώων, η ευημερία των ζώων, η υγεία των εδαφών. Όλα αυτά τα θέματα μας έχουν φέρει εδώ εμάς. Αυτό το ζητάει και η επιστήμη, το ζητάει και ε, η κοινή γνώμη. Είναι μάλλον η τελευταία ευκαιρία να γίνει πραγματική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Βεβαίως και αγωνιούν οι αγρότες. Δηλαδή όταν μιλούμε για ποιότητα δεν θα πρέπει οι αγρότες να περιχαρακώνονται και να λένε τι θα απογίνουμε, αμάν τι θα απογίνουμε. Δεν μας βοηθάει αυτό. Δεν μπορούμε να ταμπουρωνόμαστε και να λέμε αυτά τα ξέραμε στο παρελθόν, έτσι τα έχουμε πάρει από τους παλιούς, έτσι τα κάνουμε. Ε, δεν γίνεται αυτό, πρέπει να τα αλλάξουμε. Και δεν θα πρέπει να είναι ε, στο κέντρο ε, αγρότες οι οποίοι είναι στριμωγμένοι με την πλάτη στον τοίχο και αυτοκαταργούνται. Χρειαζόμαστε και την αξιοπρέπεια των αγροτών και την αυτοπεποίθηση. Εγώ δεν χρειάζομαι επιδόματα και ελεημοσύνη ως αγρότησα. Χρειάζομαι να με βοηθήσουν ε, να είναι αναγνωρισμένο το επάγγελμά μου, να μπορώ να επιβιώσω και να ζω ανεξάρτητα από τις επιδοτήσεις. Και έχω και μια ερώτηση, κύριε Βόιτσεχόφσκι. Ε, μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε 409 κάθετος 19 ε, αναφέρει σχετικά ότι μπορεί κάθε χώρα να κάνει ε, ό,τι θέλει μέχρι να πάρει απόφαση του Συμβούλιο. Τι θα κάνετε στη Πράσινη Συμφωνία, αυτή την απόφαση θα την ευθυγραμμίσετε με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ από την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, ο κύριος Κούσμιουκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Καταρχάς, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πολύ λεπτομεριακή ανάλυση που κάνατε όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική. Θα πρέπει στην κοινή αυτή γεωργική πολιτική να ενσωματώσουμε τώρα τη στρατηγική που μας παρουσιάζεται, τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε, θεωρώ, να αντιμετωπίσουμε κάποιε νέε προκλήσει. Θα έχουμε όμω και νέε απαιτήσει αυτή τη στιγμή για του γεωργού, καθώ επίση και νέα ανώτατα όρια παραγωγή, έτσι δεν είναι. Πώ μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε όμω τι νέε αυτέ δράσει. Το Μάιο του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μία πρόταση για έναν προπολογισμό κατά 17% χαμηλότερο για την κοινή γεωρική πολιτική. Δεδομένων λοιπόν των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο γεωρικός τομέα κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Επίση μην ξεχνάμε ότι τα εθνικά στρατηγικά σχέδια, εκ μέρου των κρατών μελών δηλαδή, θα πρέπει και αυτά να ληφθούν υπόψη και χρειάζονται και αυτά βέβαια χρηματοδότηση και γνωρίζετε ότι υπάρχουν πλέον πολλές χώρες στις οποίες έχουν διαδηλώσει με έντονο τρόπο γεωργοί, βγάζοντα τα τρακτέρ μάλιστα στους δρόμους. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διασφαλίσουμε περισσότερα χρήματα για την κοινή γεωργική πολιτική, πόσο μάλλον τώρα που προτείνεται και νέες στρατηγικές όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ή η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο. Ευχαριστώ πολύ. Η ε, κυρία Χάζεκαμπ από την ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε πίτροπε. Η πολιτική, η γεωργική, οι επιδοτήσεις, η σφαγή σε μεγάλη κλίμακα των ζώων, ε, έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε μια διατροφή που δεν είναι υγιεινή και είναι και σε μεγάλη βιομηχανική κλίμακα. Ε, καταστρέφουμε το περιβάλλον. Οι μικρής κλίμακας σε γεωργία αντιμετωπίζουν προβλήματα. Εκατομμύρια ζώα σφάζονται. Και αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο. Και βέβαια χάνεται η βιοπικιλότητα. Είναι ένα στραβό σύστημα οι αγρότες πρέπει να έχουν ε, καλή τιμή για τα ζώα τους, να είμαστε τίμοι για τα ζώα, για τους αγρότες, για το περιβάλλον, για όλους. Ενώ έχουμε συμφωνίες όπως είναι TTIP, η συμφωνία με τη Μερκοσούρ. Ανοίγουμε τα σύνορά μας για φτηνά προϊόντα και προϊόντα τα οποία δεν προστατεύουν ούτε το περιβάλλον ούτε τα ζώα. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει να καταργηθούν οι ενισχύσεις στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Τζαρούσο από τους μη εγγεγραμμένους. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, Μεγάλε είναι οι απαιτήσει που έχουμε από τη στρατηγική, από το αγρόκτημα στο πιάτο. Να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα. Μείωση των λιπασμάτων, μείωση των φυτοφαρμάκων. Αν αυτό κρίνεται αναγκαίο, αυτό θα πρέπει να γίνει και επίσης υπάρχει και μια υποχρέωση για να, μειωθούν, να μειωθεί η σπατάλη των τροφίμων. Και αυτό προβλέπεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Λέτε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ετικετοθεσία όσον αφορά τη βιωσιμότητα των προϊόντων αυτών που να δίνει πραγματικά τη θρεπτική αξία των τροφίμων αλλά επίσης και το οικολογικό τους αποτύπωμα και να λαμβάνει υπόψη και την προστιθέμενη αξία των γεωργών. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίξουμε περισσότερο ότι η βιολογική παραγωγή πραγματικά θέτει το γεωργό στο κέντρο της παραγωγικής διαδικασίας εργασία. Μόνο μέσω των βιολογικών προϊόντων και τη καλλιέργεια αυτή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τι κλιματικέ αλλαγέ. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν πραγματικά να ενταχθούν οι στρατηγικοί από το αγρόκτημα στο πιάτο γεωργή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει απαραίτητη χρηματοδότηση τη κοινή γεωργική πολιτική και απαραίτητη ορθή διαχείριση. Α μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντο. Σα ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε λοιπόν. κυρία Μακίνες, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η σημερινή συζήτηση ελπίζω να ξυπνήσει την Επιτροπή και το Σώμα και να τους θυμίσει ότι είναι ενοχλημένοι, θυμωμένοι και νιώθουν να, τους, να δέχονται επίθεση οι αγρότες μας. Το θέμα αυτό και η στρατηγική μας για από το χωράφι στο πιάτο είναι κάτι που πρέπει να λάβει υπόψη τους αγρότες και αυτό το μήνυμα ελπίζω να το μεταφέρετε στους συνομιλητές σας. Η στρατηγική αυτή έχει να κάνει και με την ανταγωνιστικότητα, έχει να κάνει με το θεμητό εμπόριο, τη δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Γεωργία. Πρέπει να πω ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείτε και εσείς και άλλοι στο σώμα ε, βέβαια είναι φορτισμένη ε, μιλάμε για εντατική, για... πρέπει να προσέχουμε τη γλώσσα, γιατί ε, πολλοί από εμά ξέρουμε ότι υπάρχουν όχι μόνο μικροί αγρότες, υπάρχουν και μεσαίοι, υπάρχουν και μεγάλοι. Δεν πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι κάποιοι είναι καλύτεροι από κάποιους άλλους. Πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην έρευνα, στην καινοτομία, στην καλύτερη τεχνολογία οι αγρότες για να μπορούν να προσφέρουν αυτά που τους ζητάμε. Και μην ξεχνάμε ότι οι αγρότες ήδη το κάνουν πριν από εμά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 θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης και το σεβασμό, το σεβασμό των γεωργών, των αγροτών μας και γενικά των αγροτικών κοινοτήτων. Στην πράξη όμως πώς μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Η απάντηση στις νέες προκλήσεις δεν μπορεί να έρθει χωρίς τις ίδιες τις προσπάθειες των γεωργών. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι εμείς πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Εμείς πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη και δικαιοσύνη απέναντί τους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια βιωσιμότητα της δικής μας γεωργίας που να είναι αξιοπρεπής όμως για τους ίδιους τους γεωργούς οι οποίοι ουσιαστικά ε, συμβάλλουν στην ίδια τη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών. Κύριε Επίτροπε, εσείς πώς θα διαμορφώσετε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική προκειμένου να έχουμε μια βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών. Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό στο πλαίσιο της στρατηγικής από το αγρόκτημα στο πιάτο. Η στρατηγική αυτή Πώ θα μπορούσε στην πράξη να εφαρμοστεί λαμβάνοντα υπόψη τι πραγματικέ ανάγκε του αγροτικού κόσμου. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Μίλλερ, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αυτή τη στιγμή τι ζούμε. Γίνεται πολιτική και πάλι στους δρόμους. Διαδηλώνει ο κόσμος για περισσότερη προστασία του κλίματος και της φύσης. Καλό είναι και μπράβο τους και τους χειροκροτούμε. Όταν όμως διαδηλώνουν χιλιάδες αγρότες που ε, στενάζουν από τη γραφειοκρατία και από την αγωνία για την επιβίωση, τους αγνοούν οι Βρυξέλλες. Και όλη η κατάσταση αυτή υποδαβλίζεται από τον αντιπρόεδρό μας, τον κύριο Τίμερμανς, που έρχεται και κάνει δηλώσεις για δραστική μείωση της κτηνοτροφίας. Αυτό το 40% λιβάδια που έχουμε στην Ευρώπη, τι θα το κάνουμε, πώς θα το αξιοποιούμε και ποιος θα το φροντίζει. Φυσικά γνωρίζουμε ότι όλοι πρέπει να γίνουμε πιο αηφόροι, πιο βιώσιμοι, να κάνουμε περισσότερα για τη γεωργία, η οποία αλλάζει. Αλλά αυτό θα το πετύχουμε μόνο από κοινού. Γι' αυτό η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε ακόμα περισσότερα βάρη για τους αγρότες και θα πρέπει να έχουν μια ασφάλεια προγραμματισμού. Σας καλώ να μην ε, ε, κάνετε καθυστερήσεις τώρα από την Πράσινη Συμφωνία και τούτη εδώ στρατηγική ε, στην κοινή γεωργική πολιτική. Έτσι κι από το 2023 αρχίζει. Υπάρχει το νομοθετικό οικολογικό πακέτο και μπορούμε ε, να βάλουμε ε, οικολογικά σχήματα και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Δεν θέλω να ε, γίνει πραγματικότητα μια παροιμία που λέει καταστρέφουμε τους αγρότες και εισάγουμε αυτά που τρως και τα βρίσκεις σε σούπερ μάρκετ. Ο συνάδελφος Λεμπρετών, παρακαλώ. Merci, Madame la Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή Φοντερ Λάιεν μίλησε για την πρόθεσή της να έχει ένα μοντέλο γεωργίας και παραγωγής βιώσιμο, σεβόμενη τις επιθυμίες των καταναλωτών, με σλόγγαν όπως αυτό από το αγρόκτημα στο πιάτο, Farm to Fork. Σήμερα ε, μου ζητάτε να σα πω τη γνώμη μου. Το πρόβλημα είναι ότι προ το παρόν δεν έχουμε κανένα συγκεκριμένο έγγραφο για το σχέδιο αυτό. Επιπλέον έχουμε μια μισή σελίδα παρουσίαση στο έγγραφο προ ανατολισμού μόνο. Έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, η στρατηγική αυτή από το χωράφι στο πιάτο είναι κενή περιεχομένου. Και για να είμαι επικοδομητικό, επισύνω την προσοχή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εναρμόσει τι μελλοντικέ προτάσει με την νέα κοινή γεωργική πολιτική η οποία ολοκληρώνεται. Όσον αφορά το περιεχόμενο, δεν φτάνει να μιλάμε για όριστα μέτρα, όπως για παράδειγμα τη σημαντική μείωση της χρήσης των παρασιτοκτόνων. Πρέπει επίσης να βρούμε πραγματικές λύσεις στα πραγματικά προβλήματα. Πρώτον, να διασφαλίσουμε την κυριαρχία μας στη διατροφή μας, αντί να θυσιάζουμε την γεωργία μας στις ελεύθερες συναλλαγές και την παγκοσμιοποίηση. Δεύτερον, να καταργήσουμε τα λιγοπόλια Τη μεγάλη παραγωγή. Τρίτον, να διευκολύνουμε το επάγγελμα του αγρότη, απλοποιώντας τους κανόνες και τις διοικητικές διαδικασίες που είναι τρομερές πια. Πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε με σλόγγαν και να περάσουμε στις δράσεις, γιατί οι αγρότες και οι καταναλωτές μας περιμένουν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χόισλενγκ, παρακαλώ. Ναι, κύριε Επίτροπε, είπατε κάτι σημαντικό στην αρχή της ομιλίας σας. Δεν θα πρέπει η Γεωργία να βαίνει βιομηχανικός κλάδος. Συμφωνώ, απολύτως. Αλλά χρειάζεται διαφορετική γεωργική πολιτική, γιατί τώρα εποφελούνται οι μεγάλοι από τις πληρωμές. Αν συνεχίσουμε να μοιράζουμε τις πληρωμές 70% ε, με βάση τη στρεματική ενίσχυση χωρί όρου. αυτό δεν είναι πολιτική για το περιβάλλον. Και αν τα λέτε σοβαρά όλα αυτά με τι στρατηγικέ και τι πράσινε συμφωνίε και τα αγροκτήματα και τα πιάτα, στο τέλος τι θα κάνετε στην κυνηγεωργική πολιτική. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε συντηρητική πλειοψηφία που θέλει να παραμείνουν τα πράγματα όσο έχουν. Καλά, να πρασινίσουν λιγάκι γύρω-γύρω. Ε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για τους αγρότες, ναι, αλλά έχουμε και ένα μαζικό πρόβλημα με την ε, απώλεια της βιοπικιλότητας. Τι, αυτό να μην το συζητάμε. Και το ελεγκτικό συνέδριο είπε ότι κάνουμε καταστροφική πολιτική στα φυτοφάρμακα. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από τα λοιπάσματα αυτά τα βλαβερά. Θα εξαφανίζονται τα είδη και θα, θα μπορέσουμε αυτό να το αντιστρέψουμε. Φυσικά έχετε δίκιο όταν λέτε ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τις συνέπειες που έχει η γεωργική μας πολιτική σε τρίτες χώρες. Αυτή η συμφωνία με το Μερκοσούρ θα την εγκρίνουμε και ε, μαζικά θα εισάγουμε σόγια ε, κοιτάξτε και την εμπορική πολιτική και αυτή πρέπει να αλλάξει. Και θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε διαφορετική πολιτική για την προστασία των ζώων. Δεν γίνεται με η εντατική κτηνοτροφία. Ε, χρειάζεται πηγόντως διορθώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Ο κύριος ε, Ράισεν. Οι προκλήσεις για τη γεωργία φαίνονται τεράστιες ε, ε, τρόφιμα υψηλής ποιότητας, πρέπει να φροντίζουν το τοπίο και τη βιοποικιλότητα και όσο γίνεται να είναι λιγότερες οι εκπομπές. Αυτό τι ζητάει σύγχρονη γεωργία που να χρησιμοποιεί ε, τις νέες τεχνολογίες. Θα πρέπει να τις ακολουθήσουμε, θα πρέπει να τις προωθήσουμε και να επενδύσουμε σε αυτές. Το μεγαλύτερο λάθος της νέας στρατηγικής είναι να αρχίσει πάλι να ρυθμίζει και να απαγορεύσουμε τα φυτοφάρμακα όταν δεν υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να φέρει καλά σχέδια για να επιβραβεύει τον κλάδο για τις προσπάθειές τους και να μην τους αφαιρούν τα μέσα που έχουν για να αγωνίζονται ε, έτσι ώστε να ε, έχουν μια υγιή διαχείριση της εκμετάλλευσής τους. Κύριε Επίτροπε, μην κρίνετε τις επιχειρήσεις με βάση τον αριθμό των ζώων ανακτηνοτροφία, αλλά τι κάνουν για το περιβάλλον αναμονάδα μεγάλου βοηδούς. Εκεί θα πρέπει να κριθούν και εκεί θα πρέπει να αποφασίσετε. Έχετε μπλε κάρτα, κύριε Ράισεν. Τι δέχεστε. Ναι. Ο συνάδελφος Μάντερς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω το συναφορά Ράισεν, μήπως έχει σκεφτεί ε, τίποτα για τη σπατάλη των τροφίμων που ε, επιβαρύνει πάρα πολύ τον ευρωπαϊκό ε, προϋπολογισμό. Αν κάνουμε και οικονομία από όλα αυτά τα τρόφιμα που πετάμε, δεν χρειάζεται καν να δίνουμε επιδοτήσεις. Ε, απάντηση. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και θα πρέπει να το κοιτάξουμε, να το αντιμετωπίσουμε. Πάρα πολύ σημαντικό, δεν λέω. Φυσικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει Διαφωνώ ότι δεν χρειάζονται επιδοτήσεις. Προς το παρόν χρειάζονται για να βοηθήσουμε τον κλάδο να κάνει αυτή την αλλαγή και να προχωρήσει αυτή τη μετάβαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φλάναγκαν. Η στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο, εφόσον ετοιμαστεί σωστά θα βοηθήσει και τους αγρότες και τους καταναλωτές. Εμείς ε, βλέπουμε να βάζουμε στο κρέας ε, βοηδές ε, αλλά χωρίς ε, Πολλέ λεπτομέρειε. Εμεί από την άλλη μεριά θέλουμε να υπάρχουν όλε οι λεπτομέρειε για το πώ τι παραστοκτόνα χρησιμοποιήθηκαν κλπ. Για να ξέρουμε και να διαφοροποιούμε ένα είδο βόρειο κρέατο από ένα άλλο. Πηγαίνει ο κόσμο και αγοράζει και πληρώνει περισσότερα για ορισμένα προϊόντα, το ίδιο μπορεί να συμβεί και με το βόλιο κρέα. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνει, πόσα χρήματα θα βάλει. Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Και το λέει η Επιτροπή. Εγώ λέω ότι ναι, πρόκειται φυσικά και για την ασφάλεια και για την προστασία μας. Κοιτάξτε τις προτεραιότητές σας. Εμείς βλέπουμε 22 φορές παραπάνω χρηματοδότηση για τα όπλα, ε, για τις σφαίρες από ό,τι για τη Γεωργία. Εμείς ε, έχουμε βάλει πρώτα τον πόλεμο και μετά τη διατροφή. Αυτό πρέπει να το αντιστρέψουμε και να είμαστε σοβαροί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Μπούντα, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο είναι θεμελιώδου σημασία προκειμένου να πετύχουμε πολλού και διάφορου στόχου. Ποιότητα τρόφιμα, ποιότητα τροφίμων, μια καλή διαβίωση και καλό εισόδημα για του γεωργού, αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Βέβαια, ο γεωργικό τομέα δεν είναι ο μόνο ο οποίο ευθύνεται για τη μείωση τη βιοπικιλότητα, για το ότι χάνονται κάποια είδη. Όλοι φέρουμε αυτή την ευθύνη. Οι γεωργοί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως μέρος της λύσης και όχι ως μέρος του προβλήματος, όσον αφορά για παράδειγμα το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Τώρα η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο θα στεφθεί με επιτυχία μόνο αν πραγματικά παραμείνει ρεαλιστική και αν μέσω της στρατηγικής αυτής καταφέρουμε τελικά να καταλάβουμε και τα δύναμα σημεία, αλλά και τις μεγάλες ευκαιρίες που μας δίνει ο γεωργικός τομέας. Στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δεν δίνουμε τις απαραίτητες ευκαιρίες στους γεωργούς να προσαρμοστούν. Αυτή τη στιγμή πολύ φοβάμαι ότι και οι γεωργοί αλλά και οι καταναλωτές θα πρέπει να καταβάλουν υψηλότερο τύπημα. Και τελικά οι δύο αυτοί οι δύο αυτές πλευρές θα βρεθούν χαμένες και πολύ φοβάμαι ότι ενδεχομένω να δούμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα κίνημα κίτρινων γυλαίκων. Η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο πραγματικά θα πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για το γεωργικό τομέα. Μόνο τότε θα στεφθεί με επιτυχία. Χρειαζόμαστε καλύτερη χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα με λιγότερα χρήματα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε πρόσβαση στην γεωργία ακριβία καθώ επίση και στι νέε τεχνολογίε καθώ επίση και στα νέα επιστημονικά δεδομένα. Σα ευχαριστώ. Ο συνάδελφο Αντριέ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από το ακρόκτημα στο πιάτο θα πρέπει να σκεφτόμαστε με μικρές αποστάσεις, ανθρώπινες εκμεταλλεύσεις, οικογενειακές. Σημαίνει ότι θα έρθει πιο κοντά ο καταναλωτής στον παραγωγό. Αυτή η επιλογή σημαίνει επαναπροσανατολισμό του γεωργικού μοντέλου, όπου θα πρέπει να ζουν αξιοπρεπώς οι αγρότες από το επαγγελμά τους και οι καταναλωτές να έχουν ποιοτικά προϊόντα. Αυτή η στρατηγική επίσης σημαίνει μέτρα για να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων, που είναι 25 με 30% της παραγωγής τροφίμων. Επίσης, μείωση των χημικών χημικών φυτοφαρμάκων για να έρθουν τα βιολογικά προϊόντα πιο εύκολα στην αγορά. Βεβαίω, ναι, η Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να αποτελέσει πραγματική ευκαιρία για του αγρότε και την Ήπεθρο. Και επίση θα πρέπει να έχει και κομβικό ρόλο στο νέο οικονομικό μοντέλο που μα παρουσιάζεται με αλφαγιώτα και είναι αναπότρεπτο. Γι' αυτό το λόγο η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει πρώτα απ' όλα να πλαισιώνει και να συνοδεύει τους αγρότες σε αυτή τη μετάβαση. Το κρίσιμο είναι ε, να ξεπεράσουμε τις εξαγγελίες τώρα και να περάσουμε σε πρακτική υποστήριξη όλων αυτών. Ευχαριστώ, ο κύριος ε, Χάιτεμα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη Επίτροπε. Επί δεκαετίες είχαμε μια κοινή γεωργική πολιτική που δεν λειτουργεί καλά αυτή τη στιγμή και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο το επικρίνει πολύ. Για ποιο λόγο. Έχουμε μέσα μέτρα πρασινίσματος που αποφασίζονται στις Βρυξέλλες και οι αγρότες πρέπει να τα εφαρμόσουν. Έχει δοκιμάσει κανείς πώς γίνεται και τι αποτέλεσμα δίνει αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ελέγξει τα αποτελέσματα και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους αγρότες ε, όταν καινοτομούν, όταν επιχειρούν για να έχουν κίνητρα και να ε, ενισχύσουμε αυτή την επιχειρηματικότητα και να έρθει το πρασίνισμα. Και θα πρέπει αντίστοιχα να επιβραβεύονται οι αγρότες. Κοιτάξτε σε όλη την Ευρώπη τι, γίνεται το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Ε, τι φοβάμαι τώρα. Με αυτή τη στρατηγική θα επιστρέψουμε στην παλιά πολιτική. Μόνο μέτρα από τις Βρυξέλλες από πάνω προς τα κάτω που θα τα επιβάλλουμε και δεν θα μπορεί να ορθοποδήσει πια ο αγρότης. Οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας για την κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να εστιάζουν στο αποτέλεσμα και να επιβραβεύουν το αποτέλεσμα και να κοιτάξουμε στη νέα στρατηγική. Ας πούμε, δεν μπορούμε ακόμα να χρησιμοποιήσουμε αλεύρι από έντομα στην κτηνοτροφία. Μα είναι γελία αυτά τα πράγματα. Ε, ας πούμε, ε, ακόμα προωθούμε τα τεχνητά λιπάσματα ενώ έχουμε πήξει στο άζωτο και δεν χρησιμοποιούμε την κοπριά. Ευχαριστώ πολύ και συνεχίζουμε με τη συζήτησή μας. Ο συνάδελφος Νταρέ παρακαλώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρουσίασε τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο που υποτίθεται ότι θα κάνει τον γεωργικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μοντέλο αναφοράς βιωσιμότητος. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε και ασφάλεια στα γεωργικά τρόφιμα για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε και για τους γεωργούς το κατάλληλο εισόδημα, καθώς επίσης και μια πολιτική η οποία θα μειώνει τα φυτοφάρμακα και θα προωθεί την βιοπικιλότητα. Πραγματικά όμως εδώ πέρα θα επιβάλλει νέους κανόνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους γεωργούς και τι προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου πραγματικά να καταφέρουμε να προστατευθούμε από γεωργικά προϊόντα τα οποία δεν τηρούν τα δικά μας τα πρότυπα και έρχονται από χώρες όπως η Καμπότζη για παράδειγμα ή το Βιετνάμ. Νομίζω ότι μόνο αν λάβουμε αυτά τα περιοριστικά μέτρα, τα προστατευτικά μέτρα, θα καταφέρουμε να προφυλάξουμε τους γεωργούς και τους πολίτες μας. Ευχαριστώ κύριος Μπιτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Επίτροπε. Η πρόταση μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ που συζητάει σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει ενό γράφου που ετοίμασε η προηγούμενη θητεία και που δεν συνάδει με τι προσδοκίε τη νέα αυτή θητεία, που ήδη έχει ψηφίσει για το κατεπήγον του κλίματο. Και όντω επήγει το κλίμα. Η πρόταση για τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ δεν είναι στο ύψο των όσων διακυδεύονται και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κύριε Επίτροπε. Συνεπώ, η στρατηγική αυτή από το χωράφι στο πιάτο είναι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διορθώσει τα, τα λάθη και τι αδυναμίε. Κι όμω πρέπει να αποτελέσει μοχλό για να συνοδεύσει, να χρηματοδοτήσει την οικολογική μετάβαση για του Ευρωπαίου αγρότε. Συνεπώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ θα τα αντιστοιχεί σε αυτά. Τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ δηλαδή με νέου στόχου που εισάγει η νέα πράσινη συμφωνία. Πώ είναι δυνατόν μία από τι πιο σημαντικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίζεται πριν από τη στρατηγική. Και πώ είναι δυνατόν να πετύχουμε του στόχου τη πράσινη συμφωνία, χωρί να κινητοποιήσουμε την ΚΑΠ, η οποία σήμερα δεν περιλαμβάνει κανένα κοινό και σαφή στόχο για μείωση των παρασιτοκτόνων, για ε, προστασία της βιοπικιλότητας, για μείωση των αερίων του θερμικού ποίου και χωρίς να πληγεί η διατροφική μας κυριαρχία. Είναι δικιά μας ευθύνη, είναι ιστορική σημασίας, προκειμένου να μην χάσουμε την ευκαιρία αυτή, να αλλάξουμε σε βάθος τα συστήματα με τα οποία διατρεφόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Α, συγγνώμη, πριν την κυρία Τόμασιτς, έχετε μπλε κάρτα, τη δέχεστε, κύριε Μπιτόμου. La carte bleue, vous... Δέχεστε την μπλε κάρτα, ναι. 30 δευτερόλεπτα έχετε για την ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί, αγαπητές συνάδελφε. Δεν... Ε, λέτε ότι δεν συμφωνείτε με τη στρατηγική από το χωράφι στο πιάτο. Λέτε ότι δεν συμφωνείτε η ΚΑΠ να μπορεί να προχωρήσει. Και λέτε ότι δεν συμφωνείτε με το ότι πρέπει να συνεχίσουμε να παράγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τρόφιμα. Εσείς, συγγνώμη, πώς βλέπετε την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο με εισαγωγή προϊόντων. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε διατροφική ασφάλεια και ασφάλεια τροφίμων αν εισάγουμε μόνο από άλλες τρίτες χώρες. Πώς θα διασφαλίσουμε ε, την ε, επιβίωση των αγροτών και των ανθρώπων στην ε, Ήπεθρο αν δεν πάρουμε τέτοια μέτρα. Απάντηση. Εγώ δεν είπα ότι δεν συμφωνώ. Ζήτησα να υπάρχει συνοχή ανάμεσα στη στρατηγική από το χράφι στο πιάτο με την κοινή γεωργική πολιτική. Δεν είναι ακριβώς ότι αντιτίθεμε. Λέω ότι σήμερα με εκπλήσει που προχωράμε με μια στρατηγική χωρίς να έχουμε καταλήξει για την κοινή γεωργική πολιτική ε, να επηρεάζει η στρατηγική την ΚΑΠ. Όσον αφορά τις εναλλακτικέ και τη δυνατότητα να πετύχουμε την διατροφική κυριαρχία, πρέπει να συγκλίνουν η υποχρέωσή μας για την προστασία της βιοπικιλότητας, για την προστασία του κλίματος, δεν είναι δυνατόν συγχρόνως να παράγουμε όλο και περισσότερο, δεν είναι δυνατόν να αυξάνονται τα παρασυτοκτόνα. Ευχαριστώ. Προχωρούμε. Η κυρία Τόμαση, τη παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η κοινή γεωργική πολιτική είναι η πιο ακριβή και λιγότερο αποδοτική ευρωπαϊκή πολιτική. Έχουν γίνει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν έχουν οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα έχουμε μια πολύ υψηλή παρέμβαση κρατική με αποτέλεσμα η κοινή γεωργική πολιτική να είναι μη αποδοτική, μη ανταγωνιστική και ιδιαίτερα ακριβή και δαπανηρή. Ανοίγεται μια νέα δημοσιονομική περίοδο μπροστά μα και πρέπει να καλύψουμε και άλλε πολιτικέ, όπω την κυκλική οικονομία και μια γενικότερη πολιτική βιωσιμότητα. Πολύ φοβάμαι όμως ότι δυστυχώς, θα καταλήξουμε σε μη αποτελεσματικά μοντέλα, σαν αυτά τα οποία γνωρίζουμε από το παρελθόν. Νέα ακριβά προγράμματα, νέες υψηλέ επιδοτήσεις, μακροπρόθεσμα δεν μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμη λύση. Χρειαζόμαστε καινοτομία στη γεωργία και θα πρέπει να υπάρχουν προγράμματα κατάρτισης ανοιχτά προς όλους τους γεωργούς. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε πραγματική βιωσιμότητα και πραγματικό ανταγωνισμό στο τομέα αυτό και μόνο έτσι μπορούν να μειωθούν και επιδοτήσεις. Ευχαριστώ κυρία Μόντικ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Στην Φιλανδία συνηθίζουμε να λέμε ότι η αρχή κάθε σοφίας είναι η αναγνώριση των γεγονότων. Αν αναγνωρίσουμε τα γεγονότα, αναγνωρίζουμε ότι τα μέτρα δεν είναι επαρκή μέχρι τώρα. Αλλιώς θα καταλήξουμε να αποθηκεύουμε άνθρακα στους αγρούς μας, αντί να παράγουμε τρόφιμα. Τα φυτοφάρμακα, τα παριστοκτόνα καταστρέφουν και τον κόσμο και τη φύση. Πρέπει να απαλλαγούμε από αυτά. Δεν μπορούμε βέβαια να τιμωρούμε τους αγρότες, γιατί οι αγρότες είναι ειδικοί στη δουλειά τους. Η κοινή γεωργική πολιτική όμως και οι ενισχύσεις πρέπει να βοηθούν τους αγρότες να πετύχουν μια μετάβαση προς μια περισσότερο οικολογική παραγωγή. οι καταναλωτές θέλουν να πληρώσουν παραπάνω για τρόφιμα τα οποία είναι περισσότερο υγιεινά και παράγονται με ηθικό τρόπο. Και είναι καλό στη σήμανση των τροφίμων να αναφέρονται αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο συνάδελφος Θοίδο Άλβαρεθ, παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, ξεκινάμε από τη βάση ότι περισσότεροι εδώ μέσα θέλουμε μια γεωργία περισσότερο βιώσιμη, η οποία να συνεισφέρει να πετύχουμε τους στόχους μας για το 2030. Η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο, ελπίζουμε ότι συνεισφέρει σε αυτό. Πολλοί λένε ότι η γεωργία μας θέλει να γίνει κάτι που τα καταπίνει όλα. Η... Με τη γεωργία σαν θέλουμε να κάνουμε τη γεωργία όπω είναι το iPhone, που να μπορεί να τα κάνει όλα. Προσοχή όμως, δεν είναι δυνατόν να έχουμε κάτι το οποίο να εξυπηρετεί όλους τους σκοπούς. Δεν μα ενδιαφέρει. Κάποιοι θέλουν η Ευρωπαϊκή Γεωργία να χρησιμεύει για να προστατεύει το περιβάλλον, για να αντιμετωπιστεί κλιματική αλλαγή, για να μειωθούν οι διαφορές για να μειώσουμε τη χρήση των αντιβιωτικών των φυτοφαρμάκων, για να προστατεύσουμε τη βιοπικιλότητα, για να ενημερώνεται καλύτερο ο πολίτης, για να βελτιωθεί η προστασία των ζώων κλπ. κλπ. Μην ξεχνάμε όμω ότι ο πρώτο στόχο τη γεωργία μα και τη κοινή γεωργική πολιτική μα είναι να έχουμε προϊόντα ποιότητα σε προσιτέ τιμέ που να βοηθούν τους αγρότες και να τους ανταμείβουν για τις προσπάθειές τους. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το πώς θα προχωρήσει αυτή η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους να ε, συνεχίσουν να πετυχαίνουν τους στόχους μας και να ανταμείβονται για τις προσπάθειές τους. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νόιχελ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Υποτίθεται ότι σήμερα συζητούμε ακριβώς για τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο. Και βλέπω ήδη ότι έχετε νευράκια. Γιατί ουσιαστικά συζητάμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Και στους διαδρόμους αυτό συζητάνε όλοι. Η παλιά πρόταση για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ε, ε, μπορεί να σταθεί με την Πράσινη Συμφωνία. Γι' αυτό σας έχει πιάσει εκνευρισμός. Αυτοί που υποτίθεται ότι είναι εδώ εκπρόσωποι όλων των αγροτών. Γιατί αναγνωρίζουν και οφείλουν να αναγνωρίσουν ότι η παλιά πρόταση δεν είναι συμβατή με τη νέα πράσινη συμφωνία. Και το νιώθω αυτό τον εκνευρισμό. Μπορώ να σας πω ότι το καταλαβαίνω κιόλα. Αλλά μην νομίζετε ότι εσεί εκπροσωπείτε όλους τους αγρότες. Ένα τμήμα τους μόνο. Υπάρχουν πολλοί αγρότες που θέλουν να πάρουν ένα καινούριο δρόμο και εγώ είμαι εδώ για να υποστηρίξω αυτού ακριβώς τους αγρότες. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Ο συνάδελφος Χλαβάτσεκ, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, να αποθέτουμε πάρα πολλές ελπίδες σε εσά. Η παραγωγή τροφίμων, οι γεωργοί, κατηγορούνται εντελώς άδικα. Και νομίζω ότι πάρα πολλοί πολίτες ε, ξεχνάνε ότι οι δικοί μας οι γεωργοί παράγουν τελικά τα πιο ασφαλή τρόφιμα στον κόσμο ή από τα πιο ασφαλή τρόφιμα στον κόσμο σε οικονομικά προσιτές τιμές. Η γεωργία επίσης είναι ένας ιδιαίτερα ρυθμισμένος τομέας. Απελευθερώνουμε το εμπόριο, δημιουργούμε νέους κανονισμούς, προβλέπουμε επιδοτήσεις και ενισχύσεις και από την άλλη η γεωργία είναι αυτή οι οποίοι αισθάνονται έντονα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Και ακριβώς για αυτό το λόγο η γεωργία θα πρέπει να αποτελέσει λύση οποιασδήποτε αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Δυστυχώς η στρατηγική από το γρόκτημα στο πιάτο επί του παρόντος δεν περιλαμβάνει στο κέντρο της τους γεωργούς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυξάνει κάποιες τιμές στα τρόφιμα και υπεριθμίζει τον τομέα αυτό. Έχουμε φτάσει πραγματικά τα όρια μας. Θα έπρεπε να έχουμε μια πραγματική στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο υπέρ των γεωργών. Για ποιο λόγο εσείς αυτή τη στιγμή στρέφεστε κατά των γεωργών και όχι κατά, για παράδειγμα, το σούπερ μάρκετ ή του αθέμητου ανταγωνισμού. Η κυρία Σαροντών έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι ακολουθώντας ενδεχομένως τις νουθεσίες της Γκρέτας έχετε επινοήσει και ένα νέο πρόγραμμα από το αγρόκτημα στο πιάτο. Μία στρατηγική που έχει ως βασικό πυλώνα να γίνουν οι γεωργοί και οι αλείς θεματοφύλακες της κλιματικής αλλαγής. Νομίζω ότι εδώ πέρα δημιουργείται ένα μεγάλο πράσινο αδελφό. Μας αναφέρατε διάφορες βασικές αρχές, όπως για παράδειγμα το να έχουμε τρόφιμα σε, χαμηλή, σε χαμηλές τιμές. Με αυτό θα στραφεί κατά της ίδιας της ποιότητας των τροφίμων. Κατά αυτόν τον τρόπο προωθείτε τα βιομηχανοποιημένα τρόφιμα. Και λέτε επίσης ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε υποκατάστατα τροφίμων τα οποία τα προκύπτουν από τα φύκια μαζί το, η ποιότητα των τροφίμων λέτε επίση ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια νέα ετικετοθεσία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην δημιουργήσετε εδώ πέρα ένα νέο σύστημα διακριτικής μεταχείρισης. Νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει αυτή τη στιγμή να ασχοληθούμε περισσότερο με την ασφάλεια των τροφίμων και όχι να προωθούμε όπω το κάνετε τις μεγάλε πολυεθνικές. Ευχαριστώ, συνάδελφο Ροπέ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το σημερινό σύστημα έχει πολλές αδυναμίες και καταστρέφει τους αγρότες σε μερικές περιοχές και παραγωγή σε άλλες περιοχές. Ε, το γαλακτοκομικό τομέα, για παράδειγμα. Οι λιανικές αλυσίδες επίσης ε, απειλούνται και οι καταναλωτές. Οι περισσότερες ε, αλυσίδες σούπερ μάρκετ πολλούσαν πράγματα που δεν θα πρέπει να τα κρύβουν από τους καταναλωτές. Σήμερα η παραγωγή τροφίμων φτάνει στα πιάτα μας αφού προηγουμένως έχει ταξιδέψει χιλιόμετρα και χιλιόμετρα. Χρειάζεται κάτι τέτοιο. Βοηθάει αυτό καθόλου το περιβάλλον, το κλίμα. Η στήριξη των αγροτών σε διάφορες χώρες έχει μειωθεί ξανά και ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά έχουμε καταλήξει να έχουμε πρώτης κατηγορίας και δεύτερης κατηγορίας αγρότες, οι οποίοι επιπλέον αντιμετωπίζουν πολλούς ε, φραγμούς όσον αφορά την ελευθερία ε, διακίνησης των προϊόντων τους. Άσε που εισάγουμε προϊόντα χαμηλής ποιότητας, αφιβόλου ποιότητας, γενετικά τροποποιημένα κλπ. Οι αγρότες θα πρέπει να μπορούν να δουλέψουν στη γη τους για να εξυπηρετούν τον κόσμο και να μπορούν και εκείνοι να ζουν αξιοπρεπώς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Αγγιλάρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ο αγροτικός τομέας στην Ισπανία κινητοποιείται τον τελευταίο καιρό γιατί αντιμετωπίζει κρίση. Πρόκειται για ε, προϊόντα τα οποία τελικά δεν ε, καλύπτουν το κόστος παραγωγής του όταν πολλούνται. Πρόκειται για εμπορικέ συμφωνίες οι οποίες αντιβαίνουν στις αρχές μας δεν υπάρχει αποδοτικότητα και έχουν αναγκαστεί πολλέ ε, καλλιέργειε να κλείσουν ξανά και ξανά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει τώρα ότι έχει αυτή τη νέα στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο. Όμως τίποτα δεν λέμε για τις ανησυχίε, τι πραγματικέ των αγροτών. Γιατί επικεντρωνόμαστε μόνο στην μείωση των φυτοφαρμάκων, στην αύξηση τη προστασία των ζώων, στι νέε υποχρεώσει υπέρ του περιβάλλοντος Πώ θα ανταποκριθούμε στην κρίση τη αγορά που αντιμετωπίζει ο τομέα στην Ισπανία αλλά και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. αν συνεχίζουμε να μην καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για έναν οικονομικό τομέα, ο οποίο αν δεν είναι αποδοτικό, δεν θα είναι και βιώσιμο. Συνεπώ, θα συνεχίσουμε έτσι να είμαστε μακριά από την πραγματικότητα στους αγρού μα και δεν θα προσφέρουμε λύσει σε έναν κλάδο που χρειάζεται περισσότερη κατανόηση και επιγόντω στήριξη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κόκαλης, παρακαλώ. Ως μέλος της ε, Επιτροπής ε, συμφωνώ με τη στρατηγική αυτή ο Ιπποκράτης είπε ότι θα πρέπει ε, τα φαγητά να είναι το φάρμακό σας και το φάρμακό σας να είναι τα τρόφιμα. Συνεπώς χρειαζόμαστε μια νέα κοινή γεωργική πολιτική που να ε, συνάδει με την στρατηγική μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η ΚΑΠ δεν πρέπει να αφήσει κανέναν ξεχασμένο. Πρέπει να βοηθήσει τη δίκαια μετάβαση. Ο κόσμος χρειάζεται σε προσιτές, σε τιμές, καλής ποιότητας ε, τρόφιμα και με βιώσιμο τρόπο παραγωγή. Οι αγρότες για να τα καταφέρουν χρειάζονται ε, θέσεις απασχόλησης ε, ποιότητας, ενίσχυση. Πλέον πρέπει η ΚΑΠ να συνάδει με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να έχουμε μια βιώσιμη ΚΑΠ με το σωστό προπολογισμό που θα στηρίζει τους αγρότες για να πετύχουν την βιοπικιλότητα, την προστασία του περιβάλλοντος ε, και τους στόχους της Ένωσης γενικότερα. Και ο Ιπποκράτης στήριζε ε, τέτοιες αρχές. Ας τον ακούσουμε λοιπόν και ας προχωρήσουμε στην Νέα Ευχαριστώ. Αμάρο Άλβαρο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Κύριε Επίτροπε, πριν από λίγο αναφερθήκατε σε κάποιες πολύ σημαντικές ανησυχίες, ε, τις οποίες ε, συμμεριζόμαστε πολύ και στη δική μου την πολιτική ομάδα συμφωνούμε μαζί σας. Προφανώς θα πρέπει να αποφύγουμε την απερίμωση των αγροτικών περιοχών, θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη διατροφική ασφάλεια και γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειάζεται πιο υψηλός προπολογισμό για την κοινή γεωργική πολιτική. Αλλά κύριε Πρόεδρε, ενώ συζητάμε αυτή τη στιγμή την περίφημη αυτή στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο, υπάρχει κάτι το οποίο με έχει προβληματίσει πάρα πολύ από την αρχή της συζήτησης, γιατί θεωρώ ότι είναι εντελώς άδικο για τους γεωργούς αυτή τη στιγμή, από τη μία στιγμή στην άλλη, να λέει η Ευρώπη ότι αν δείτε ξαφνικά οι γεωργοί είναι υπεύθυνοι για όλα τα κακό σκήμενα στις χώρες μας. Μα είναι εντελώς άδικο αυτό για τους αγρότες. Διότι, κύριε Επίτροπε, το γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά και το γνωρίζουμε όλοι εδώ, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να έχουμε μια καλή στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο αν δεν συμμετέχουν ε, οι γεωργοί. Καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε μόνο τους καταναλωτές δεν πρόκειται να πάει πουθενά η στρατηγική αυτή. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε στο πλαίσιο στρατηγικής αυτής τους γεωργούς, θα πρέπει να τους ενισχύσουμε, να τους ενδυναμώσουμε. Δηλαδή, Μέσω τη στρατηγική αυτή από το αγρόκτημα στο πιάτο χρειάζονται και τα απαραίτητα μέσα, τα απαραίτητα εργαλεία. Δεν μπορούμε να έχουμε έτσι μια κοινή στρατηγική η οποία να μην συνοδεύεται από χρηματοδότηση. Είμαστε λοιπόν εδώ για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά και για να έχουμε όμως και τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα. Ευχαριστώ κυρία Μύρια Μνάλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, Θέλουμε να προσφέρουμε βιώσιμα τρόφιμα και σε προσιτές τιμές και για όλους. Αυτή είναι στόχη κλειδί και για την Πράσινη Συμφωνία και γι' αυτό προσπαθούμε να προχωρήσουμε τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο σαν μια βοήθεια προς όλους ώστε να μπορούν όλοι να σέβονται αυτούς τους στόχους και να μειώσουμε και τη σπατάλη. Ξέρουμε ότι συνολικά τα ιδιοτροφικά συστήματα είναι υπεύθυνα για το 1 τρίτο των αερίων του θερμοκηπίου. Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο κλάδος ενισχύει το αίτημά μας για ουδετερότητα όσον αφορά τον άνθρακα το 2005. Οι σοσιαλιστές θέλουμε μια στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο που θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τη σπατάλη, που θα μας βοηθήσει να έχουμε πιο βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, αλλά θα δημιουργήσει και νέες ευκαιρίες στην αλυσίδα την διατροφική για όλους. Η στόχη μας επίσης για μείωση των φυτοφαρμάκων, των παρασιτοκτόνων και των αντιβιωτικών και αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Θέλουμε μια πολιτική που να διασφαλίσει επίσης την ανεκνησιμότητα των τροφίμων, να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει τι τρόφιμα τρώει, ώστε να μειωθεί ο καρκίνος και άλλες ασθένειες και να μειωθούν και οι ενδοκρινικοί διαταράκτες. Οι πολιτικές μας λοιπόν πρέπει να προχωρήσουν σωστά και τότε η Πράσινη Συμφωνία θα αποτελέσει πηγή ευκαιρίε και για αυτούς που παράγουν τρόφιμα, και τους αγρότες αλλά και τους αλεί. Είναι και στοιχεία κλειδί για να έχουμε βιώσιμη παραγωγή από την οποία όλοι έχουν να αποφεληθούν. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μάρτιν Χόισικ. Α, όχι, έχει μπλε κάρτα προηγουμένως κάποιος συνάδελφος. Είναι από την κυρία Τούν. Τη δέχεστε την μπλε κάρτα. Ναι, φυσικά λέει κυρία Ντάλη. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ που δέχτηκατε την μπλε κάρτα. Είπατε, αναφερθήκατε στην ανακνευσιμότητα των τροφίμων. Και τι εννοείτε με αυτό. Σημαίνει απόσταση, προέλευση κλπ. Σκεφτήκατε όμως και θα στηρίζατε την ιδέα για ε, την ε, διτή χρήση, δηλαδή ότι στις διαφορετικές αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τρόφιμα έχουν διαφορετική ποιότητα, κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν συνήθως οι καταναλωτές. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Όλοι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν την ίδια ποιότητα τροφίμων όταν η συσκευασία είναι ίδια. Ευχαριστώ πολύ. Απάντηση. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ναι, Βεβαίω, είμαστε απόλυτα σαφείς όσον αφορά αυτήν την διπλή ποιότητα, γιατί πιστεύουμε ότι όλοι οι καταναλωτές, όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουν την ίδια ποιότητα τροφίμων όπου και αν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο κύριο Χόισεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε. Καλωσορίσατε. Γνωρίζουμε όλοι τα μαζικά προβλήματα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αν καταρρεύσει η μελισσοκομεία, χαθούν οι επικονιαστές και λοιπά. Και είναι ε, ένα πολύ επιβλαβές ε, γνωστό φυτοφάρμακο που κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στις μέλισσες. Πολλές φορές ορισμένοι ε, κατηγορούν τους αγρότες. Δεν φταίνε οι αγρότες. Τα βιοσυστήματα θέλουμε να προστατεύουμε. Και εγώ τι περιμένω από τη στρατηγική αυτή, αλλά και από την κοινή γεωργική πολιτική. Να μπορούν να βρουν εναλλακτικέ λύσεις. Έχουμε ε, δεσμευτικούς στόχους μείωση των φυτοφαρμάκων, αλλά και για το hazard. Πρέπει να φύγει αυτό το φάρμακο. Είναι πάρα πολύ επιβλαβές. Ε, και χρειαζόμαστε καλύτερη πρόσβαση στην αγορά για τα εναλλακτικά προϊόντα προστασίας των φυτών. Ελπίζω η στρατηγική αυτή να μην είναι μόνο κενά λόγια, αλλά να φέρει ασφαλή ε, τρόφιμα ε, και προστασία για τους αγρότες, αλλά και προστασία και για τον πλανήτη. Ευχαριστώ. Ο Αντιπρόεδρος, κύριος Σκολάγια, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε όσον αφορά την ενίσχυση των καταναλωτών για να παίρνουν συνειδητέ τεκμηριωμένε αποφάσει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η προστασία των καταναλωτών αποτελούσε πάντα προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δυστυχώ η εμπιστοσύνη των καταναλωτών έχει κλειδονιστεί από την ποιότητα ορισμένων τροφίμων. Μας δίνεται όμως τώρα η ευκαιρία να διορθώσουμε τα κακό κείμενα στα πλαίσια τη στρατηγική αυτή. Μία πρόσφατη μελέτη που έγινε από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο δείχνει ότι η ποιότητα των τροφίμων και των προϊόντων είναι πάρα πολύ σημαντική για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Είναι πολύ σημαντικό οι καταναλωτέ αυτοί να έχουν τι απαραίτητε πληροφορίε. Και το πιο σημαντικό είναι η σήμανση, η ετικέτα που θα πρέπει να ενημερώνει τον καταναλωτή για την προέλευση του προϊόντο. Δεύτερον, η υγειονομικά στοιχεία. Κάποιες ε, δοκιμές δείχνουν ότι υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία πολλούνται με διαφορετική περιεκτικότητα σε γλυκαντικές ουσίες ή σε λιπαρά σε κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τέτοιες αποκλήσεις στα πλαίσια μιας τέτοιας στρατηγικής. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Προκατσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο βρίσκει σύμφωνος και τους γεωργούς και τους καταναλωτές, ιδίω στη δική μου τη χώρα, την Ιταλία. Από την άλλη όμως, η στρατηγική αυτή δεν είναι μια στρατηγική οικονομικά ουδέτερη η σωστή επιλογή που έχει γίνει για την βιολογική βιώσιμη γεωργία ουσιαστικά οδηγεί σε πιο υψηλές τιμές για τα προϊόντα. Αναφέρομαι εδώ πέρα για παράδειγμα στις βιολογικές καλλιέργειες σε σχέση με τις πιο εντατικές βιομηχανοποιημένες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε λοιπόν μια κοινή γεωργική πολιτική που να μπορεί πραγματικά να πλαισιώσει και να προστατεύσει τους μικρούς και μεσαίους γεωργούς έναντι των μεγάλων πολυεθνικών. Αν δεν το διασφαλίσουμε αυτό, τότε θα απλώ σε λόγια χωρί πράξει. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερώνουμε σωστά του καταναλωτέ όσον αφορά την προέλευση των προϊόντων, καθώ επίση και όσον αφορά τη θρεπτική του αξία. Αυτό δεν μπορεί να είναι προαιρετικό. Πρέπει να αποτελεί υποχρέωση, υποχρεωτική ενημέρωση και πρέπει να προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Πίτροφε. Ευχαριστώ, κύριο ε, Μανίου παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μια ευρωπαϊκή επιστημιστική πολιτική είναι εκ των κάνευ έτσι ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικά και υγιεινά τρόφιμα. Εδώ θα πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο αποχώρησης από τα φυτοφάρμακα και να απαγορευτούν τα πιο επικίνδυνα άμεσα, όπως η γλυφοσάτη. Υποστήριξη της βιολογικής γεωργίας. Ε, να μην μειωθεί η χρηματοδότηση του δεύτερου ε, πυλώνα. Να ε, σταματήσουν ε, να δίνουν πολλές πρωτεΐνες στην κτηνοτροφία, αλλά όλα αυτά δεν θα γίνουν χωρίς τους αγρότες που σήμερα δεν μπορούν να επιβιώσουν. Μια χούφτα εκμεταλλεύσεων ε, είναι ιδιοκτήτης πολύ μεγάλων εκτάσεων και μονοπολεί τα κονδύλια. Για να γίνει καλύτερη διανομή ε, θα πρέπει να κοιτάμε πόσοι εργάζονται σε κάθε εκμετάλλευση και όχι την έκταση. Θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 30% όπως προτείνει η Επιτροπή των Περιφερειών η αμοιβή των γεωργών. Μόνο έτσι θα τους επιτρέψουμε να ζουν αξιοπρεπώς και να ανταποκριθούν στην πρόκληση της οικολογικής ε, γεωργίας του αύριο. Ευχαριστώ η κυρία Μόρτλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εξαιότιμη κύριε Επίτροπε. Πολύ θα μας άρεσε σήμερα να συζητήσουμε και με τον συνάδελφό σας κύριο μας, όχι για εκείνον. Η, στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο, χωρίς εμάς που ασχολούμαστε με τη γεωργική πολιτική, ε, είναι ανεπίτρεπτη. Δεν μπορούμε να συζητάμε για τους αγρότες, λες και είναι όλοι εγκληματίες. Θα ξανακατεύουν στους δρόμους, εάν η νομοθεσία σας ε, είναι ακατανόητη για εκείνους. Γιατί αυτοί δεν ε, εργάζονται κατατοδοκούν ή δεν κάνουν ό,τι τους καπνίσει όσο γίνεται περισσότερα λιπάσματα ας πούμε. Ε, ο κύριος Τίμερμανς θέλει να μειώσει δραστικά τα φυτοφάρμακα και να βελτιώσει την ποιότητα των τροφίμων. Πολύ ωραία. Δεν αρχίζουμε από μηδενική βάση. Έτσι κι αλλιώς στην πράξη βελτιστοποιείται η χρήση και μειώνεται. Και τώρα έχουμε ε, επίσημα στοιχεία των αρμόδιων αρχών ελέγχου τροφίμου που λένε ότι είναι τα πιο ασφαλή παγκοσμίω τα δικά μας τρόφιμα. Μην παίζετε με τη φωτιά των ψευδών ειδήσεων. Ε, να ψάξετε να βρείτε καλές λύσεις, όχι ενόχους. Ε, οι ε, αγρότες είναι ανοιχτοί στην καινοτομία, στις καλές ιδέες, αλλά δεν μπορεί η αγορά να τους στραγγαλίζει ε, και να μην πληρώνει, να μην επιβραβεύει τις προσπάθειες, τότε θα πρέπει να τα πληρώσει ο Φρανς Τίμερμανς όλα αυτά. Εμείς χρειαζόμαστε τους αγρότες στην Ευρώπη, τους τιμούμε. Η ε, γεωργία και η δασοκομεία ε, είναι οι μόνες δραστηριότητες που παράγουν οξυγόνο από τη φωτοσύνθεση και δεσμεύουν διοξίδιο του άνθρακα. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να αφήσει ε, ε, αβοήθητους στη βροχή ε, τους αγρότες ο κύριος Τίμερμανς. Δέχεστε μπλε κάρτα, λέει ο πρόεδρος, κυρία Μόρτλερ. Όχι. Κυρία Μόρτλερ, έχετε μπλε κάρτα. Ja, bitte, Α, ναι, ναι. Παρακαλώ, Κύριο Χόισλινγκ. Κυρία Μόρτλερ, γνωρίζετε ότι στην Ιρεμβέργη ε, υπάρχει τώρα μία ε, έκθεση που λέγεται Biofach και χωρίς φυτοφάρμακα μπορούν να δρουν οι αγρότες. Εσείς ε, υπενήσεστε ότι δεν γίνεται καμία γεωργία χωρίς φυτοφάρμακα. Μα έγινε δημοψήφισμα, μεγάλη δημοσκόπηση λαϊκή στη Βαβαρία, μη δεσμευτική, και ο κόσμος είναι προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν θέλετε να αλλάξει τίποτα. Αγαπητές συνάδελφοι, εδώ μου προσάπτεται πράγματα και υποθέτεται διάφορα που δεν είπα. Εμείς πάντα μειώνουμε ε, και λιπάσματα και ε, φυτοφάρμακα. Και μην υποδίεστε ε, ότι στη βιολογική γεωργία δεν χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα και λιπάσματα. Και θα πάω αύριο σε αυτή την έκθεση BioFac, ούτε κρύβομαι και μιλάω με όλους. Τώρα έχασα και τον ήρμό μου. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Θέλω να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι. Γιατί, για ρωτήστε. Γιατί παίρνετε... Ο πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μόρλερ. ακούστε και η ερώτηση. Η κυρία Γιούτελαντ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Πράγματι, είναι ένα θέμα ε, ζωής ή θανάτου στην Ευρώπη. Πρέπει να υπάρξει αυτή η οικολογική μετάβαση για το περιβάλλον, για το κλίμα. Η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της Πράσινης Συμφωνίας και πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή. Ε, μιλάμε για το 1 τρίτο των εκπομπών ε, αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, χάνεται και βιοπικιλότητα. Σκέφτομαι τις μέλισσες τώρα. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μέλισσες. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίσουμε και μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Πρέπει να υποφεληθούμε από αυτή την ευκαιρία. Η γεωργία μας πρέπει να είναι βιώσιμη. Πρέπει να υποφεληθούμε από τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας για να αλλάξουμε την κατάσταση η βιοπικιλότητα στη Γεωργία είναι πάρα πολύ σημαντικό και να ε, φροντίσουμε και για την αντιμετώπιση της αντίστασης στα αντιβιωτικά. Είναι και αυτό μέρος της στρατηγικής. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Σκαρ Κρίστενσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εγώ είμαι γεωργός. Και προφανώ με ενδιαφέρει πάρα πολύ η προτινόμενη από εσά στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο. Τα τρόφιμά μα, αυτά τα οποία τρώμε, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και θα πρέπει να είναι προφανώ υγιεινά, θα πρέπει να είναι θρεπτικά, θα πρέπει να είναι βιώσιμα στην παραγωγή του, θα πρέπει να είναι φιλικά ω προ το κλίμα. Θα μπορούσε να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η εν λόγω στρατηγική, θα καταστήσει πιο εύκολο για το καταναλωτή να μάθει πώ παράγονται τα τρόφιμα, αν είναι φιλικά προ το κλίμα, αν είναι φιλικά προ τα ζώα και αν τα προϊόντα αυτά ουσιαστικά συμβάλλουν στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσα συμπεριλάβει όλα τα είδη αγροκτημάτων, και τα μεγάλα και τα μικρά αγροκτήματα. Και όταν μιλάμε για βιωσιμότητα, κύριε Επίτροπε, δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για μέγεθο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμπεριλάβετε στη δικασία αυτή όλου του γεωργού. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Μικ Ευχαριστώ. Η στρατηγική από το είμαστε στο πιάτο είναι μια ευκαιρία ώστε να αντιμετωπίσουμε συνολικά το θέμα. Το θέμα το πόσο κοστίζει η βιοπικιλότητα, η υγεία, η προστασία ε, των ζών κλπ. Η στρατηγική αυτή αναφέρεται σε στήριξη των παραγωγών κατά την μετάβαση αυτή. Όμως, το θέμα των προσιτών τιμών δεν μας έχει απασχολήσει μέχρι τώρα. Οι αγρότες μας είναι εκείνοι που προσφέρουν τρόφιμα και βιοπικιλότητα. Και είναι σαφές ότι απειλείται αυτή η παραγωγή. Υπάρχει μεταποίηση, υπάρχουν ε, οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και έχει υπάρξει μεγάλη μείωση των μονάδων των μικρών τα τελευταία δέκα χρόνια. Πριν από λίγο καιρό ήταν 20 εκτάριο μέσο όρο. τώρα είναι 33. Στην Ιρλανδία έχουμε χάσει 130.000 ε, μονάδες καλλιέργειας τα τελευταία χρόνια εξαιτία της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στρατηγική αυτή μπορεί να βοηθήσει να αντιστραφεί αυτή η τάση και να φύγουμε από τη βιομηχανική παραγωγή. Ευχαριστώ κύριος Φράνς Πόκοβιτς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι τα τρόφιμα που θέλουμε πρέπει να είναι ασφαλή και ε, ποιοτικά και η παραγωγή να γίνεται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και τα ζώα. Για να πετύχει η πράσινη συμφωνία πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαζόμαστε με τους αγρότες, γιατί αυτοί καλούνται να την εφαρμόσουν την συμφωνία αυτή. Σε αυτή λοιπόν τη στρατηγική και την πράσινη συμφωνία και το αγρόκτημα στο πιάτο, στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής θα πρέπει να ε, υπάρξουν ε, μέτρα που να είναι κίνητρα και όχι φόβητρα για τους αγρότες. Θα πρέπει οι άνθρωποι να κάνουν ευχάριστα αυτά που κάνουν και όχι τρέμοντας και αγωνιώντας. Ωραία, μείωση των φυτοφαρμάκων, μείωση ε, των λιπασμάτων, ε, ε, μικρές αποστάσεις, βραχίες αλυσίδες διανομής και καλές τιμές για τους καταναλωτές αλλά και για τους αγρότες. Δεν θα πρέπει να βάζουμε εμπόδια στους παραγωγούς, ούτε να τους εκμεταλλεύονται τα σούπερ μάρκετ και αλυσίδες διανομής. Να έχουμε θετικό πνεύμα, όχι όλο φόβους και τιμωρίες. Ο κύριος Σίδλ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Επίτροπε. Εγώ περιμένω από τη στρατηγική, από το αγρόκτημα στο πιάτο, μία ε, πρόσβαση σε βιώσιμα τρόφιμα. Ε, εκεί θα πρέπει να συμμετέχουν οι αγρότες, οι καταναλωτές, η μεταποιητική βιομηχανία, λυσίδες, σούπερ μάρκετ, ε, υποχρεωτικά μέτρα για το περιβάλλον, για τη βιοποικιλότητα και μια σειρά άλλων. Είναι η κρίκη της αλυσίδας. Μείωση λιπασμάτων, μείωση φυτοφαρμάκων, μείωση αντιβιωτικών και μάλιστα δραστική, κυκλική οικονομία για να μην έχουμε και σπατάλη τροφίμων. Οπωσδήποτε πρέπει να μειωθεί και αυτή. Και αυτό που χρειαζόμαστε είναι ε, διαφορετική προσέγγιση ε, στις εμπορικές συμφωνίες και σε προϊόντα γενετικής μηχανικής που εισάγονται στην Ευρώπη. Κύριε Πίτροπε, πρόκειται για την αξιοπιστία τελικά όλων των τομέων της πολιτικής μας. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κατάινεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πίτροπε. είναι αναγκαίο να εξετάσουμε το θέμα διατροφής, το θέμα διατροφής πιο συνολικά. Και η στρατηγική αυτή αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε ολόκληρο το θέμα της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων. Αυτό δεν σημαίνει ότι αφήνουμε μόνο του τον αγρότη ή ότι κοιτάμε μόνο αυτόν. Φυσικά και πρέπει να τον έχουμε υπόψη μας, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την μεταποίηση και την μεταφορά και την σπατάλη και την απώλεια τροφίμων. Είναι και αυτά ε, πράγματα που σχετίζονται με τη γεωργία και την επηρεάζουν. Η οδηγία για τις αθέμητες πρακτικές αποτελεί μια αρχή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο μία αποδοτική γεωργία μπορεί να παράγει καλά τρόφιμα και να μας προστατεύσει από την κλιματική αλλαγή. Οι αγρότες πρέπει να έχουν επαρκή έσοδα. Στην Φιλανδία Χαίρομαι πάρα πολύ για την πολιτική που έχουμε όσον αφορά την Γεωργία και ελπίζω και η νέα γενιά να μπορέσει να συνεχίσει τη δραστηριότητα αυτή στην Ήπεθρο. Ευχαριστώ. Έχω μια ανακοίνωση. Κλείνει η εγγραφή για το ΚΑΤΣΙΑΗ γιατί έχουν ζητήσει πολλοί συνάδελφοι το λόγο. Και πρέπει να πω ότι έχουν εγγραφεί να μιλήσουν στο ΚΑΤΣΤΙΑΗ και συνάδελφοι που πήραν το λόγο στη συζήτηση. Καθώς επίσης και συνάδελφοι που ρώτησαν με την μπλε κάρτα. Δεν θα τους δώσω το λόγο και στο ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Πρόκειται για τρεις συναδέλφους, παρακαλώ να το γνωρίζουν, που έχουν δηλωθεί, αλλά έλαβαν ήδη το λόγο. Η κυρία Σνάιντερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, φιλόδοξη είναι η στόχη της στρατηγικής από το αγρόκτημα στο πιάτο, αλλά αυτό θα το κάνουμε μόνο μαζί με τους αγρότες, όχι απέναντι στους αγρότες. Οι προλαλήσαντες από την ομάδα μου το είπαν αυτό. Πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχουν οι αγρότες. Η εκμετάλλευση η γεωργική τι σημαίνει, παραγωγή υγιεινών τροφίμων και δική μας δουλειά είναι να βάλουμε το σωστό θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο. Για μένα είναι πολύ μεγάλη σημασία το γεγονός αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο θα πρέπει να προστατεύει την ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων μας απέναντι στις διεθνείς αγορές. Επιπλέον απαιτήσει όπως η μείωση προϊόντων φυτοπροστασίας θα γίνουν πραγματικότητα μόνο εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο επιτρέψουν την ε, αδειοδότηση και χρήση νέων τεχνολογιών. Επίσης θα πρέπει να έχουν ε, ένα σωστό εισόδημα οι αγρό να αμείβονται για τα προϊόντα και να επιβραβεύονται για το ρόλο που παίζουν για την κοινωνία. Ο καταναλωτής είναι εδώ πρωταγωνιστής. Αν το καταλάβει ο καταναλωτής και πληρώνει αυτά τα προϊόντα, τότε και μόνο τότε θα φτάσουμε σε αυτό το στόχο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα σύστημα ετικετοθεσία ευρωπαϊκό μετά από συνεννόηση. Ευχαριστώ κυρία Κλάρα Αγγιλέρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η πλειοψηφία εδώ στο σώμα είμαστε υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης, ε, του στόχους της, όπως επίσης και με τη Συμφωνία των Παρισιών τόσο η ομάδα μου όσο και περισσότεροι εδώ μέσα θέλουμε αυτούς τους στόχους. Όμως, το να επικεντρωνόμαστε στο πρόγραμμα αυτό, τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο ή την πράσινη συμφωνία να μιλάμε για μεγάλες αλλαγές στη γεωργία χωρίς να αναγνωρίζουμε τι ήδη γίνεται, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να επικεντρωνόμαστε μόνο στα φυτογενομικά μέτρα. Είναι σημαντικά, αλλά πρέπει συγχρόνως να διευκολύνουμε τους αγρότες ώστε να μπορούν να καινοτομήσουν, να καταπολεμήσουν την χρήση των φαρμάκων κλπ. Πρέπει να υπάρχουν και εναλλακτικέ, συνεπώς. Χωρίς να δεσμευτούμε υπέρ της γεωργίας και των αγροτών, δεν είναι δυνατόν η στρατηγική αυτή να θριαμβεύσει. Οπότε με τη δέσμευση όλων να προχωρήσουμε, αλλά να μην ξεχάσουμε τους αγρότες. Ευχαριστώ. Η κυρία Αλίεβα Βέλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Σε παγκόσμιο επίπεδο φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να θέσει τους κανόνες για ένα βιώσιμο γεωργικό σύστημα, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί όμως μόνο μέσω μιας δίκαιης, ισορροπημένης προσέγγισης. Αν θέλουμε να έχουμε πραγματικά μια φιλόδοξη στρατηγική και μια επιτυχημένη μετάβαση, θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητη χρηματοδότηση και να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ως προς αυτό λοιπόν καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει συνέργεια μεταξύ των διαφορετικών στρατηγικών και μέσων χρηματοδότησης, να συμπεριλαμβάνονται όλα αυτά στην κοινή γεωργική πολιτική και βέβαια και στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο. Και θα πρέπει να υπάρχει και μια ενιαία αμοιβαιότητα ανάμεσα σε όλε αυτέ τι πολιτικέ. Προφανώ οι γεωργοί μπορούν να δραματίσουν σημαντικότατο ρόλο στην επίτευξη των στόχων στρατηγική. Άρα πρέπει να του βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα απαραίτητα κίνητρα. Μερικές φορές ε, οι γεωργοί κατηγορούνται ότι δεν λειτουργούν σωστά. Μόνο αν λοιπόν εμείς διασφαλίσουμε τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, όλων των διαφορομένων, τότε θα καταφέρουμε να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση και θα στεφτεί με Κυρία Σόιντροβα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, δεν είναι εύκολη η θέση σας καθόλου. Οι αγρότες παρακολουθούν τούτη εδώ τη συζήτηση. Γιατί ξέρουν ότι έχει σχέση με εκείνους και περιμένουν να τους υποστηρίξουμε. Γνωρίζουν την κλιματική αλλαγή και τι σημαίνει ο αντίκτυπός της. Και ότι θα πληρώσουν εκείνη την ύφη. Δεν είναι μόνο η Πράσινη Συμφωνία, είναι πολλά περισσότερα. ας πούμε στην τσεχική δημοκρατία, άμα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα φυτοφάρμακα, θα πολλαπλασιαστούν οι αρρώστιες των φυτών λόγω της κλιματικής αλλαγή και της υπερθέρμανσης. Επίσης, κοιτάξτε παρακαλώ τι φθηνέ εισαγωγέ από τρίτε χώρε. Ε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τις αλυσίδες διανομής. Ε, οι καταναλωτές ε, ψωνίζουν τώρα πια όλοι σε σούπερ μάρκετ, τα οποία σούπερ μάρκετ έχουν τεράστια εξουσία απέναντι στους αγρότες. Τι κάνουμε με τις αλυσίδες διανομής. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους αγρότες που ζουν στην υπεθρό και που νοιάζονται για τη βιοπικιλότητα, για τα δάση, για τη φύση γενικότερα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μορέτη. Κύριε Επίτροπε, η διατροφική αλυσίδα ουσιαστικά ευθύνεται για ένα σημαντικό ποσοστό όσον αφορά τι εκπομπέ του εξτρίου του άνθρακα. Άρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια πρόκληση. Αυτή τη στιγμή καλούμεθα να παράγουμε περισσότερο με λιγότερου σπόρους ενώ παράλληλα πρέπει να διασφαλίσουμε και την ποιότητα και τη βιωσιμότητα. Οι πολίτε όμω ζητάνε αυτή τη στιγμή ασφάλεια και διαφάνεια, αλλά η νομοθεσία από μόνη τη δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε μια σημαντική αλλαγή του όλου συστήματο, ακόμα και του τρόπου ζωή μα. Η ολιστική λοιπόν σφαιρική προσέγγιση είναι θεμελιώδου σημασία. Μεγαλύτερη συνέργεια ανάμεσα στι ε, υγειονομικέ γεωργικέ υπηρεσίε που θα πρέπει να αλλοσυμπληρώνονται και να μην βρίσκονται σε αντιπαράθεση. Επίση, θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε την αξία των τροφίμων. Ότι θα πρέπει τα τρόφιμα ουσιαστικά να είναι βιώσιμα, υγιεινή να αυτά τα οποία καταλήγουν στο πιάτο μα. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ουσιαστικά μια, ένα ομοιόμορφο σύστημα ετικετοθεσία και σήμανση που να ενημερώνει του καταναλωτέ χωρί να το παραπλανεί, χωρί να το επηρεάζει. Ένα σύστημα ετικετοθεσία που να βασίζεται μόνο σε επιστημονικά δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λετσέ. κύριος Μπενουάλιο Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πίτροπε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι έχω πολύ την πιστοσύνη στην ευρωπαϊκή παραγωγή, σε ό,τι παράγεται σε εμά και από ό,τι άκουσα σήμερα το πρωί, πριν να το λέμε και να το ξαναλέμε και να ευχαριστούμε του αγρότε μα. Η στρατηγική τώρα από το αγρόκτημα στο πιάτο συμβιβάζει τον καταναλωτή με τον αγρότη για τρία πράγματα. Πρώτον, στη στρατηγική αυτή πρέπει να συμμετέχει ο γεωργικό κόσμο, γιατί όντω εμπλέκονται στη στρατηγική αυτή, όπω και οι καταναλωτέ. Δεύτερον, να υπάρχουν νέε εγγύησει όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τι επενδύσεις για να πετύχει η μετάβαση αυτή. Οι αγρότες δεν είναι αυτοί που θα πρέπει να διορθώνουν τις ελλείψεις στον προπολογισμό ή να φροντίσουν μόνοι τους για την Πράσινη Συμφωνία. Και τρίτον, προστασία. Προστασία των καταναλωτών, προστασία των ε, γεωργών, του περιβάλλοντος, πράγματα που δεν μπορούν να πετύχουν παρά μόνο αν υπάρχουν ε, έλεγχοι ενισχύσεις, έλεγχη των προϊόντων που έρχονται στην επικράτειά μας και να υπάρχει και δικαιοσύνη απέναντι στους αγρότες και τους καταναλωτές. Ευχαριστώ και πάλι για τη στρατηγική σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λουτσιέν. Ε, ο κύριος Μοχάμετ Σα... Σαχίμ λέγομαι. Να σας βοηθήσω. Σαχίμ. Ευχαριστώ. Yeah. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, πρόεδρε, επίτροπε, τώρα θα πρέπει να πιάσουμε τον Ταύρο από τα κέρατα ή την αγελάδα από τα κέρατα. Αυτή η στρατηγική χωρίς αναρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, είναι μια τρύπα στο νερό. Κάθε μέρα εργάζονται σκληρά οι αγρότες για να φτιάχνουν τίμια προϊόντα για μας. Φροντίζουν τα ζώα τους και θα πρέπει να έχουν και υπεύθυνη χρήση με τη ε, φύση. Και δεν αναγνωρίζεται αυτό, δεν υποστηρίζονται. Το μόνο κοινό σε αυτή την πολιτική είναι ότι σχεδόν σε κάθε κράτος μέλος το 80% της επιδότησης πάει στους 20 πλουσιότερους. Και αυτό είναι στους 100. Αν το πάμε στους 200 δεν υπάρχει ούτε ένας αγρότης, αλλά μεγάλοι γεωκτήμονες και πολυεθνικές εταιρείε ε, που έχουν τζίρο εκατομμύρια για να μην πω εκατομμύρια. Και βεβαίως χαιρόμαστε για τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο, αλλά χωρίς μεταρρύθμιση της ΚΑΠ εγκαταλείπουμε τους αγρότες που ε, διαχειρίζονται σωστά τη γη τους και το νερό και φέρνουμε νερό στο μήλο των ε, μεγάλων πολυεθνικών και των μεγάλων γεωκτημόνων και κτηνοτρόφων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καλινόφσκι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, Οι Ευρωπαίοι γεωργοί αντιμετωπίζουν τώρα νέες προκλήσεις και επιβαρύνονται με νέα καθήκοντα λόγω της νέας Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ο νέος προτινόμενος όμως προϋπολογισμός για τη γεωργία από ό,τι φαίνεται θα μειωθεί. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αποκλείεται να στεφθεί με επιτυχίε στρατηγική σα. Θα πρέπει άμεση άμεσε ενισχύσει να πηγαίνουν πραγματικά στου γεωργού. Μιλάμε για μια πραγματική παθολογία αυτή τη στιγμή του συστήματο. Υπάρχουν ε, πολλοί οι οποίοι λαμβάνουν άμεσα ενισχύσει και δεν είναι γεωργοί, αλλά είναι απλώς ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων. Λοιπόν, κύριε Επίτροπε, τι προβλέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να μειώσει την κατανάλωση συγκεκριμένων προϊόντων και για να μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μέσω της γεωργίας. Από ό,τι φαίνεται αυτό είναι ο βασικό πυλώνα τη στρατηγική σα, έτσι δεν είναι. Μήπω όμω αυτό οδηγήσει τελικά σε μειωμένο εισόδημα για του γεωργού. Ευχαριστώ. Η κυρία Κάρμεν Αβραμ, παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ. Η Πράσινη Συμφωνία είναι κάτι πολύ σημαντικό και οι αγρότες αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες και μάλιστα κάτω από συνθήκες που δεν είναι σαφείς. Πρέπει να προσφέρουν καλά τρόφιμα σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, εκατομμύρια. Σήμερα όμως η Γεωργία φαίνεται να είναι πολύ δύσκολη υπόθεση, πολύ ακριβή και εξαρτάται από πολλούς ε, άγνωστους παράγοντες. Γι' αυτό και πάρα πολλοί αγρότες εγκαταλείπουν τις δραστηριότητές τους και πολλοί άλλοι σκέφτονται να το κάνουν. Οπότε πώς θα αντικατασταθούν οι αγρότες αυτοί που εγκαταλείπουν. Οι νέες γενιές πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι θα φροντίσουν για την επιτυχία της γεωργίας. Και πρέπει συγχρόνως με τις φιλόδοξες στρατηγικές μας να ξεκινήσουμε ένα επίγονο πρόγραμμα δίνοντας κίνητρα στους νέους να επιστρέψουν στην Ήπεθρο και στη γεωργία και να προχωρήσουν εκείνη την επανάσταση για την οποία συζητάμε εμείς σήμερα. Ευχαριστούμε κυρία Σαντέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο μπορεί να προσφέρει πολλά στον ε, αγροτροφικό μας τομέα και στον ε, καταναλωτή. Αλλά για να πετύχει πρέπει να υπάρχει συνέπεια και ρεαλισμός. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια γιατί η κλιματική πρόκληση απαιτεί κονδύλια στο ύψος της πρόκλησης ακριβώς αυτής. Δεν μπορούμε να περιμένουμε περικοπές Όπω προτείνονται και από την άλλη να ζητάμε τους αγρότες να κάνουν περισσότερα με λιγότερα. Επίσης, πρέπει να βελτιωθεί η διάρθρωση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και της Πράσινης Συμφωνίας. Χρειάζεται ρεαλισμός, γιατί πρέπει τις αποφάσεις μας να τις βασίζουμε στην επιστήμη και όχι στην ιδεολογία. Να μην βάλουμε τον κλάδο σε αδιέξοδα, αλλά να χρησιμοποιούμε καινοτομία τεχνολογική τη στιγμή που ο κόσμο προχωράει προς αυτή την κατεύθυνση. Και μην ξεχνάμε ότι οι ακρότες μας είναι η λύση και πρέπει αυτοί να βρεθούν στο κέντρο τη στρατηγικής μας. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της οικονομικής βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα ακολουθεί η διαδικασία Έχουν ζητήσει το λόγο ένα διαδικαστικό. Ο κύριος Μάντερς, είπατε ότι όσοι έκαναν ερώτηση με μπλε κάρτα δεν δικαιούνται να πάρουν το λόγο στο ΚΑΤΣΙΑΙ. Ε, αυτό να το γράψει ο κανονισμό. Εγώ διαμαρτύρομαι. Αν μα το είχατε πει από την αρχή, δεν θα είχα σηκώσει μπλε κάρτα. Διαμαρτύρομαι εντόνω για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΙ. Καμία σχέση έχει με τον κανονισμό, κύριε Μάντερ, αυτό. Δεν χρειάζεται να εγγραφεί στον κανονισμό. Γιατί ο κανονισμός λέει ότι αποφασίζει ο πρόεδρος πόσες μπλε κάρτες θα δώσει. Αλλά όταν ανέλαβα την Προεδρία σας ανακοίνωσα τι θα κάνω γιατί είχα πάρα πολλά αιτήματα για το ΚΑΤΣΔΙ και έχω. Κάπως πρέπει να το ρυθμίσω. Ο κύριος Μπασέσκου, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η γεωργία είναι ένας οικονομικός τομέας, μια οικονομική δραστηριότητα θεμελιώδου σημασίας, ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη και βέβαια και για τη χώρα μου, τη Ρουμανία. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι ο ανταγωνισμός στην ευρωπαϊκή αγορά μεταξύ των ίδιων των γεωργών είναι ιδιαίτερα έντονο, τρευλωμένο πάρα πολλέ φορέ και λόγω των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων. Για παράδειγμα, νεκτάριο στη Ρουμανία έχουμε επιδοτήσει 109 ε, ευρώ, ενώ στη Γαλλία είναι 220 ευρώ η αντίστοιχη επιδότηση ανά εκτάριο. Δεν λέω ότι θα πρέπει να μειωθούν οι επιδοτήσει που πηγαίνουν στη Γαλλία, αλλά τουλάχιστον κύριε Επίτροπε, α αυξηθούν οι δικέ μα, οι επιδοτήσει που πηγαίνουν στη Ρουμανία στου Ρουμανού γεωργού. Το ίδιο φαινόμενο όμως βλέπουμε και στην κτηνοτροφία. Έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου οι πρώτες ύλε εισάγονται από, τις, από τα παλιά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στη δική μου τη χώρα οι πρώτες ύλε είναι πια πάρα πολύ ακριβές. Ο κύριος Ολέκας. Κύριε Ολέκας, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ο κύριος Ολέκας απουσιάζει η κυρία Χίλντε Βότμανς. Βότμανς, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφε. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλή η συζήτηση. Η στρατηγική ε, από το αγρόκτημα στο πιάτο, οπωσδήποτε σημαντικό. Εγώ είμαι κόρη αγρότη και πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε τι κάνουμε για τους αγρότες μας. Δεν είναι από δύο Πομπέι τράγοι. Φυσικά θα πρέπει οι αγρότες να συνεργαστούν και για την Πράσινη Συμφωνία και για τα μέτρα. Αλλά ας είμαστε ειλικρινεί. Τα τελευταία χρόνια κρατηθείτε κάθε μέρα έκλειναν ε, ε, ε, χίλιες γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χίλια αγρότες κατεβάζουν ρολά, βάζουν λουκέτο πολλά χρόνια. Στην ε, Φλάνδρα έχουμε ένα ωραίο τηλεπτικό πρόγραμμα «Αγρότης μόνος ψάχνει». Ε, σε λίγο θα ψάχνουμε εμείς τους αγρότες. Τι θα κάνετε, θέλετε να υπάρχουν αγρότες στην Ήπεθρο. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη θέση των αγροτών στην διατροφική αλυσίδα, νέες αγορές, να υποστηρίζουμε ε, τους ε, αγρότες μας. Ακόμα η Ρωσία μποϊκοτάρει τα γεωργικά μας προϊόντα. Κύριε κυρία Πιετικάινεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μας παρουσιάσετε τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο. Ελπίζω ότι η στρατηγική αυτή θα επικεντρωθεί στην παραγωγή βιώσιμων τροφίμων υψηλής ποιότητος που θα λαμβάνει υπόψη όλη την αλυσίδα παραγωγής από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι την απώλεια ή ακόμα και τη σπατάλη των τροφίμων. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για την υγεία των πολιτών και τις καλύτερες λύσεις που θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Και βέβαια, Γεωργή, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να μειωθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η τρέχουσα κοινή γεωρική πολιτική και η προβλεπόμενη χρηματοδότηση για την κοινή γεωρική πολιτική δεν πρόκειται να φέρει τα αναμενόμενα αυτά αποτελέσματα. Θα βελτιώσετε λοιπόν τις προτάσεις για την κοινή γεωρική πολιτική προκειμένου να μπορούμε να έχουμε πραγματικά βιώσιμα τρόφιμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Γνωρίζω καλά τον αγροτικό κόσμο και τις επιπτώσεις που είχε η, και έχει η κλιματική αλλαγή στην ζωή των αγροτών μας. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε δίκαια έσοδα ώστε οι αγρότες μας να παράγουν τρόφιμα ποιότητας και να αποφεύγεται η κατάληψη της υπαίθρου και της γεωργίας. Πώς να διασφαλίσουμε λοιπόν καλά τρόφιμα με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζονται και δίνουν σημασία μόνο στην ανταγωνιστικότητα με μοντέλα που τελικά δεν είναι βιώσιμα για τη γεωργία και θέτοντας σε κίνδυνο τελικά την βιωσιμότητα. Η κατανομή η προστασία των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του γεωργικού κόσμου πρέπει να αποτελούν μέρος της στρατηγικής αυτής και όχι μόνο τα συμφέροντα που εσείς εκπροσωπείτε και εξυπηρετείτε. Ευχαριστώ κύριο Σαλβατόρε Ντεμέιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε. Τη δύσκολη αυτή λεπτή στιγμή η γεωργοί είναι ουσιαστικά ένα ζωντανό τμήμα της οικονομίας. Εργάζονται πραγματικά, κάνουν πραγματικές θυσίες. Έχουν μια τεχνογνωσία η οποία περνάει από γενιά σε γενιά. Επομένως, ε, μιλάμε πολύ συχνά για προκλήσεις, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι οι προκλήσεις δέχονται σε καθημερινή βάση Γεωργή, γεωργοί και είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν και άλλες μελλοντικέ προκλήσεις, αλλά θα πρέπει πραγματικά να είναι πρωταγωνιστές της όλης διαδικασίας και όχι ένοχοι της όλης διαδικασίας. Μάχονται προκειμένου να έχουμε πραγματικά μια βιώσιμη γεωργία, η οποία δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Α μην ξεχνάμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική είναι αυτή που έφερε κοντά του Ευρωπαίου πολίτε και συνέβαλε πραγματικά πραγματικά στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτή την πρόκληση αλλά και με άλλε προκλήσει. Λέτε τώρα ότι θα πρέπει να δούμε την εποχικότητα, ότι θα πρέπει να δούμε τις διαφορές που υπάρχουν από τη μία περιοχή στην άλλη. Λέμε ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε καμία περίπτωση αυτοματισμούς, αλγόριθμους. Ας σεβαστούμε τις ιδιαιτερότητες της κάθε γεωργικής περιοχής. Ευχαριστώ κύριος Μίλαν Ούρεκ. Είναι παρόν. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριο Σούρικ. Εμείς εκπονούμε τώρα μια νέα στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο και στη Σλοβακία. Ε, και εκεί προσκρούσαμε στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για τις γεωγραφικές ε, ε, προελεύσεις, την ομασία γεωγραφικής προέλευσης. Ε, οι αγρότες πιέζονται και πρέπει να ρίχνουν τις τιμές. Η στραματική ενίσχυση δεν είναι δίκαιη. Στη χώρα μου, ανά εκτάριο, είναι η ενίσχυση 200 ευρώ στις γειτονικές χώρες, Αυστρία και λοιπά, είναι πολύ υψηλότερη. Και μερίδα του λέοντος την παίρνουν μεγάλες εταιρείε και μεγάλες εκμεταλλεύσεις. Ποια στήριξη μικρών ε, ε, αγροτών. Ο συνάδελφος ε, Τσοχεντάρου. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να διασφαλίσει τα εξής. Πρώτον, να στηρίζει τους αγρότες και εδώ μιλάω για τις ε, ενισχύσεις και για κίνητρα. Όλοι θέλουμε ασφαλή τρόφιμα, ε, αξιοπρέπει συνθήκες εργασίας και προδιαγραφές. Δεύτερον, στήριξη για το περιβάλλον. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να προσφέρει συγκεκριμένα και δεσμευτικά μέτρα. Εγώ είμαι από τη Ρουμανία οι ίδιες ενισχύσεις για τους ε, Ρουμάνους, οι ίδιες πρέπει να είναι με τους Γάλλους, τους Γερμανούς κτλ. Να έχουμε επίσης τις ίδιες ε, προδιαγραφές και την ίδια ποιότητα τροφίμων που να πουλιέται παντού στην Ευρώπη. Και τρίτον, να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα διαβούλευσης, βάσει του οποίου οι αγρότες από ολόκληρη την Ευρώπη θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τα προϊόντα τους. Ο κύριος Κέλλη, τελευταίος, αλλά όχι φυσικά λιγότερο σημαντικός. Με τον συνάδελφό μου τον κύριο Βάλλες δεν συμφωνώ πάντα, αλλά αυτή τη φορά συμφωνώ απόλυτα στη διάκριση που κάνει ανάμεσα τις μεγάλες μονάδες και καλλιέργειες και τους μικρούς αγρότες, τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που υπάρχουν και παράγουν τρόφιμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προστατεύοντας το περιβάλλον. Νομίζω λοιπόν ότι οι μεγάλες βιομηχανίες που εμπορεύονται τα τρόφιμα ε, δεν πρέπει να περνάνε έτσι. Πρέπει να υπάρχει διάκριση ανάμεσα αυτές και τις ε, μικρές ε, ποιοτικέ εκμεταλλεύσεις. Και τώρα υπάρχει μια ευκαιρία στο επόμενο βήμα για την επόμενη κάπου και μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής της καινούρια να γίνει αυτή η διάκριση. Όσοι το αξίζουν να παίρνουν την στήριξή μας και κυρίως αυτοί οι οποίοι παράγουν ε, τρόφιμα ποιότητας και όχι βιομηχανικά. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Παρακαλώ τον Επίτροπο τον κύριο Βοητσεχόφσκι να πάρει το λόγο για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σας ευχαριστώ για τις δηλώσεις σας, για τις παρατηρήσεις σας. Νομίζω ότι δεν θα έχω το χρόνο για να απαντήσω σε κάθε ερώτηση και παρατήρηση ξεχωριστά, ωστόσο πρέπει να σας πω ότι όλη η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αναγκαία, επίκαιρη και επικοδομητική. Να ευχαριστήσω λοιπόν την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξη Πέθρου και τον κύριο Λίνς. Δεν έχουμε οριστικοποιήσει ακόμα τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο. Βρίσκεται σε εξέλιξη. Αποφασίσαμε απλώς για κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, διότι Υποβλήθηκε επίσημα η πρόταση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη οποία αναπόσπαστο μέρος αποτελεί στρατηγική αυτή. Αναφερθήκατε σε κάποιες πολύ σωστές ιδέες. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτές λίγο. Ξέρετε ότι ασχολούμαι με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και με τη γεωργική της πτυχή. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω όλες τις παρατηρήσεις ή τις περισσότερες τουλάχιστον από αυτές που κάνατε. Ωστόσο, πρέπει να σα υπενθυμίσω ότι η Επίτροπος Κυριακίδης, ε, που Κυριακίδη, που είναι υπεύθυνη για την υγεία, ε, έχει επίσης ένα καθοριστικό ρόλο και για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Αλλά από τη δική του πλευρά βέβαια εξίσου σημαντική είναι και η γεωργοί και θα πρέπει όντω να διδραματίζουν κέριο ρόλο. Συμφωνώ απόλυτα λοιπόν με αυτό που είπατε, ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να λειτουργήσει υπέρ των γεωργών και όχι κατά των γεωργών. Θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα κίνητρα. Γι' αυτό το λόγο στην πρωταρχική μου δήλωση αναφέρθηκα στον προπολογισμό. Διότι αν πραγματικά θέλει κανεί να δώσει τα απαραίτητα κίνητρα στου γεωργού για να χρησιμοποιούν λιγότερα λοιπάσματα, λιγότερα φυτοφάρμακα, να διαχειρίζονται καλύτερα τα ύδατα, τότε θα πρέπει να του δώσει και του απαραίτητου πόρου, έτσι δεν είναι. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να προβλέπονται στον πρώτο πυλώνα, τα οικολογικά συστήματα και προγράμματα, καθώ επίση και όλα αυτά τα οποία πρέπει να συμπεριλάβουμε στον δεύτερο πυλώνα. Αναφερθήκατε στη σειρά την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Συμφωνώ μαζί σας. Και εγώ θα ήθελα να εγκριθεί πρώτα η στρατηγική και εν συνεχεία μόνο να γίνουν οι απαραίτητε μεταρρυθμίσει στην κοινή γεωργική πολιτική. Δυστυχώ όμω, από το 2018 συζητάμε τη μεταρρύθμιση τη κοινή γεωργική πολιτική και Η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη κυρία Φοντελάιεν αυτή τη στιγμή δεν έχει υποβάλει νέα πρόταση εκ νέου μεταρρύθμιση τη κοινή γεωρική πολιτική. Το κεφάλαιο αυτό δεν μπορούμε να το ανοίξουμε τώρα, δεν έχουμε το απαραίτητο χρόνο. Θα πρέπει πάντως να γίνουν απαραίτητε προσαρμογέ στη νέα αυτή κοινή γεωργική πολιτική και θα είμαστε σε επαφή προφανώ και με το Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο προκειμένου νέοι κανόνε τη κοινή γεωργική πολιτική να αντανακλούν στο μέλλον τι βασικέ πτυχές τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο. Η στρατηγική αυτή αποτελεί ευκαιρία ιδίω για τι μικρομεσαίες αγροτικέ επιχειρήσει, οι οποίε, όπω είπατε εξαφανίζονται πάρα πολύ γρήγορα. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, στην Ευρώπη υπάρχει ο απαραίτητος χώρος και για πιο εντατικές αν θέλετε βιομηχανίες, αλλά και για μικρότερες ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ιδίως αυτές οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις είναι έτοιμες, θεωρώ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες περιβαλλοντικές προκλήσεις. Δεν θέλουμε όμως ε, οι μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις να κάνουν τι μικρές να εξαφανιστούν. Χρειαζόμαστε ισορροπία, χρειαζόμαστε βιωσιμότητα. Και αυτό θα πρέπει να ισχύει μεταξύ των πολλών διαφορετικών αγροκτημάτων. Βέβαια και η βιολογική καλλιέργεια είναι πάρα πολύ σημαντική και θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο στα πλαίσια της στρατηγικής από το αγρόκτημα στο πιάτο, όχι μόνο προς το μέγεθός της, θα θέλαμε να προωθήσουμε όχι μόνο τη βιολογική καλλιέργεια, αλλά και τη βιολογική κατανάλωση. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι πολίτε να εκτιμούν περισσότερο πλέον τα βιολογικά προϊόντα. Και θα έλεγα ότι αυτό αποτελεί ήδη μία επιτυχία τη Ευρωπαϊκή Γεωργία. Το ότι έχουμε πάρα πολύ καλά γεωργικά προϊόντα και βιολογικά γεωργικά προϊόντα, τα οποία τηρούν τα ύψιστα πρότυπα ποιότητα και ασφάλεια παγκοσμίω. Νομίζω λοιπόν θα πρέπει προφανώ να υπερασπίσουμε του παραγωγού τροφίμων, Πολλοί αναφερθήκατε στην προστασία των γεωργών σε σχέση με εισαγωγέ. Προφανώς θα πρέπει να έχουμε τα ίδια πρότυπα για τα προϊόντα τα οποία έρχονται από τρίτες χώρε. στην εσωτερική μας αγορά. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι έχουμε και την εργαλειοθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Τώρα, όσον αφορά τη γραφειοκρατία, τα στρατηγικά σχέδια θα είναι καθοριστική σημασία, θα πρέπει να επεξεργαστούμε βέβαια ακόμα περισσότερο και σας υπόσχομαι ότι η αξιολόγηση των εθνικών αυτών προγραμμάτων θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία, προκειμένου σε καμία περίπτωση η γραφειοκρατία αυτή να μην αποτελεί τροχοπέδι στην δραστηριότητα των γεωργών. Αυτό έχει συμβεί μερικές φορές στο παρελθόν και θα πρέπει να αποφευχθεί. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση που είχαμε, όχι μόνο εδώ, στην Ολομέλεια, εν γέννη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ πλέον ότι οι γεωργοί έχουν μεγαλύτερη βεβαιότητα και προβλεψιμότητα για τις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σας διαβεβαιώνω μία ακόμα φορά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο να εφαρμοστούν για τους γεωργούς υπέρ των γεωργών και για το καλύτερο δυνατόν μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Σας ευχαριστώ. Με την τοποθέτηση του κ. Επιτρόπου ολοκληρώνεται η συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Και ερχόμαστε στο επόμενο θέμα της μέρης της διάταξης. Ακολουθούν οι συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπινών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Η πρώτη συζήτηση αφορά τη Γουινέα Κόνακρη, ιδίως τη βία σε, βάρος συγγνώμη, ε, διαδηλωτών. Θα αρχίσει η συζήτηση με τους συντάκτες ε, του ψηφίσματος. Έχει το λόγο πρώτη η κυρία Πιερέτ Χέρτσμπεργκερ Φοφανά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ε, δημοκρατία της Γουινέας δοκιμάζεται. Ε, είναι έντονη η βία που απειλεί την δημοκρατική σταθερότητα. Η πολιτική εξουσία και η κυριαρχία είναι και θα πρέπει να παραμείνει στα χέρια του λαού. Θα πρέπει να γίνει σεβαστή η λαϊκή βούληση στους κρατικούς θεσμούς. Από πέρυσι που ε, εξαγγέλθηκε δημοψήφισμα για την τροποποίηση του συντάγματος, η, πολιτική, η αντιπολίτευση και η κοινωνία των πολιτών αμφισβητούν αυτό το προσχέδιο και το ε, πολιτικό κλίμα ε, ε, χαρακτηρίζεται από βία. Ακούμε τι γίνεται για αστυνομική βία, παίρνουμε εκθέσεις και αυτό έχει συγκινήσει τον κόσμο και τον έχει ανησυχήσει. Συγγνώμη, ακούω τον κόσμο γύρω-γύρω να μιλάει και δεν μπορώ. Κύριε Αρενά, σας παρακαλώ, δεν μπορώ να ακούσω τη φωνή μου. Ε, συγγνώμη πρόεδρε, αλλά δεν μπορώ να μιλώ όταν κάποιος μιλάει δίπλα μου. Τι να κάνουμε τώρα. Έλεγα λοιπόν. Ζητώ συγγνώμη. Όταν η αστυνομία, ας πούμε, χρησιμοποίησε μια γυναίκα ως ασπίδα για να προστατεύεται από τις πέτρες που πετούσαν οι διαδηλωτές, ο κόσμος ολόκληρο συγκλονίστηκε από τη βία αυτή. Είναι κρίσιμο το ερώτημα που μπορούμε να θέσουμε. Πόθεν αυτή η βία, τι την προκαλεί. Ενθαρρύνουμε τη Γουινέα να ανοίξει ε, ένα διάλογο για να βρεθούν ιδανικέ απαντήσεις σε αυτές τις ε, ε, σημαντικές ερωτήσεις με συμμετοχή του κόσμου για να λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες πολιτικές ιδέες με τρόπο ε, ειρηνικό και χωρίς αποκλεισμούς. Ε, καλούμε επιγόντως τη Γουινέα να σταματήσει αυτό το δηλητηριασμένο κλίμα. Δεν είναι δυνατόν να ρίχνουν χημικά, δακρυγόνα, ξύλο στους διαδηλωτές και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ε, ρισκάρουν τη ζωή τους την ίδια κατεβαίνοντας στη διαδήλωση. Η κυβέρνηση λέει ότι η χώρα είναι κυρίαρχη και καμία άλλη χώρα εξωτερική ή πολιτικός φορέας δεν μπορεί να παίρνει αποφάσεις για την ίδια. Ωστόσο στο εσωτερικό ε, της χώρας απειλούνται εκείνοι που δεν ε, υποστηρίζουν την πολιτική γραμμή που έχει επιλέξει η κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, ε, να έχει σχέσεις με την Αφρική, με διαφορούς παράγοντες και φορείς, να υποστηρίζει ε, τους αγωνιστές ανθρωπινών δικαιωμάτων για μια δημοκρατία χωρίς αποκλεισμούς, όπως εδώ έτσι και στους συναδέλφους στην Αφρική. Αγαπητοί συνάδελφε, σας άφησα 45 δευτερόλεπτα παραπάνω. Στο μέλλον παρακαλώ, θα σας παρακαλούσα να τηρείτε το χρόνο σας και να μην κάνετε τέτοιες ε, παρατηρήσεις ενδιάμεσες. Η κυρία Μαρία Ρενά έχει το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο πρόεδρος Κοντέ θα πρέπει να αποδεχθεί την πραγματικότητα γιατί η παράταση της θητείας του σπήρε ζάνια αστάθειας ε, στη Γουινέα και στην περιοχή. Και μάλιστα οι διαμαρτυρίε κοινωνία των πολιτών κατά του δημοψηφίσματο προκάλεσαν την βία καταστολή από τι δυνάμει ασφαλεία, που ουσιαστικά άνοιξαν πύρα απέναντι σε άμαχο πληθυσμό. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, να υπάρχει ανάλογη απάντηση και, γιατί ήδη έχει δημιουργηθεί μια κρίση εδώ και χρόνια στην περιοχή. Από τον Οκτώβριο του 2019 τουλάχιστον 28 πολίτες έχουν χάσει τη ζωή τους και από το 2015 πάνω από 70 διαδηλωτέ έχασαν τη ζωή του. Ε, έχει βγει στην αντιπολίτευση, δεν υπάρχει ελευθερία έκφραση ε, και ο πληθυσμό είναι φοβισμένο. Απευθύνουμε έκκληση στην κυβέρνηση τη Γουινέα να διαχειριστεί καλύτερα τι διαδηλώσει, να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ασφαλεία για του διαδηλωτέ και επίση να ξεκινήσει ανοιχτή αμερόληπτη έρευνα κατά των δραστών της βίας και των ε, φόνων. Επίσης, ε, πολλά μέλη της αντιπολίτευσης φυλακίστηκαν ε, ασκώντας την ελευθερία έκφραση και το δικαίωμα του, συνε, ε, η παράταση της θητείας για τρίτη φορά καταστρατηγεί τη δημοκρατία. Ο Αλφα Κοντέ ήταν κάποτε υπέρμαχος της δημοκρατίας και της αναλέγης θα πρέπει να θυμηθεί τις ρίζες του λοιπόν. Επίσης ζητούμε από τον Πρωθυπουργό να συνεργαστεί με την ΕΚΟΒΑΣΗ για να βρεθεί μια πολιτική λύση. Επίσης, καλούμε την ΕΙΕΔ να σταθεί στο πλευρό της Γουινέας σε μια προσπάθεια διαλόγου και μεσολάβησης για να αντιμετωπιστούν ε, οι βιοπραγίες που συνδέονται με τις εκλογές. Σας ευχαριστώ κύριο Τσαρνέτσκι τώρα για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Πιστεύω ότι θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση, πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι εκκλήσεις μόνο και παρακλήσεις. Όχι μόνο να επιστήσουμε την προσοχή της Γουινέας, αλλά να εξαρτήσουμε την παροχή ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας προς τη Γουινέα από την τήρηση των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των στοιχειωδών προτύπων και ελευθεριών. Και ο πρόεδρος της ε, Γουινέας ε, θα πρέπει να θυμηθεί πόσοι ε, ηγέτες ε, έχασαν από δημοψήφισμα την εξουσία τους. Ο κύριος Ρέντσι στην Ιταλία, ο Κάμερον ε, από το δημοψήφισμα του Brexit. Πολλοί πρωθυπουργοί έχασαν την εξουσία τους μετά τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων. Αυτό θα πρέπει να είναι επιχείρημα που θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε στις συνομιλίες με τον πρόεδρο της Γουινέας. Ο κύριος Βιγιανόεβα Ρουΐς, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Η κυρία Βιγιανόεβα Ρουΐς. Η διαμαρτυρία δεν είναι έγκλημα, είναι ανθρώπινο δικαίωμα και πολιτικό δικαίωμα. Η θεμητή αντίδραση των πολιτών που θέλουν να, να έχουν τον έλεγχο του πεπρωμένου Παρ' όλα αυτά βλέπουμε μια γενικευμένη παλιδρόμηση στα αστικά και πολιτικά δικαιώματα στον κόσμο. Γίνεται καταστολή των διαμαρτυριών. Το βλέπουμε και στη Χιλή, το βλέπουμε και στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στην Ασία. Σήμερα μιλούμε για τη Γουινέα. Έχουμε μαζικέ διαδηλώσει εκεί που ζητούν από τον πρόεδρο Κοντέ να μην υπερβεί το συνταγματικό όριο των δύο διαδοχικών προεδρικών θητιών. Επίση, ε, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μα προ του διαδηλωτέ. Έχουμε εκκλήσεις ε, των Οργανισμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ε, των Οργανωμένων Εθνών και των Αφρικανικών χωρών. Θα πρέπει να γίνουν σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ε, στοιχειώδεις και θεμελιώδει ελευθερίε. Θα πρέπει να απελευθερωθούν οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί κρατούμενοι, οι εκτιμιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη μια, υπερασπίζει τα τα ανθρώπινα δικαιώματα και από την άλλη πουλά όπλα στη Γουινέα. Και δεν αναλαμβάνουμε δράσεις ώστε οι πολυεθνικές μας να, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και δεν θα πρέπει να εργαλειοποιούμε τη διαχείριση του ελέγχου των εξωτερικών συνέρων, ούτε να παραμελούμε ή να ψηφούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε εμπορικές συμφωνίες όπως η συμφωνία με το Κοτόνου Ευχαριστώ. Ο κύριος Λέγκα για δύο λεπτά. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αυτοί που θα χρειαστεί να αλλάξουν το Σύνταγμα για να παραμείνουν στην εξουσία, κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να σκεφτούν να αλλάξουν την καριέρα του. Γιατί ε, αυτό ισχύει για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, φαντάζομαι, αλλά και για τον κύριο Κοντέ. Και αυτό, φίλοι μου, δεν είναι το μόνο που έχουν κοινό αυτοί οι δύο πρόεδροι πέρα από την, το ταλέντε τους για να καταπνίγουν τις φωνές και τις ανησυχίες των πολιτών, να τους βάζουν να βάζουν δημοσιογράφους στη φυλακή και να διώκουν τους αντιπάλους ε, της αντιπολίτευσης που ασκούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα, να... ο Πούτιν και Κοντέ είναι στην στον ίδια μοίρα. Η Γουινέα, ωστόσο, έχει κάτι που θέλει η Ρωσία έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή αλουμινίου εκτός Κίνας. 27% προέρχεται οι εισαγωγή στη Ρωσία από τη Γουινέα και αυτό καταστά ιδιαίτερα σημαντική την Γουινέα. Δεν είναι λοιπόν η έκπληξη το γεγονός ότι ο πρώην πρέσβης της ε, Ρωσίας στη Γουινέα υποστήριξε ανοιχτά τις ξεδιάτροπες προσπάθειες του Πρόεδρου να παραμείνει στην εξουσία. Από το 2002, 11 ηγέτες της Αφρικής έχουν λάβει τέτοια μέτρα για να παρατείνουν την εξουσία τους και ο Αλφα Κοντέ είναι ο δεδέκατος στην λίστα αυτή, η οποία δεν είναι και ιδιαίτερα τιμητική. Θα πρέπει κάποιος να ξέρει πότε είναι η ώρα να κάνει πίσω, να αφήσει την εξουσία, γιατί ο λαός της Γουινέας ε, τους αξίζει δημοκρατία και το Σύνταγμα για το οποίο έχουν τόσο σκληρά αγωνιστεί. Ο λαό τη Γουινέας θεωρεί ότι του αξίζει κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ότιον για ένα μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Ο πρόεδρο Αλφα Κοντέ ήταν κάποτε η ελπίδα για τη δημοκρατία στη Γουινέα. Σήμερα γίνεται αναβολή των κοινοβουλευτικών ε, εκλογών, από τραποποίηση του συντάγματο για να ξαναπάρει την εξουσία για τρίτη θετία, αγαπητοί συνάδελφοι. Αλλά αυτό που είναι ακόμα χειρότερο είναι ότι οι διαδηλώσει καταπνίγονται, διαδηλώσει οι οποίε προκύπτουν ακριβώ επειδή προτείνεται αυτή η αλλαγή, η τραποποίηση του συντάγματο. Άνθρωποι που λένε ότι δεν συμφωνούμε, θέλουμε να γίνουν δημοκρατικέ εκλογέ όπω προβλέπεται από το Σύνταγμα. Αλλά η κυβέρνηση καταπνίγει τι ε, διαμαρτυρίε αυτέ, τι διαδηλώσει αυτέ συλλαμβάνει τους ε, εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιτρέψουμε να γίνει περαιτέρω κλιμάκωση. Αυτό που περιμένουμε από την κυβέρνηση είναι να τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πολιτικά δικαιώματα και κυρίως να απελευθερωθούν άμεσα οι κρατούμενοι, οι πολιτικοί κρατούμενοι και να διατηρηθεί να υπάρχει εγγύηση του δικαιώματος διαδήλωσης και το καλύτερο θα ήταν να μπορέσουν να εκφράσουν την απόψη τους οι άνθρωποι αυτοί μέσω της δημοκρατικών εκλογών, γιατί αυτό αξίζει στην ε, Γουινέα. Θα πρέπει λοιπόν να μην υπάρξει υπερτερό αναβολή των εκλογών και το εγχείρημα για την τροποποίηση του συντάγματος δεν πρέπει να ευδοκιμήσει και ο Αλφα Κόντε θα πρέπει να κάνει πίσω και η δημοκρατία θα πρέπει να μιλήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ τώρα για το ΕΛΚ. Ο κύριος Κέλλη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν εκλέχτηκε ο Αλφακόντα το 2010, θεωρήσαμε ότι γεννήθηκε μια νέα δημοκρατική δύναμη στην Γουινέα. Όταν όμω ε, ανέβηκε τελικά στην εξουσία, όπω και πολλοί άλλοι, θέλησε να την κρατήσει για τον εαυτό του. Και αυτό προφανώ είναι σκληρό για το λαό τη Γουινέας που έχει βγει στου δρόμου και διαδηλώνει. Και το ίδιο και για την αντιπολίτευση. Τώρα λοιπόν θέλει να τροποποιήσει και το Σύνταγμα προκειμένου να παραμείνει για περαιτέρω χρονικό διάστημα στην εξουσία. Δεν προκαλεί λοιπόν έκπληξη το γεγονό ότι έχουν ξεσπάσει διαμαρτυρίε. Και πάλι αντιδρά σκληρά ε, με εκτελέσει, τραυματισμού. Είναι σημαντικό λοιπόν να τα συζητήσουμε αυτά σήμερα και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να στηρίσει ο Αλφα Κόντε το Σύνταγμα έχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριο Σορίνιο για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σίγουρα αντιδημοκρατικοί άνεμοι πνέουν στην Γουινέα Κόνακρη και εδώ και 10 χρόνια ο πρόεδρος Κοντέ ετοιμάζεται για συνταγματική μεταρρύθμιση σηκωμένη και ραμμένη στα μέτρα του προκειμένου να ανανεώσει για τρίτη φορά την προεδρική του θητεία. Ε, μάλιστα η δημιουργήθηκαν και ένα των βουλευτικών εκλογών πολλές διαμαρτυρίες με βία καταστολή, ε, εκατοντάδες ε, τραυματίες και πάνω από 20 ε, νεκρούς. Και μάλιστα είχαμε περιορισμό των θεμελιωδών ελευθεριών, της ελευθερίας έκφρασης, της ελευθερίας του συνέρχεστη που κατα... κατεστάλλει από τις δυνάμεις ασφαλείας. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κοβάσα θα πρέπει να ε, προσπαθήσουν να αναχαιτήσουν αυτή την ε, κλιμάκωση της βίας και να ζητήσουν διεξαγωγή δίκαιων και ελεύθερων βουλευτικών εκλογών. Γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία της Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων στο δημοκρατικό αυτό των εκλογών. Επίσης, καλές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες ε, είναι απαραίτητες. Και σίγουρα αυτή η κατάχρηση εξουσία ε, που πραγματοποιεί ο Κοντέ επιδεινώνει το βιωτικό επίπεδο του πληθυσμού της Γουινέα. Θα πρέπει να επαγρυπνούμε και εμείς και η διεθνή κοινότητα γιατί βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή καμπής για το μέλλον της Γουινέας Κόνακρη. Ο κύριος Μπέρικ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Εκτός μικροφώνου όμω. Κυρία Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Μου προκαλεί κάποια έκπληξη το γεγονό ότι η Δημοκρατία τη Γουινέα αποτελεί αντικείμενο αυτή τη συζήτηση στα κατεπήγοντα. Όλοι γνωρίζουμε ε, ότι οι διαδηλώσει ε, είναι βίαιε στη χώρα αυτή, αλλά υπάρχουν πολλέ εικασίε ε, στο ψήφισμα αυτό. Ακόμα και το Συμβούλιο, το οποίο ενημερώθηκε από την Διεθνή Αμνηστία είναι προσεκτικό στις δηλώσεις τους και πραγματικά μιλάμε για βίαιες διαδηλώσεις λοιπόν κατά της κυβέρνησης επίσης. Δεν προκαλεί λοιπόν έκπληξη το γεγονό όταν ε, αντιδράσεις, οι αντιδράσει είναι επίση ε, βίαιε. Ο πρόεδρο Κοντέ ήταν ο πρώτο δημοκρατικά εκλεγμένο ε, πρόεδρο τη Δημοκρατία τη Γουινέα και δήλωσε ότι ήθελε να τροποποιήσει και το Σύνταγμα γιατί αποτελούσε ένα υπόλοιμα της απεικιοκρατίας. Αυτό δεν αποτελεί δικτατορία. Προσφέρει δημοψήφισμα, προγραμματίζονται εκλογές οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στους ε, εκλογείς να αποφανθούν για το μέλλον της χώρας τους οι ίδιοι. Ένα από τα προβλήματα λοιπόν είναι το γεγονό ότι κάποια κόμματα τη αντιπολίτευση ε, όχι μόνο απειλούν ότι θα εμποκοτάρουν τι εκλογέ, αλλά ότι δεν θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή εκλογών και Α, αντί για τη διπλωματία αυτή, λοιπόν, την υποπτήφεται διπλωματία την οποία ασκούμε σε αυτέ τι συζητήσει για τα καταπήγοντα, θα μπορούσαμε συγκεκριμένη βοήθεια να δώσουμε στου ανθρώπου τη Νέα Γουινέα. Θα μπορέσουν, λοιπόν, ε, οι άνθρωποι, ο λαό τη Νέα Γουινέα να αποφανθούν κατά πόσο επιθυμούν την τροποποίησή του συντάγματο. Δεν έχει νόημα λοιπόν να κάνουμε δηλώσει για πράγματα τα οποία δεν μα αφορούν και τα οποία μόνο να επιδεινώσουν μπορούν την κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Καστάλτο λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το 2019 ήταν μια χρονιά που βιώσαμε ένα κύμα διαμαρτυριών σε όλους τους χρόνους του κόσμου για πολύ διαφορετικές χώρες μεταξύ τους σε διαφορετικό επίπεδο και πλούτου και ευημερίε. Και η Γουινέα Κονάκρη είναι μια πόλη η οποία ζητά όλο και περισσότερη, μια χώρα συγγνώμη, η οποία ζητά όλο και περισσότερη συμμετοχική δημοκρατία. Υπήρξαν διαμαρτυρίε κατά τη άδικη συνταγματική μεταρρύθμισης του Προέδρου Αλφακοντέ ε, Διαμαρτυρίε ε, και είχαμε και πράξει βίε και από του διαδηλωτέ, αλλά κυρίω από τι δυνάμει ασφαλεία. Ε, είδαμε ότι όπως πολύ συχνά συμβαίνει η απάντηση των αρχών ε, η οποία αμφισβητείται είναι απλώς ε, καταστολή της βίας και περιορισμός των θεμελιωδών ελευθεριών. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ ανησυχητική, συνάδελφοι, και εμεί θα πρέπει να παρακολουθούμε και να είμαστε σε εγρήγορση για τα όσα συμβαίνουν και να απαιτήσουμε να υπάρξει διάλογο με όλα τα κοινωνικά ε, στρώματα και να αποφύγουμε και εμφύλιο πόλεμο, αλλά κυρίω πρέπει να ζητήσουμε από τι επιχειρήσει μα να σταματήσουν να εξάγουν όπλα σε χώρε όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά του λαού και κατά τη κοινή γνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριανή τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η εποχή της γαλλικής επιρροής ε, στην Αφρική αρχίζει να αποπακρίνεται. Ε, πλέον η Γουινέα Κονάκρη ε, επιδίδει, επιδίδει σε μια διαδικασία χειραφέτησης από την γαλλική απεικιοκρατία και προσπαθούμε να δούμε και τι έγινε από το κράτος στις διάφορες πτυχές της κοινωνίας της Γουινέα. Η Γουινέα Κονάκρη είναι μια χώρα στην οποία υπάρχουν πάρα πολύ ισχυρές εξωτερικές παρεμβάσεις αποφάσεις οι οποίες δεν της επιτρέπουν να προχωρήσει. Υπάρχει και η ε, ε, αντίσταση στο δημοψήφισμα στη χώρα. Η χώρα μπορεί να αποφασίσει ελεύθερα αν θέλει να αλλάξει το σύνταγμά της αν αυτό επιθυμεί. Σήμερα ο πρόεδρος Αλφα Κοντέ ε, ε έχει πολλές επικρίσεις από την, ε, ε, για τη συμπεριφορά του, για την καταστολή και τα όσα κάνει για τη δημόσια τάξη. Ναι, ε, τα επεισόδια αυτά της καταστολής είναι απαράδεκτα, αλλά κάποια πράγματα τα οποία γίνονται και έξω δεν είναι και αυτά απαράδεκτα. Εμείς θα πρέπει να σταματήσουμε, αν θέλουμε να έχουμε επιρροή στην Αφρική, για να δούμε και τι γίνεται και από την Κίνα, την Ινδία και άλλες χώρες. Από το 2000 έχουμε πάνω από 100 ε, χώρε οι οποίε αποφάσισαν να αλλάξουν το σύνταγμά του, ε, γιατί οι φύνοντε θέλαν να παρατείνουν την εξουσία του. Το, το ίδιο έγινε και στο Καμερούν που έχουμε τον ίδιο ηγέτη εδώ και 30 χρόνια. Εάν θέλουμε πραγματικά να διαδραματίσουμε κάποιο ρόλο, θα πρέπει να υπάρχει και ένα δημοψήφισμα το οποίο θα δώσει στο λαό τη Γουινέα τη δυνατότητα να επιλέξει ή να απορρίψει αυτή τη σταγματική αναθεώρηση και θα πρέπει να φροντίσουμε να γίνει νόμιμο αυτό το δημοψήφισμα με ειλικρίνεια και από εκεί και πέρα οι πολίτες της Γουινέας Κονάκρη θα επιλέξουν το σύνταγμά του. Ξεκινάμε τώρα τη διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε όμως και ψηφοφορία εντός ολίγου και έχουμε και άλλη μια συζήτηση. Υπάρχουν έξι άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ακούσω έναν από κάθε πολιτική ομάδα. Από το ΕΛΚ, ο κύριος ε, Τζεχόφσκι, για το SND ο κύριος Λόπε Αγγιλάρ και από την ΚΟΕ ο κύριος ε, Γόλης. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Τζεχόφσκι. Σας ευχαριστώ. Κυρία Υπάρχουν λοιπόν τα ερωτήματα αυτά. Γιατί θέλουμε να διακυβεύσουμε αυτή τη συζήτηση, θέλουμε να έχουμε επιρροή στην Αφρική. Θέλουμε η Αφρική να γνωρίσει τη δημοκρατική αυτή πορεία από, τον, από την απεικιοκρατία στην δική δημοκρατία. Εγώ ήμουν ιδιαίτερα ευτυχή όταν το 2010 ξεκίνησε με την προεδρική τη θητεία ο πρόεδρο ε, Κοντέ. Παρακολούθησα την πορεία του και την πολιτική του με προσοχή. Έδειξε το απαραίτητο ενδιαφέρον και διαπίστωσα ότι η πολιτική κατάσταση σε αυτή την πολύ όμορφη και πλούσια χώρα άλλαξε. Άλλαξε σταδιακά. Σήμερα λοιπόν Μένω έκπληκτό παρακολουθώντα τα τεκτενόμενα στη χώρα από τον Οκτώβριο και μετά. Δεν είναι φυσιολογικό να εκτελείται κόσμο στου δρόμου από δυνάμει ασφαλεία οι οποίε ε, αντεδρούν τόσο βία κατά του λαού. Να μην υπάρχει πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και σε τέτοιε άλλε υπηρεσίε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει το χέρι μα για να ξεπεράσουμε αυτό. Οι ε, ηγέτες Αφρική, της Αφρικής που ναι μεν εξελέγησαν δημοκρατικά αλλά στη συνέχεια έκαναν κάποιες χαραγωγήσεις για να επανακλεγούν, να αναθεωρήσουν τα συντάγματά τους και να διοργανώσουν ψευδοδημοψηφίσματα για να παρατείνουν επαόριστον ε, την ε, παραμονή του στην εξουσία. Δυστυχώς είναι η ελισίδα που εξηγεί την αστάθεια, την καταστολή, την οδύνη ε, και τα δεινά των πληθυσμών των λαών της Αφρικής. Είχαμε πραγματικά παροξισμό το 2009 και τη σφαγή, 200.000 ε, νεκρούς, ε, βιασμούς γυναικών ε, και δυστυχώς ακόμη και ενέτειο 2020 συνεχίζονται τέτοιες βιοπραγίες. Θα πρέπει λοιπόν στη ρίζα του να χτυπήσουμε το κακό, να αποφευχθούν ε, τέτοιες, ε, τέτοια έκτροπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί μερικές φορές ε, φτάνουν κάποια λόγω δράσεων των λαθροδιακινητών σε χώρε νομίζω ότι είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνουν ακόμα και στα νησιά τα Κανάρια χωρίς να αντιμετωπίζουν, χωρίς να έχουν συνείδηση τι θα ακολουθήσει. Θα πρέπει επιτέλου να δράσουμε. Κύριο Γουάλλα. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ψήφισμα καταδικάζει τι συνεχεί βιοπραγίε στην δημοκρατία τη Γουινέα και τι καταστρατηγήσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εγώ καταδικάζω την ε, παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων παντού. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όμως ε, χαίρεται να καταδικάζει τέτοια, τέτοια παραβίαση όταν γίνεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από το Νοέμβριο του 2018 η Γαλλική Αστυνομία συστηματικά καταπιέζει τους διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για τις συναφιλελεύθερες ε, ε, μεταρρυθμίσεις του Μακρόν, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και άλλα μέσα. Και Είχαμε πολλούς τραυματίες, δύο νεκρούς, πολλές, ε, πολλούς τραυματισμούς ε, κρανίου. Πέντε άνθρωποι έχασαν το χέρι τους, άλλοι έχασαν την όρασή τους. Και αυτό δεν το καταδικάζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά στρουθοκαμιλίζουμε όταν έχουμε καταστρατηγήσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός ε, της Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν ζητούμε από την Ισπανία να αντιμετωπίσει του καταλανούς διαδηλωτέ με δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Και ολοκληρώνω τη συζήτηση με τη δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο, κύριε Ντάλη. Uh, Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επιμακρόν εταίρος της Γουινέας Κονάκρη που έχει κάνει τεράστια πρόεδρο από τις πρώτες δημοκρατικές εκλογές το 2010 που έφεραν στην εξουσία τον ε, ε, αυτή τη στιγμή πρόεδρο, τον κύριο Κοντέ. Η σταθερότητα και η ευημερία της χώρας είναι πολύ σημαντική για την περιοχή, όπως είναι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το Φεβρουάριο του 2018, που είχαμε τοπικές εκλογές, η κοινωνική και πολιτική κατάσταση έχει ε, γίνει ιδιαίτερα τεταμένη. Η προοπτική ενός νέου συντάγματος που θα επιτρέψει στον ε, πρόεδρο Κοντέ να παραμείνει στην εξουσία πέραν ε, του τέλους της δεύτερης και τελευταίας θητείας του ένωσε τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης σε ένα εθνικό μέτωπο για την υπεράσπιση του συντάγματος και οδήγησε και σε πολύ συχνές διαδηλώσει κατά τη τρίτη θετίας του Προέδρου. Οι διαμαρτυρίε αυτέ ε, ε, πολύ συχνά ε, διαλύονταν από δυνάμεις ασφαλείας, ε, είχαμε κράτηση διαδηλωτών και υπάρχουν πολύ σημαντικές ελευθερίες, όπως για παράδειγμα η ελευθερία της έκφρασης, η οποία δεν έγινε σεβαστή. Από τον Οκτάβριο του 2019 περίπου 30 άτομα έχασαν τη ζωή τους ε, και θεωρείται ότι έχουν σκοτωθεί από πειρά δυνάμεων ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει επανειλημμένως μια κατάλληλη διεξαγωγή έρευνες για να δούμε ε, υπό ποιε συνθήκε ε, συνέβησαν αυτά τα γεγονότα και ε, για να βρεθούν ενώπιον του δικαστηρίου οι υπεύθυνοι. Η προετοιμασία για τι νομοθετικέ εκλογέ, οι οποίε θα γίνουν στην 1 του μορτίου, οδήγησε σε περισσότερε εντάσει. Όσον αφορά τις αμφιβολίες για την αξιοπιστία των εκλογικών καταλόγων, δύο πολιτικά κόμματα είπαν ότι θα μποϊκοτάρουν τις εκλογές. Το 2015 και το 2008 οι Επιτροπές Εκλογών ε, σύστησαν περαιτέρω αναθεώρηση του εκλογικού νόμου, ο οποίος δεν αντανακλούσε ε, σωστά το εκλογικό σώμα δεν έγινε η αναθεώρηση, έγινε παρά μόνο σε μερικά τμήματα. Οι πρόσφατες λοιπόν εκλογές ε, θα συνδυαστούν με ένα δημοψήφισμα για ένα νέο σχέδιο ψηφίσματος το οποίο επιβλήθη το Δεκέμβριο, το οποίο Σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα ε, να ε, προχωρήσουν οι προθέσεις του κυρίου Κοντέ. Και αυτό οδήγησε σε περαιτέρω διχασμό της χώρας. Υπάρχει συνεχιζόμενη λοιπόν αστάθεια και πόλωση και φυσικά ε, υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία είναι εθνοτικής φύσεως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συστηματικά με τους τοπικούς εταίρους και με το Ηνωμένα Έθνη, την Αφρικανική Ένωση, την Οικονομική Ένωση των Δυτικοαφρικανικών Κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία έχουν ζητήσει να υπάρξει ηρεμία και έχει διευκολύνει και το διάλογο μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Η εμπιστοσύνη σε ένα αξιόπαστο και διάφανο εκλογικό σύστημα και διαδικασία είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη να εξασφαλίσουμε συμμετοχή και αποδοχή του αποτελέσματος. Κάθε χώρα έχει το δικαίωμα φυσικά να τροποποιήσει, να εξυγχρονίσει το, σύστημα, το σύνταγμά τη, αλλά η αλλαγή του θεμελιώδους αυτού νόμου, του συντάγματο, θα πρέπει να είναι αντικείμενο ευρεία διαβούλευση που θα οδηγήσει και σε ευρεία συνένεση. Κάτι το οποίο δεν έχουμε σήμερα. Ένα δημοψήφισμα λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές δεν συνάδει με τις καλές πρακτικές ε, που συστήνει η Αφρικανική Ένωση ε, και η ΕΚΟΕΝΤΣ. Επίσης, ε, η Δυτικοαφρικανική Ένωση έχει κερδίσει ακριβώς τα δημοκρατικά της εύσημα βασιζόμενη σε αυτές τις συνθήκες. Και ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο ο εκπρόσωπο του υπάτου εκπροσώπου του κ. Μπορέλ την περασμένη Παρασκευή ζήτησε να γίνει ένα διάλογο, στον οποίο θα συμμετέχουν όλοι, για να αποφύγουμε περαιτέρω κλιμάκωση τη βία και να εξασφαλίσουμε τι συνθήκε για διαφάνεια στι διαδικασίε, ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν και όλα ε, τα εκλογικά κόμματα στι εκλογέ. Μόνο όταν γίνεται σεβαστός ο πολιτικός χώρος ε, και σταματήσουν ε, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μπορέσουμε να έχουμε κατάλληλες συνθήκες για να υπάρξει αυτός ο διάλογος. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει όλοι οι παράγοντες ε, να θέσουν την ενότητα και την ειρήνη της Γουινέας στην πρώτη γραμμή. Να συνεχίσουν λοιπόν να συμβάλλουν στην όλη διαδικασία. Εμεί θα συνεργαστούμε με του εταίρους μα, τα Ηνωμένα Έθνη, την Αφρικανική Ένωση και την ΕΚΟΑΣ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται στεναρά για την Γουινέα Κόνακρη ε, σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τους υπερασπιστές ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά υποστηρίζουμε την ανθεκτικότητα ε, του λαού και θα πρέπει η κρίση στη Γουινέα Κόνακρη να είναι στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας. Ευχαριστώ και ολοκληρώθηκε η συζήτηση αυτή. Υποβλήθηκαν έξι ψηφίσματα και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σήμερα. Η επόμενη συζήτηση, το επόμενο θέμα, έχει να κάνει με την παιδική εργασία στα ορυχεία της Μαγδασκάρη. Δυστυχώς έχουμε καθυστερήσει ιδιαίτερως σήμερα και γι' αυτό λοιπόν θα σας παρακαλούσα να μην χρησιμοποιήσουμε μπλε κάρτες. Δεν μπορώ να σα επιτρέψω στη συζήτηση αυτή. Ο συνάδελφος ο κ. Μπίλτε έχει το λόγο, ο οποίο είναι και ο Συγγραφέα ε, τη ε, ο εισηγητή. Ή συνάδελφο, διορθώνει πρόεδρο. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Η συναδελφο διορθωνει πρόεδρο. ευχαριστω είναι 13 χρονών και δεν πρόκειται να ξαναπάει σχολείο. Για 20 ε, σέντ την ημέρα δουλεύει στα ορυχεία, στο Μελγάς. Και ο Φρεντερικ, 8 χρονών, ο οποίος δουλεύει στα ορυχεία Μαρμαριγία και είναι μόνο λίγα από τα 73.000 παιδιά τα οποία εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες με παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είναι δύσκολο λοιπόν να κατηγορήσουμε την χώρα αυτή που αναγνωρίστηκε ότι έκανε προσπάθειες το 2016 από, την, από τις ΕΠΑ. Γιατί 87% του εξαγωγών μαρμαριγία πήγαιναν στην Κίνα για να εξοπλίσουν την ηλεκτρονική βιομηχανία. Τα παιδιά αυτά βρίσκονται σε φρικτή η κοινωνική κατάσταση και αυτό αποτελεί όνειδος για την ανθρωπότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η συνάδελφος κυρία Ροζ για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι, αγαπητοί Πρόεδρε, βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στο Κοινοβούλιο για να πούμε ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παιδική εργασία στη Μακαδασκάρη, γιατί είναι μια κατάσταση απαράδεκτη, η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η πρόεδρο τη Επιτροπή, Ursula von der εξήγηλε μια πολιτική μηδενική ανοχή τη παιδική εργασία, αλλά θα ήταν υποκριτικό να θεωρήσουμε ότι έχουμε χρησιμοποιήσει επαρκώ τι δυνάμει μα προ την κατεύθυνση αυτή. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν το θέμα των δικαιωμάτων των παιδιών σε ό,τι αφορά τις ε, συγκεκριμένες ε, υποχρεώσει που συνεπάγεται σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επίση, να κοιτάξουμε την ευθύνη των εταιριών. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά τα στοιχεία αυτά. Θα πρέπει να, επι... να ελέγχουν τη διαδικασία εφοδιασμού σύμφωνα με τι ε, διαδικασίε που προβλέπει ο ΩΣΑ. Και όλα αυτά θα πρέπει να κοιτάξουμε στο πολυεθνικό επίπεδο. Το Συμβούλιο θα πρέπει να δώσει εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προχωρήσει σε ό,τι αφορά τη σύναψη τη ε, σύμβαση αυτή και να είναι γρήγορη η έγκριση τη. Αναμένουμε μια δυναμική απάντηση από πλευρά ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό, η κυρία Ίντσιρ. Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Φανταστείτε το τηλέφωνό σα ή το αυτοκίνητό σα να κατασκευάζονταν μόνο εις βάρος ε, άλλων ανθρώπινων ε, ζώων. Χιλιάδες ε, παιδιά απασχολούνται στα ορυχεία της Μαδαγασκάρης και από εκεί προέρχονται ανταλλακτικά υλικά που χρησιμοποιούνται για να φτιαχτούν τα κινητά μας και τα αυτοκίνητά μας εις βάρος της παιδικής ζωής. Τα παιδιά θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο και όχι στα ορυχεία. Θα πρέπει να μορφωθούν, να μπορέσουν να υλοποιήσουν αργότερα τα όνειρά του. Το σύνολο τη κοινωνία, ο ιδιωτικό τομέα αλλά και η διεθνή κοινότητα φέρουν ευθύνη για την κατάσταση αυτή. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη ρίζα του προβλήματο που είναι μεταξύ άλλων και η φτώχεια και γι' αυτό θα πρέπει να υιοθετήσουμε διορθωτικά μέτρα. Και οι ευρωπαϊκέ εταιρείε θα πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνε του καθ' όλη τη διάρκεια της αλυσίδα αξία και του ανεφοδιασμού σε τέτοια ορυκτά και μεταλλεύματα. Δεν μπορούμε να ψηφούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των παιδιών και ελευθερίε των παιδιών. Είναι αδιαπραγμάτευτα αυτά τα δικαιώματα και οι ελευθερίε. Θα πρέπει να γίνουν σεβαστά οπωσδήποτε. Και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να δούμε πώ θα ε, φροντίσουμε του πιο ευάλωτου ε, συμπολίτε μα, που είναι τα παιδιά στην κοινωνία μα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τσαρνέτσκι για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, πολύ σπάνια στην πολιτική έχουμε τόσο ξεκάθαρη κατάσταση, ε, τόσο ασπρόμαυρη κατάσταση που δεν έχει καμία δικαιολόγηση, καμία αιτιολόγηση, καμία εξήγηση που να επιτρέπει, που να δικαιολογεί μια τέτοια κατάσταση. Όλοι έχουμε παιδιά, έχουμε εγγόνια και θυμόμαστε ε, παιδιά στην εφηβεία ή και νεότερα ε, και θεωρούμε διανόητο να εργάζονται τα παιδιά σε τέτοια ηλικία. Και γι' αυτό θα πρέπει να μην φυστούμε προσπαθειών ε, και να υψώσουμε στεναρά τη φωνή μας, τη φωνή μας τη ηθικής αντίθεσης, αλλά και πολιτικής αντίδρασης και άσκησης πίεσης προς τη Μαδαγασκάρη και σε άλλες χώρες, ε, γιατί είναι αδιανόητη και απαράδεκτη αυτή η κατάσταση. Να βοηθήσουμε με ανθρωπιστικά κονδύλια, με οικονομική βοήθεια τις χώρες αυτές, αλλά να σταματήσει αυτή η πρακτική. Ο κύριος Σόλτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ενώ εμείς μιλάμε 11.000 ε, ε, παιδιά απασχολούνται σε ορυχεία μαρμαριών ε, στη Μαδαγασκάρη. Μερικά είναι και παιδιά 5 ετών και εργάζονται σε επικίνδυνες συνθήκες μόνο για να εξασφαλίσουν το παστοζίν για τις οικογένειές τους. Πόσο θα αγνοούμε τη μοίρα αυτών των παιδιών που συμμετέχουν σε εξορίξεις μαρμαριών στα ορυχεία της Μαδαγασκάρης για τις δικές μας ευρωπαϊκές εταιρείες η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η θα πρέπει να αναλάβουν ε, ευθύνε και να προβλέψουν ένα νομικό πλαίσιο ώστε οι εταιρείε μας να ανεφοδιάζονται με ηθικό και δοντολογικό τρόπο με τέτοια ε, ορυκτά και υλικά. Και όπως είπαμε θέλουμε μηδενική ανοχή για την ε, παιδική εργασία και αυτό το στόχο μας να τον υλοποιήσουμε. Επίσης θα πρέπει να θεωρούμε το ηθικό εμπόριο προϊόντων και να υλοποιήσουμε του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ. Και γι' αυτό απευθύνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο και με την Κίνα και άλλου σημαντικού εισαγωγεί μαρμαριγιών και διάλογο με την κυβέρνηση τη Μαδαγασκάρη για να σταματήσει η εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας ε, το συντομότερο δυνατό και δυνατό μέχρι το 2030 στη Μαδαγασκάρη. Η κυρία Ζόφκο, για 1,5 λεπτό. Στο ψήφισμά μας καταδικάζουμε απερίφαστα την απαράδεκτη χρήση παιδική εργασία ε, πάση μορφής και ζητούμε από τις αρχέ της Μαδαγασκάρης να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ε, να εγγυηθούν τα δικαιώματα των παιδιών, την ασφάλεια και την ακαιρεότητά τους. Πολλά παιδιά απασχολούνται σε ορυχεία μαρμαριγιών και η αύξηση αυτή τη εκμετάλλευση του ε, συνδυάζεται με τη μείωση της τιμής της πρώτης ύλης, κάτι που ενίσχυσε την ε, παιδική εργασία. Είναι επικίνδυνες και άθλιες συνθήκες στα ορυχεία, απειλούν τη ζωή και την υγεία των παιδιών. Ε, είναι εκτεθειμένα χρόνια σε αναπνευστικά προβλήματα, σε σοβαρές ασθένειες και αντιμετωπίζουν και ψυχολογική και σωματική εκμετάλλευση. Η εξάλληψη της φτώχειας είναι η μόνη προϋπόθεση για την κατάργηση και της παιδικής εργασίας. Θέλουμε συγκεκριμένα μέτρα σε τομείς όπως η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η επασχόληση. Η Μαδαγασκάρη υιοθέτησε νομοσχέδια και διατάξεις για τον περιορισμό της παιδικής εργασίας και αύξησε το νόμιμο όριο ηλικίας από τα 15 στα 16 για την, για την εργασία. Βέβαια, ζητούμε από τι αρχέ και την κυβέρνηση να δώσουν προτεραιότητα στην τήρηση των διεθνών υποχρεώσεών του, ε, συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και να σεβαστεί τα ανθρώπινα και παιδικά δικαιώματα. Δυστυχώ, μέχρι στιγμή οι αρχέ τη Μαδαγασκάρη δεν επέβαλαν κυρώσει λόγω έλλειψης σπόρων για κατάλληλο έλεγχο και πλήρη ε, συμμόρφωση με την υπάρχουσα νομοθεσία. Θα πρέπει όμως και εμείς να αναλάβουμε το ρόλο μας και με το ψήφισμά μας ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την ε, πρόθεση ε, πρωτοβουλειών και σχεδίων ώστε να καταπολεμηθεί η παιδική εργασία στη Μαδαγασκάρη. Έχουμε ταχθεί αναφαδόν υπέρ της καταπολέμησης της παιδικής εργασίας με την εμπορική μας πολιτική και άλλωστε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε για μηδενική ανοχή στην παιδική εργασία στην εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Κύριε Πρόεδρε, κανείς και σίγουρα κανένα παιδί δεν αξίζει να εργάζεται σε επικίνδυνες ε, ε, και απειλητικές για τη ζωή του συνθήκες. Σίγουρα η προστασία των παιδιών είναι βασικό στοιχείο της πολιτικής μας προσέγγισης. Και με το ψήφισμά μας νομίζω ότι στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα προς τον κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενη μιλήτρια η κυρία Βάτμανς, για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επιτροπέ, συνάδελφοι. Όλοι γνωρίζουμε τι εικόνε, τι έχουμε δει. Παιδιά σε ορυχεία, εγώ τις, έχω δει τις εικόνες αυτές με τα ίδια μου τα μάτια. Τα παιδιά στη σειρά, στοιχισμένα από τα πιο κοντά προς τα πιο ψηλά, μικρά προς μεγάλα. Λες και είναι στο σχολείο, αλλά πηγαίνουν στα ορυχεία για να δούμε ποιοι είναι οι πιο μικροί, για να μπορέσουν να μπουν μέσα στα στενά, τα τρομακτικά, τα σκοτεινά τούνελ. Συνάδελφοι, όταν έχει δει κανεί τέτοιες εικόνες το βάζει ω προτεραιότητά του να έχει καταργήσει την παιδική εργασία μέχρι το 2025. Και κοιτώντα τα αριθμητικά στοιχεία, μιλάμε για 152 εκατομμύρια ε, παιδιά τα οποία ξαναγκάζονται να δουλέψουν. Ένα στα δέκα παιδιά δηλαδή στον κόσμο πηγαίνει να δουλέψει αντί να παίζει, αντί να πάει στο σχολείο. Και συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σας γιατί ήταν δύσκολες διαπραγματεύσεις, να το πούμε. Ήταν πραγματικά πολύ χρειάστηκε πολύ εξουσία και εξουσία από τις γυναίκες. Αλλά ήταν τελικά πολύ δυναμικό το ψήφισμα σε ό,τι αφορά τα 11.000 παιδιά αυτά τα οποία εργάζονται στα αρχεία Μαρμαριά. Να βοηθήσουμε λοιπόν τα παιδιά αυτά, γιατί ένα στα δύο παιδιά στο Μαγδασκάρι εργάζονται, αλλά να λάβουμε και απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζήτω από την ε, Επιτροπή και από την Ursula von der Leyen, την οποία υποστηρίζω ένθερμα, να το βάλει αυτό ως προτεραιότητα. Πριν τις θερινές διακοπές να καταθέσετε ένα σχέδιο δράσης από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να έχουμε καταργήσει με την κυριαρχία μέχρι το 2025. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Για το ΕΛΕΚ ο συνάδελφος ο κ. Κέλλη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Πρόκειται για ένα από τα πιο λιπερά ψηφίσματα που έχουμε συζητήσει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι αφορά παιδιά και παιδική εργασία. Σε αυτή την περίπτωση, ε, στα ορυχεία μαργιών στη Μαδαγασκάρη. Αυτά τα νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα οποία ξεκινούν από την ηλικία των 5 ετών να εργάζονται στα ορυχεία και εκτιμάται ότι το 62% των ανθρακορίχων είναι, των ε, εργαζομένων στα ορυχεία είναι ε, ανήλικοι. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σχολείο και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους για το μέλλον. Ε, η υγεία τους δε, κυρίως οι πνεύμονές τους, επηρεάζεται και αυτό επηρεάζει και την ανάπτυξή τους. Επίσης δουλεύουν και για πενιχρούς μισθούς. Είναι λοιπόν δίκαιο να αναλάβουμε και εμείς την ευθύνη να ε, προωθήσουμε το τέλος αυτής της ε, παιδικής εργασίας μέχρι το 2025. Πρόκειται για ένα στόχο των επιτρόπων, τον οποίο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε. Ευχαριστώ. Για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, η κυρία Ρενά για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Είμαι πάρα πολύ εκνευρισμένη για τη συζήτηση αυτή που κάνουμε σήμερα. Συμφωνώ ότι η παιδική εργασία στη Μαδαγασκάρη είναι απαράδεκτη, αλλά αγαπητοί συνάδελφοι, όταν έπρεπε να ψηφιστεί νόμος ε, για τη δέουσα επιμέλεια, την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια των επιχειρήσεων, η δεξιά, το Ρινιού, το ΕΛΚ καταψήφισε. Όταν ε, τίθεται θέμα κεφαλαίου βιώσιμη ανάπτυξη με κυρώσει εχθέ για το Βιετνάμ, ε, ώστε να απαγορεύεται η παιδική εργασία στο Βιετνάμ, το Ρινιού και το ΕΛΚ καταψήφισε. Όταν ε, ε, πρέπει να προωθήσουμε μια συζήτηση για τις διεθνείς εμπορικές συμβάσεις ε, που θα θέτει ενώπιον των ευθυνών τους τις επιχειρήσεις, το ΡΙΝΙΟΥ και το ΕΛΚ καταψηφίζουν. Όταν έπρεπε να γίνει λότητα για τα ορυχεία, το ΕΛΚ και το ΡΙΝΙΟΥ όλοι, ένα τμήμα τους, όχι όλοι, καταψήφισαν. Αλλά το να εργαστούμε κατά της παιδικής εργασίας και να ε, ψηφίσουμε κάτι το οποίο δεν έχει καμία δέσμευση είναι υποκρισία. Θα το υποστηρίξω γιατί είναι σημαντικό, αλλά θεωρώ ότι είναι υποκριτικό από πλευράς του Κοινοβουλίου μας να έχει μια τέτοια στάση. Ευχαριστώ. Η κυρία Χαράντσοβα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. 47% των ε, παιδιών από τη Μαδαγασκάρη ετών 5 έως 15 εργάζονται αντί να πηγαίνουν σχολεία. Και δεν τους στερούμε μόνο την εκπαίδευση. Πολλά από αυτά ε, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους καθημερινά σε επικίνδυνες εργασίες όπως εργασία στα ορυχεία. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην παιδεία, έχει δικαίωμα σε ένα ε, βιωτικό επίπεδο το οποίο υποστηρίζει την ε, φυσική ε, σωματική, ε, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξή του. Η παιδική εργασία παραβιάζει αυτά τα δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να σταματήσει η παιδική εργασία μέχρι το 2025. Αυτό σημαίνει πέντε ακόμα χρόνια που εκατομμύρια παιδιά θα υποφέρουν και στη Μαδαγασκάρη και αλλού και θα χαθούν πολύ περισσότερε ζωέ και θα ε, καταστραφεί και το μέλλον του. Θα πρέπει να δοθεί ένα τέλο λοιπόν στην παιδική εργασία ακόμα νωρίτερα, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε χώρε για να επιταχύνουν την εφαρμογή τη νομοθεσία και δράσεις οι οποίες θα επιτύχουν αυτό το στόχο. Η ομάδα Renew Europe λέει ότι θα πρέπει οι δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ε, μεταφραστούν σε πιο ουσιαστικές πράξεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πυρπάκας για 1,5 λεπτό από την ε, Ταυτότητα και Δημοκρατία. κυρία Πυρμπάκα, συγγνώμη. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το ζήτημα που πραγματευόμαστε θέτει ένα αμφιβόλο το παγκόσμιο σύστημα παραγωγής που εδράζεται μόνο στην οικονομία. Η απασχόληση παιδιών για εξαγωγή ε, φθηνών προϊόντων στην Ευρώπη, αψηφώντας ε, τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες, δείχνει το φιλελεύθερο παραγωγικό μοντέλο που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και που οδηγεί σε εκμετάλλευση των παιδιών, όπως συμβαίνει στα ορυχεία της Μαδαγασκάρης. απασχολούμε παιδιά ε, είναι αυτό το οικονομικό μοντέλο που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η παιδική εργασία, το να δουλεύουν τα παιδιά, αυτό επιθυμούμε. Για την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία το μέλλον ε, βρίσκεται στον πραγμα... ρεαλιστικό τοπικισμό και όχι στην παγκοσμιοποίηση χωρίς σύνορα. Θα πρέπει να βρούμε έναν έξυπνο προστατευτισμό που θα ενημερώνει τον ε, καταναλωτή για την προέλευση προϊόντων που χρησιμοποιούν ή περιέχουν μεταλλεύματα ή ορυκτά που έχουν εξαχθεί, εξορυχθεί με τέτοιο τρόπο. Πώς είναι δυνατόν να εισάγουμε προϊόντα που παρασκευάστηκαν με την εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας. Θέλουμε έναν έξυπνο προστατευτισμό λοιπόν που θα εδράζεται στις δίκαιες εμπορικές συναλλαγές και στον τοπικό χαρακτήρα. Μια Ευρώπη που θα προστατεύει ε, τους λαούς και τα έθνη θα, δεν θα εξυπηρετεί τα κρατικά συμφέροντα, αλλά τα συμφέροντα του λαού. Ακούστε ε, τους λαούς και την ψήφο τους. Ήρθε η ώρα για δράση, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ και παρακαλώ να μην υπερβαίνετε το χρόνο αγόρευσή σας, γιατί 11 και 59 πρέπει να ολοκληρώσουμε. Χρόνο φίδου, λοιπόν. Από τους πράσινους, η κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε η ανθρώπινη και, το ανθρώπινο και περιβαλλοντικό τίμημα των σύγχρονων κινητών μας και των γελιστερών αυτοκινήτων μας είναι απαράδεκτο, γιατί το τίμημα αυτό είναι η παιδική εργασία, η καταναγκαστική εργασία, χωρίς καμία γνώση για τα καταναλωτή από πού προέρχονται όλα αυτά τα προϊόντα. Και αν το Κοινοβούλιο θέλει να παίρνει στα σοβαρά τον εαυτό του, θα πρέπει να προσέξει ε, την παραγωγή τέτοιων προϊόντων και να αποφεύγουμε να εισάγουμε προϊόντα που χρησιμοποιούν υλικά που προέρχονται από ορυχεία. Και δεν ε, αρκεί να μιλούμε μόνο για την ε, δεσμευτική δέουσα επιμέλεια που είπε η προαλλαλήσα. Θα πρέπει να το συνδυάσουμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Α μην είμαστε υποκριτέ. Θα θέλουμε να εξαλείψουμε την παιδική εργασία. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο, αλλά χρειαζόμαστε μέσα και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε υποχρεωτική νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δέουσα επιμέλεια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Κύριο Μπιέλλαν, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η παιδική εργασία στη Δημοκρατία τη Μαδαγασκάρης είναι γενικό πρόβλημα. Πάνω από 230.000 παιδιά απασχολούνται, γίνονται αντικείμενα εκμετάλλευση στα ορυχεία. Ακόμη και από τα δέκα του χρόνια παιδιά δουλεύουν στα χρυσορυχεία, στα, χρυσορυχεία, στα και στα ορυχεία Ζαφύρου. Και παρόλα αυτά ζουν ε, σε μεγάλη φτώχεια και πάσχουν από αναπνευστικά προβλήματα και αρρώστιε όπω η ελονοσία, ενώ εξαναγκάζονται σε εργασία υπό επικίνδυνε ε, συνθήκε. Και παρόλο που οι αρχέ τη Μαδαγασκάρης ε, ρύθμισαν νομοθετικά το θέμα τη εργασία των παιδιών άνω των 15 ετών. δυστυχώ η ευέλικη εφαρμογή του νόμου αυτού είναι ανεπαρκή. Ζητούμε λοιπόν από τι αρχέ τη Μαδαγασκάρης να σεβαστεί τα δικαιώματα των παιδιών, να εγγυηθεί την ασφάλεια και την κατάλληλη παιδεία του και να δράσει με βάση τις ε, διεθνείς υποχρεώσεις της από συμβάσει και διεθνεί συνθήκες. Επίσης, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η στρατηγική μας για την Αφρική να εδράζεται σε φιλοδοξίες που θα είναι φάμιλες με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξη και να ασκήσουμε πιέσει για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Ευχαριστώ, κύριο Σίντζιτς, για ένα λεπτό. Δυστυχώ, χωρίς μικρόφωνο, κύριο Σίντζιτ. Το γεγονός ότι στη Μαδαγασκάρη τα παιδιά δουλεύουν ε, στα ορυχεία για 12 ώρες και για 40 λεπτά του ευρώ τη μέρα είναι ντροπή για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και δεν είναι το μοναδικό παράδειγμα. Έχουμε στα ορυχεία Κοβαλτίου στην Κίνα παρόμοια εκμετάλλευση των παιδιών και γι' αυτό φταίει ο νεοφιλελευθερισμός και το οικονομικό σύστημα που ε, καταστρατηγεί τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικολογικά δικαιώματα. Πρόκειται για ένα νεοφιλελεύθερο σύστημα που εξολοθρεύει το μέλλον των ε, νέων γενιών. Είναι ένα σύστημα που είναι η αντίθεση της βιωσιμότητας και της αφορίας για την οποία υποτίθεται κοπτόμαστε. Θα πρέπει λοιπόν ε, να βρούμε ένα άλλο σύστημα για να εξασφαλίσουμε το μέλλον και αποκέντρωση της ε, ιδιοκτησίας ε, στην ενέργεια και τα προϊόντα, τα τρόφιμα. κύριος Χέτμαν. Πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά δυστυχώ στη Μαδαγασκάρη εξαναγκάζονται σε εργασία και ε, πολλέ χιλιάδε απασχολούνται στο ρηχέ σε επικίνδυνες συνθήκες. Οι αρχέ της Μαδαγασκάρης έκαναν κάποια πρόοδο και ρύθμισαν νομοθετικά το πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να αναλυφθούν και αποφασιστικέ δράσεις. Ζητούμε λοιπόν από τη Μαδαγασκάρη να διενεργήσει σωστέ επιθεωρήσεις και ελέγχου, να τιμωρήσει τις καταχρήσεις και να ανακαλέσει την άδεια των ορυχείων που χρησιμοποιούν ε, την παιδική εργασία. Βέβαια, αιτία της ε, κατάστασης αυτής ε, είναι η φτώχεια πάνω από 70% των ε, κατοίκων της Μαδαγασκάρης ζουν στα όρια της φτώχειας και πάνω από 60% των παιδιών είναι μονίμως υποσυτισμένα. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να εξαλείψουμε τη φτώχεια για να φροντίσουμε και το θέμα της παιδικής εργασίας. Θα πρέπει να βοηθήσουμε με αναπτυξιακή βοήθεια τη Μαδαγασκάρη και προτεραιότητα αυτή τη αναπτυξιακή βοήθεια να είναι η πρόσβαση στην παιδεία. Η παιδεία είναι απαραίτητη και για το μέλλον του κάθε παιδιού αλλά και για το μέλλον της ίδιας της χώρας. Ευχαριστώ. Φόλατ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 11.000 παιδιά και στη Μαγατασκάρη και 152 εκατομμύρια παιδιά σε όλη τον κόσμο ε, που χάνουν τη ζωή του για την παραγωγή τέτοιων ε, υλικών. Αυτό αποτελεί ε, ένα ζήτημα για την Ευρώπη και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατεπηγόντως να δράσει προκειμένου επικοδομητικά να κοιτάξουμε μια δεσμευτική συμφωνία για τις διασυνοριακές εταιρείε σε όλο τον κόσμο προκειμένου να μπορέσουμε όλοι να συμμετέχουμε σε αυτό. Και είναι κρίμα το γεγονό ότι δεν έρχεται το Συμβούλιο σήμερα στη ζήτηση αυτή. Γιατί σε θελούσια βάση δεν λειτουργεί το σύστημα. Οι μεγάλε ε, ε, αλυσίδε ανεφοδιασμού δεν μπορούν να αποφύγουν την παιδική εργασία. Χρειαζόμαστε λοιπόν δεσμευτικού κανόνε και κυρώσει. Η απαγόρευση τη παιδική εργασία θα πρέπει επιτέλου να καταστεί ορόσημο για τι διεθνεί μα σχέσει, γιατί είναι υποκρισία αυτή που κάνουμε. Θα πρέπει το κέρδος να μπαίνει πίσω από την προστασία της ζωής και της αξιοπρέπειας των παιδιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος. Η κυρία Βυσνιεύσκα είναι η επόμενη στον κατάλογο, δεν τη βλέπω όμω στην αίθουσα. Αν θέλει να ζητήσει το λόγο, Ιτάλος να ακούσουμε τον συνάδελφο του κύριο Γεντρών. Για ένα λεπτό. you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η εργασία ε, όταν κανείς είναι ενήλικος ονομαστεί εργασία, αλλά στην παιδική ηλικία η εργασία θα έπρεπε να είναι το παιχνίδι, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν η παιδική εργασία αποτελεί ένα οξύμορο. Δυστυχώς, ε, παιδιά μέχρι και 5 ετών ε, είναι πάνω από το ίμιση των ε, ατόμων που εργάζονται στα ορυχεία στην Μαγαδασκάρη. 11.000 λοιπόν παιδιά εργάζονται στα ορυχεία μαρμαριών στην Μαγαδασκάρη. Ξέρετε τι σημαίνει λοιπόν αυτό, ότι τα παιδιά αυτά εργάζονται και για μας, για τους Ευρωπαίους τελικά. Στη Μαγατασκάρη. ο κόσμος εξαρτάται από τα ορυχεία. το βιός τους εξαρτάται. Θα πρέπει να σταματήσει όμως η εκμετάλλευση των παιδιών και θα πρέπει να σταματήσει εδώ. Να σταματήσουμε και την υποκρισία μας, εγκρίνοντας το νόμο που θα απαγορεύσει την παιδική εργασία σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ραφάλσκα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει καμία δικαιολόγηση για τη χρήση της παιδικής εργασίας. Και μάλιστα πολύ συχνά παιδική εργασία υπό άθλιες, επικίνδυνες και πολύ δύσκολες συνθήκες. Ε, και δυστυχώς πάνω από 351 εκατομμύρια παιδιά απασχολούνται διεθνώς και 100 εκατομμύρια με επικίνδυνες εργασίες. Αυτό δείχνει την κλίμακα μεγέθους του προβλήματος. Και δραματική κατάσταση έχουμε και στη Μαδαγασκάρη με υψηλό επίπεδο φτώχειας. 74% του πληθυσμού βρίσκονται στο κατόφυλλο της φτώχειας και σίγουρα η ανέχεια είναι ε, ο σημαντικότερος ε, λόγος και παράγον της παιδικής εργασίας. Τα περισσότερα παιδιά είναι υποσυτισμένα στη Μαδαγοσκάρη και οι ε, γυναίκες ε, χάνουν τη ζωή τους και στη διάρκεια του τοκετού ο αριθμός είναι διπλάσιος από ό,τι στην Ευρώπη, στην Πολωνία. Και πολύ συχνά τα παιδιά απασχολούνται σε επικίνδυνες συνθήκες, κυρίως στα ορυχεία μαρμαριγιών. Θα πρέπει λοιπόν να στήσουμε την Πεδαγασκάρη να σεβαστεί τα δικαιώματα των παιδιών και να σταματήσει η παιδική εργασία και θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικό ο τρόπος που πετούμε αυτή την τήρηση. Για τη διαδικασία Catch έχω έξι άτομα που ζήτησαν τον λόγο από τρει πολιτικέ ομάδε. Θα πάρω έναν από κάθε, από κάθε πολιτική ομάδα. Η Επίτροπο χρειάζεται πολύ χρόνο για να μιλήσει. Αν δεν έχετε αντίρρηση, να δώσω σε τρία άτομα το λόγο. Νόβακ. Ένα λεπτό. Η χώρα μου, η Σλοβενία, είναι μικρή χώρα, αλλά παρόλα αυτά έχουμε πάρα πολύ στενές σχέσεις με τη Μαδαγασκάρη, διότι πολλοί Σλοβαίνοι ιερείς ε, είναι γεραπόστολοι ε, στις χώρες αυτές. Δεν εργάζονται φυσικά μόνο ως ιερείς, αλλά ασχολούνται και με την ε, ευημερία του πληθυσμού εκεί. Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα είναι ο Πέτερο Πέκαχο, ο οποίος ε, πηγαίνει σε παραγκουπόλεις ε, και βοηθά για να μπορέσουν να εγκατασταθούν οι άνθρωποι σε ειδικέ εγκαταστάσεις. και δίνουν τη δυνατότητα σε οικογένειε να ζήσουν σε μικρέ κατοικίε και να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε σχολείο. Έχουν οργανώσει τη ζωή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τους προσφέρουν ε, εργασία και εκπαίδευση για τα παιδιά. Αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα για να βοηθήσουμε τον τρίτο κόσμο. Και το παράδειγμα του το ακολούθησε και ο Πάπας και η ε, κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης. Παρακαλώ καθίστε ησύχως και να δώσω το λόγο στην κυρία Κιμίτση. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Μαδαγασκάρη είναι μία από τις πιο φτωχές χώρες στον κόσμο και παρά το γεγονός ότι επισήμως απαγορεύεται η παιδική εργασία, ε, περίπου το 1 τέταρτο των παιδιών από 5 έως 15 ετών είναι υποχρεωμένοι να, εργάζονται σε φοιτίες ε, βανίλιες, ε, στα ορυχεία και φυσικά σε οικιακές εργασίες. Και είναι δραματική η κατάσταση των παιδιών που κάθε μέρα εργάζονται στα ορυχεία. Είναι πάρα πολύ σκληρές οι συνθήκες και επικίνδυνες για την υγεία του. Τέσσερα ε, σεντ ε, το κιλό παίρνουν για να ε, κόβουν ε, τις πέτρες από τα ορυχεία και να έρχονται σε επαφή με ζημιογόνες και επικίνδυνες ουσίες. Ε, γιορτάσαμε τα 30 χρόνια του ψηφίσματο για την ε, ε, προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Δεν θα πρέπει να μείνουμε στα ευρωπαϊκά σύνορα για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Θα πρέπει να καταγγείλουμε αυτέ τι απαράδεκτε παραβιάσεις, να ενεργοποιήσουμε επίση και τι κατάλληλε πολιτικέ για να αναλάβει τις ευθύνες της βιομηχανία που χρησιμοποιεί τέτοια υλικά και να βοηθήσουμε τι πιο φτωχέ χώρε. Κυρία Επίτροπε, θα πρέπει να δεσμευτούμε όλοι για να εφαρμόσουμε ε, τα όσα προβλέπονται από την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Ντέιλι. Παρακαλώ, ε, καθίστε ησύχως, επαναλαμβάνω. Δεν θα έλεγα, η κυρία Ντέιλι, ότι υπάρχει κάποιος που έχει συναντήσει κάποιον που υποστηρίζει την καταναγκαστική παιδική εργασία. Για όνομα του Θεού, εχθέ ε, περάσαμε ένα ψήφισμα σε μια χώρα όπου υπάρχει παιδική εργασία. Ποιο αμφισβητεί γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πιστεύετε ότι οι γονεί αυτών των παιδιών στη Μαδαγασκάρη δεν τα αγαπούν και ότι δεν θέλουν να πάνε σχολείο. Φυσικά και τα αγαπούν και θέλουν να πάνε σχολείο, αλλά δεν έχουν αναλλακτική λύση γιατί τα παιδιά του είναι θύματα του καπιταλισμού, τη ε, βιομηχανική γεωργίας, τη κλιματική αλλαγή και τη ξηρασίας. Και εμεί έχουμε πολυεθνικέ από ευρωπαϊκέ χώρε οι οποίε έχουν επιχειρήσει και εργασίε εκεί. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να πω ότι αυτά τα ψηφίσματα είναι λυπηρά. Ε, πονίδιστο να ζητάμε απλώ, ε, ε, σαν να ζητάμε από ένα λύκο να μην φάει την κατσίκα. Πού είναι οι ποινέ, πού είναι οι ποινικέ ε, ευθύνε, ε, πού είναι η δεσμευτική νομοθεσία. Δεν χρειάζονται κροκοδίλια δάκρυα, χρειαζόμαστε πράξει Thank ευχαριστώ και τώρα να δώσω το λόγο στην Επίτροπο, στην κυρία Ντάλη, και θα ήθελα παρακαλώ να σας ζητήσω να σεβαστείτε τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθίστε στις θέσεις σας, αλλά με ησυχία. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, τους τελευταίους μήνες είδαμε κάποιες σοβαρές και ε, πολύ ενοχλητικές ε, και αποκαλύψεις για την παιδική εργασία στη Μαγατασκάρη σε παιδιά τα οποία δουλεύουν στο ρηχείο μαρμαριών. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε λοιπόν μια κατάσταση τέτοια όπου τα παιδιά εξαναγκάζονται. Ναι, έχω πολύ ανταγωνισμό. Συγγνώμη, ζητά η Πρόεδρο. Συνάδελφοι, δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά σταμάτησε να μιλάει η Επίτροπο. Γιατί έχει τόση φασαρία. Σα παρακαλώ πολύ ήσυχα. Σα ευχαριστώ. Η Πρόεδρο, σα παρακαλώ, καθίστε με ησυχία ή μείνετε εκτός οθούσες. Δεν μπορούμε λοιπόν να ανεχτούμε μια κατάσταση κατά την οποία τα παιδιά εξαναγκάζονται να εργάζονται υπό φρικτές συνθήκες και δεν ε, έχουν το δικαίωμα της εκπαίδευσης. Θα πρέπει λοιπόν να δράσουμε και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και τις βαθύτερες αιτίε. 46.000 τόνοι μαρμαριών εξαγάγει η Μαγαπασκάρα. Το 2018 το η συντατική πλειονότητα ε, πήγε στην Κίνα. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν το θέμα της δέωσης επιμέλειας στην ε, αλυσίδα ανεφοδιασμού. Αλλά η ενίσχυση των ικανοτήτων των κρατικών αρχών ε, της Μαγατασκάρης μέσω και της αναπτυξιακής βοήθειας θα αποτελέσει ένα θέμα κλειδί. Θα θυμάστε πολλοί από εσά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει θετικέ δράσει για να καταπολεμήσει του κινδύνου στην αλυσίδα ανεφοδιασμού σε ό,τι αφορά αυτά τα ορεικτά που αποτελούν ε, κίνδυνο σε ό,τι αφορά το χρυσό, για παράδειγμα, και άλλε τέτοιε και τέτοια μεταλλεύματα. Του χρόνου θα τεθεί σε εφαρμογή η νομοθεσία αυτή. Η πρόεδρο, σα παρακαλώ, συνάδελφοι, καθίστε και μην κάνετε φασαρία γιατί μιλάει για Επιτροπός. Δεν μπορούμε να καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα και να επιτρέπουμε παιδική εργασία. Ένα οξύμερο, όπως ε, σωστά τοποθέτησε, το τοποθέτησε ο Ρόμπερτ Μιέντρον. Η παιδική εργασία λοιπόν στα ορυχεία και στις εκτορυκτικές αυτές μηχανίες να συνεχίζεται. Θα πρέπει οι διεθνείς εταιρείε οι οποίες χρησιμοποιούν μαρμαργία και η κυβέρνηση της Μαγαδασκάρης να αναλάβουν τις ευθύνες τους για να επιλύσουν το πρόβλημα αυτό και να αντιμετωπίσουν τις προβληματικές αυτές συνθήκες και να βελτίωσουν σε ό,τι αφορά την, τα δικαιώματα των παιδιών αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τοποθετηθεί εδώ και καιρό σε ό,τι αφορά τη δέουσα επιμέλεια. Όχι μόνο οι κυβερνήσεις, αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς έχουν το ρόλο τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Νοέμβριο του 2019 οργάνωσε μια σημαντική εκδήλωση όπου επέστησε την προσοχή στο θέμα το κατεπήγον πρόβλημα τη εξόρυξη μαρμαργιών. Εδώ τονίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μηδενική ανοχή σε ό,τι αφορά την παιδική εργασία. Ακολουθούσε ένα ψήφισμα για τα δικαιώματα των παιδιών που εγκρίθηκε το πέρσι από την ειδική συνέλευση του ΟΗΕ το 2021 ανακηρύχθηκε το Διεθνές ε, έτος για την ε, κατάργηση της παιδικής εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει σύντομα ε, τη μελέτη της για την δεσμευτική δέουσα επιμέλεια σε ό,τι αφορά την παιδική εργασία και περιλαμβάνει στοιχεία για την επιβολή της δέουσας επιμέλειας της εταιρείε της αλυσίδα ανεφοδιασμού σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε ό,τι αφορά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο, και σε ό,τι αφορά φυσικά το σκέλος της αλλαγής του κλίματος σε μια ενιαία αγορά δεν είναι πρακτικό να υπάρχουν ε, διαφορετικά εθνικά συστήματα και τα ωφέλη ενός πανευρωπαϊκού συστήματος είναι προφανή σε ό,τι αφορά τους ίσους όρους ανταγωνισμού, σε ό,τι αφορά τη νομική βεβαιότητα για τις ε, εταιρείε, αλλά και στο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την βιώσιμη μετάβαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλώ και υποστηρίζει και τι πρωτοβουλίε πολλαπλών φορέων για να μειωθούν οι κίνδυνοι στην αλυσίδα ανεφοδιασμού και κυρίω η παιδική εργασία. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να εργαζόμαστε σε ό,τι αφορά και τι ε, εμπορικέ συμφωνίε και άλλε συμφωνίε για διεθνή συνεργασία στην αμαγατασκάρη, αλλά και αλλού για να αντιμετωπίσουμε τι βαθύτερε αιτίε, όπω είναι η οικονομική και κοινωνική ευαλωτότητα των ατόμων, των εργαζομένων, των οικογενειών τους που τελικά καταλήγουν να σπρώχνουν τα παιδιά στην παιδική εργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λεκή Πρόεδρος. Και έτσι ολοκληρώθηκε η συζήτηση αυτή και στο τέλος κατατέθηκαν 7 ψηφίσματα για τα οποία θα ψηφίσουμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, ας περάσουμε στις ψηφοφορίες. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σας κάνω μια ανακοίνωση. Η ομάδα Renew ενημέρωσε τον Πρόεδρο για τις εξής αποφάσεις ε, για τις αλλαγές σε διορισμούς. Η Καταλίν Τσέχ αντικαθιστά τον Νίκολα Ντάντε στην Επιτροπή ΑΦΕΤ και ο Νίκολα Ντάντ κυρία Τσέχ στην Επιτροπή Ήτρε. Οι αποφάσεις αυτές ε, θα τεθούν σε ισχύ από την ημέρα της ανακοίνωσης. Περνάμε στις ψηφοφορίες τώρα. Θέλει κάποιος διαδικαστικό? Eh, Πρόεδρε, ένα διαδικαστικό, επιτρέψτε μου. Θα μπορούσατε να ζητήσετε από τις υπηρεσίε να... σε ό,τι αφορά τα email μα και τα spam, γιατί μας στέλνουν ε, τόσες πολλά email τελευταία, ε, τους τελευταίους μήνες. Τι νόημα έχει να λαμβάνουμε 600 email μα ενοχλεί και μα εμποδίζει στι εργασίε μα. Μπορείτε να ζητήσετε από τι τεχνικέ υπηρεσίε να το αντιμετωπίσουν. Ε. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια δυνατότητα. We took... We took notes. Το σημειώσαμε, συναδελφέ. Θα ενημερώσω τις υπηρεσίες. Και επίσης Ε, πάντως έχετε το, το δικαίωμα και τη δυνατότητα να βάλετε τους δικούς σας κανόνες, το δικό σας φίλτρα, ούτως ή άλλως. Περνάμε στις ψηφοφορίες. Ψήφισμα για το Γουινέα Κόνακρη, ιδίως η βία εις βάρος των διαδηλωτών. Ψηφίζουμε διανατάσεις χειρός υπέρ του κοινοψηφίσματος κατά αποχές. Εγκρίνεται. ψηφίζουμε το ψήφισμα για την παιδική εργασία σε ορυχία της Μαδαγασκάρης. Θα ψηφίσουμε πρώτα το ψήφισμα της Ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατίας. Με διαμετάσεις της χειρός, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα το κοινό ψήφισμα έξι πολιτικών ομάδων. Τροπολογίες 1 και 7 πανομοιότυπες με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Το αρχικό κείμενο καταπίπτει. Τροπολογία 8 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απόρριψη. Απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Καλώς. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικός έλεγχος στην τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ευχαριστώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ζητώ συγγνώμη, εγκρίνεται τελικά. Τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Χωρίς έλεγχο παρακαλώ. Τροπολογία 3 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5, διανατάσσεως της χειρός. Διαδικαστικό. Ναι, ένα διαδικαστικό. Το τελευταία ψηφοφορία δεν δουλεύει το μηχάνημά μου. Αλήθεια. Οπότε παρακαλώ υπολογίστε και τη δική μου ψήφο. Βάσει του εσωτερικού κανονισμού δεν αλλάζει τίποτα στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Σε προηγούμενες ψηφοφορίες λειτουργούσε η συσκευή σας ήταν μόνο στην τελευταία που χάλασε. Καλά, αφού έτσι το ερμηνεύεται. Αυτό προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός. Αν η συσκευή σας δεν λειτουργεί, αλλάξτε θέση. Ψηφίζουμε την τροπολογία 5. Διανοτάσεως της χειρός. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε ολόκληρο το ψήφισμα. Διανοτάσιο της χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προχωρούμε τώρα στην έκθεση Μέτσολα. Ψηφίζουμε για την προσφορινή συμφωνία με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν ολοκλήρωσε την πρώτη ανάγνωση. Περνάμε τώρα στι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την 64η Σύνοδο τη Επιτροπή του ΟΗΕ για τη θέση τη γυναίκα. Ψηφίζουμε πρώτα το ψήφισμα τη ομάδα ECR. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα το ψήφισμα των πέντε πολιτικών ομάδων. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Τροπολογία 1 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, Άποχες. Επαλήθευση. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Παράγραφος 1-1. Το αρχικό κείμενο. Υπέρ. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Υπήρχε ένα διαδικαστικό. Απλώς να πω κύριε Πρόεδρε ότι στην ονομαστική κλήθη που έγινε για την επαλήθευση είχατε λάθος τροπολογία στην οθόνη. Ψηφίζαμε την τροπολογία 1 και όχι 2. Αυτό που είχατε στην οθόνη ήταν το δεύτερο τμήμα, αν θυμάμαι καλά. Okay, we... Συνεχίζουμε. Παράγραφος 1, σημείο M, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Παράγραφος 1, σημείο M, αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφο 1, σημείο Β, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 1, σημείο X, αρχικό κείμενο σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία εγκρίνεται. Παράγραφος 1, σημείο AA, αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά, άποχες, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά, άποχες, εγκρίνεται. Παράγραφος 1, σημείο BB. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 1, σημείο JJ, αρχικό κείμενο με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη F. Αρχικό κείμενο σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, μονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη και σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, μονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη M, Διανατάσσεω χειρό, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα, πριν ε, την τελική ψηφοφορία ε, για το ψήφισμα συνολικά, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι δεν θα πρέπει να βγάλετε την κάρτα σας από το μηχάνημα πριν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, γιατί αλλιώς δεν θα καταγραφεί η ψήφο σας. Ψηφίζουμε λοιπόν το ψήφισμα συνολικά με ονομαστική κλίση «Άρχεται η ψηφοφορία». Πέραση της ψηφοφορίας και εγκρίνεται Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.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 Can I ask Συνάδελφοι, παρακαλώ, όσοι δεν θα μείνετε στην αίθουσα για τις επεξηγήσεις ψήφου, παρακαλώ να αποχωρήσετε ήσυχα για να μπορέσουν ε, να ακολουθήσουν οι αιτιολογήσεις ψήφου. Ναι, Παρακαλώ συνάδελφοι, αν δεν έχετε αιτιολόγηση ψήφου ή δεν θέλετε να ακούσετε τις αιτιολόγηση ψήφου, παρακαλώ αποχωρήστε από την αίθουσα, γιατί οι συνομιλίες σας ενοχλούν τους συναδέλφους που θα παραμείνουν. Συνάδελφοι, περνάμε στις αιτιολογήσεις ψήφου και ξεκινάμε με την έκθεση Μετσόλα και πρώτη επεξήγηση ψήφου. Συνάδελφοι, παρακαλώ, αθόρυβα αποχωρήστε από την αίθουσα. Πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Ζόντσα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη ικανοποίηση έμαθα ότι ο οργανισμός Frontex θα έχει και ένα επιπλέον μέσο για την καταπολέμηση των απατών και αυτό το επιγραμμικό μητρό είναι πολύ χρήσιμο γιατί χρησιμοποιούν πολύ συχνά ε, τα πλαστά έγγραφα οι κακοποιοί. Και δεν το κάνουν αυτό οι φτωχοί απλοί άνθρωποι, το κάνουν α, κάποιοι που κερδίζουν χρήματα από τέτοιε απάτες. Ε, μια επικίνδυνη κατάσταση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον κόσμο ολόκληρο. Και οι εγκληματίες που χρησιμοποιούν αυτή την κατάσταση και χρησιμοποιούν πλαστά έγγραφα ή ε, βγάζουν πλαστά έγγραφα για κακοποιούς οι εγκληματίες, οι άνθρωποι αυτοί παραβιάζουν την ε, τοπική, εθνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια δημόσια τάξη. Πολύ καλή λύση, πολύ καλή πρόταση και ελπίζω χάρη στο μέσο αυτό να μπορεί ο Frontex να αναλύει διεξοδικά όλες τις ε, καταστάσεις αυτές και να κάνει τι απαραίτητε έρευνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ένα λεπτό, το λόγο έχει ο κύριος Γκρουτζίνσκι. Κύριε Μπρουτζίνσκι, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, φυσικά και υπερψήφισα το επιγραμμικό μητρό γιατί είμαι υπέρ των μέσων που καταπολεμούν τις απάτες που σχετίζονται με πλαστά έγγραφα. Και σήμερα οι συνοριακέ αρχέ των κρατών μελών για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν τέτοια, τέτοια μορφή εγκληματικότητα, θα πρέπει να συνεργαστούν. Και γι' αυτό και ο Frontex αλλά και οι μεμονωμένες υπηρεσίες των αρμόδιων χωρών ε, για την ασφάλεια των επιγραμμικών γράφων θα πρέπει να βρίσκονται ένα βήμα πιο μπροστά από τους ε, κακοποιούς και εγκληματίες. Και γι' αυτό απευθύναμε έκλειση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει όσο το δυνατό γρηγορότερα γίνεται το κανονισμό, προκειμένου να εφοδιάσει τι αρμόδιε αρχέ των κρατών μελών και το Frontex με αποτελεσματικά μέσα για να καταπολεμήσουν τέτοιου είδου απάτε, όπω είναι αυτέ με τα πλαστά έγγραφα. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα σε αιτιολογήσεις ψήφου για την πρόταση ψηφίσματο με θέμα τη προτεραιότητε Ευρωπαϊκή Ένωση για την 64η Σύνοδο τη Επιτροπή στο ΟΗΕ για τη θέση τη γυναίκα. Ο κύριο Ράιλ είναι ο πρώτο ομιλητή. Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, καταψήφισα το ψήφισμα αυτό. Φυσικά είμαστε υπέρ των δικαιωμάτων τη γυναίκα, πρέπει να τα υποστηρίξουμε. Αλλά εδώ ζητούνται ανοησίε για την έγκαιρη σεξουαλική εκπαίδευση σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της ταυτότητας του φίλου. Αυτό για μένα είναι άρρωστο. Έχουμε άλλα προβλήματα. Για παράδειγμα, σε άλλες χώρες μία στις τρεις γυναίκες δολοφονείται και αυξάνεται ο, ο αριθμός των δολοφονιών αυτών. Η ενδοοικογενειακή βία έχει αυξηθεί από το 2014 στη Γερμανία. 140.000 το 2018 και οι δράστες είναι κυρίως μετανάστες και όχι μόνο οι μετανάστες είναι δράστες αλλά και τα θύματα είναι ε, μετανάστες Την Έση, την πατρίδα μου, οι γυναίκε ε, ε, που πηγαίνουν να ψάξουν ιδρύματα για να ζήσουν εκεί είναι κατά 60% μετανάστριε. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα και αυτά πρέπει να επιλύσουμε. Ευχαριστώ. κυρία Ζωρών λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Συνάδελφοι, αυτό το κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποτίθεται ε, με ψηφίζει ένα ψήφισμα σε ό,τι αφορά τα, δικαιώματα τη γυναίκε. σε ό,τι αφορά τι γυναίκε που εκτελούνται. Δεν λέγεται όμω για την γυναίκα αυτή η οποία ε, την πνίξανε 16 ετών. Και η Σαλομίν δεν είναι στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στην Κολομβία, ούτε στο Μπρόγκ καν. Η Σαλομίν ζει στην Ευρώπη, εδώ, στη Γαλλία ζει χίλιες επιθέσεις στην ε, Γαλλία κάθε μέρα, ε, σεξουαλικές επιθέσεις, δολοφονίες. Θεσμοποιούμε τις ε, δράσεις αυτές σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ. Τι σημαίνει αυτό, ότι θέλουμε ένα τέταρτο να λέμε γυναίκες, τέταρτα μειονεκτικής πληθυσμού. ανέχομαστε τις επιθέσεις αυτές και αυτό θα το θυμούνται οι Γαλλίδες. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι καταψήφισα το κείμενο αυτό λόγω όλων αυτών των στοιχείων που ανέφερα. Ο κύριος Τόμακ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος αυτού και πιστεύω ότι είναι κρίσιμη σημασία να αποτίσουμε φόρο τιμής για τις πολιτικές εκείνες και όλα στις μορφές καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Οι γυναίκες πρέπει να προστατεύονται. Ακόμα έχουμε γυναίκες σε πολύ φτωχέ περιοχές στην Ευρώπη που αντιμετωπίζουν την διακριτική αυτή μεταχείριση και μάλιστα καθημερινά στο πετσί τους. Δεν έχουν πρόσβαση στο χρηματοοικονομικό σύστημα, στα χρήματα, σε επενδύσεις, ε, ούτε έχουν αξιοπρεπείς ε, συντάξεις. Αυτά τα προβλήματα εξακολουθούν να μας θέσουν την Ευρώπη και θα πρέπει να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Είμαι υπέρ λοιπόν της καλύτερης εκπροσώπησης των γυναικών και είμαι υπέρ της καταπολέμησης κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών. Και μόνο ε, με τα υψηλά αυτά πρότυπα μπορούμε να καταπολεμήσουμε πραγματικά τα φαινόμενα αυτά. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαϊμπή για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι η δεύτερη φορά σε δύο μέρε που ψηφίζουμε κάτι για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίσαμε κάτι για την ανισότητα του εισοδήματο μεταξύ ανδρών και γυναικών και τώρα συζητάμε τι προτεραιότητε Ευρωπαϊκή Ένωση για την 64η Σύνοδο, Συνόδο των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση τη γυναίκα. Επομένω, ε, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση τη γυναίκα και για άλλη μια φορά σε αυτό το κείμενο, το οποίο υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία, για άλλη μια φορά διαβάζω ότι η λύση για να μειώσουμε τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι να αυξήσουμε τις συντάξεις των γυναικών και επίσης να αναπτύξουμε και τις ε, ε συντάξεις, αυτά τα επιδόματα που δίνονται ε, σε χείρα ή σε χείρο ε, μετά το θάνατο του συζύγου τους. Και μάλιστα το Common Mars υπερψήφισε και εδώ έχουμε ε, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Υπερψηφίζουν με ε, το ψήφισμα αυτό και ταυτόχρονα στην ε, Γαλλία η κυβέρνηση που εκπροσωπεί ο πρόεδρος Μακρόν αρχίζει τη διαδικασία αντιστροφής της σύνταξης χειρίας και πραγματικά θα ήθελα να ξέρω εάν πραγματικά θέλουμε να έχουμε ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Όλεκας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο μία από τι θεμελιώδει αρχέ τη κοινωνία μα, αλλά είναι και απαραίτητη προκειμένου να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και να εξασφαλίσουμε την ευημερία. Πρέπει να είμαστε πιο δραστήριοι στον τομέα αυτό, ιδίω στην καταπολέμηση διαφόρων μορφών διακρίσεων. Πρέπει να είμαστε πιο ε, δραστήριοι, να προσπαθήσουμε να μειώσουμε το μισθολογικό χάσμα και το ε, συνταξιοδοτικό χάσμα και επίσης να ενθαρρύνουμε περισσότερες γυναίκες ε, να μορφώνονται ιδίως ε, σε περιοχές τις οποίες είναι πολύ χαμηλή η εκπροσώπηση των γυναικών. Επίσης θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και την σεξουαλική εκμετάλλευση, την ανθρώπινη εμπορία, τους καταναγκαστικούς γάμους, ε, τον ακροτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων και να δώσουμε ένα τέλος ε, στη χρήση γυναικών ως ασπίδα σε ένοπλες ε, σειράξεις. Ολοκληρώνεται η διαδικασία ε, αυτή και έχουμε διακοπή μέχρι τις 3. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, επανάληψη της Συνόδου. Τα χθεσινά πρακτικά και τα εγκριθέντα ψηφίσματα υπάρχουν στη διάθεσή σας. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, θεωρούνται ως εγκεκριμένα τα πρακτικά. Περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημέρηση διάταξη, στη δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια. Να σα υπενθυμίσω ότι μπορείτε να ζητήσετε το λόγο δυνάμει τη διαδικασία μπλε κάρτα και catch the eye, χρησιμοποιώντα και το σύνηθε σύστημα, το σύστημα και το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφή. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να δώσω το λόγο στην Επίτροπο Βαλεάν για να μας κάνει τη δήλωσή της για την οδική ασφάλεια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σας αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ καταρχήν που θέσατε στην ημερήσια διάταξη ένα τόσο σημαντικό θέμα. Σημαντικό για όλους μας και για σας και για μένα, την Επίτροπο Αρμόδια για τις Μεταφορές. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις απόψει μου πριν μεταβώ στη Στοκχόλμη στις 19 Φεβρουαρίου για την τρίτη παγκόσμια υπουργική διάσκεψη με θέμα την οδική ασφάλεια. Είναι καθήκον μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να προστατεύσουμε τη ζωή και την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. 25.000 άνθρωποι χάνουν την ζωή τους στους ευρωπαϊκούς δρόμους και 135.000 υποφέρουν από βαρύτατος τραυματισμούς από τροχαία ατυχήματα. Είναι απαράδεκτα αυτά τα νούμερα. Και θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, τις δράσεις μας και την υποστήριξή μας στην ενίσχυση της ε, οδικής ασφάλειας. Οπότε η οδική ασφάλεια θα είναι και δική μου προτεραιότητα και με τη δική σας βοήθεια θα την καταστήσουμε πανευρωπαϊκή προτεραιότητα. Ας μην ξεχνούμε ότι ήδη έχουμε σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο στην οδική ασφάλεια τις τελευταίες δεκαετίες είμαστε η ασφαλέστερη περιοχή του κόσμου από την άποψη των οδικών ατυχημάτων και έχουμε πλούσια πείρα και καλές πρακτικές που μπορούμε να τις μοιραστούμε με τους άλλους εταίρους. Και είναι μια μοναδική ευκαιρία για να ηγηθούμε παγκοσμίω στο θέμα της οδικής ασφάλειας. 1,35 εκατομμύρια στον κόσμο χάνουν τη ζωή τους ε, στους ε, δρόμους και τα θανατηφόρα τροχαία είναι η πρώτη αιτία θανάτου των νέων παγκοσμίω. Και ο στόχο μα να μειωθεί παγκοσμίω κατά 50% ο αριθμό των τροχαίων, των θανατηφόρων τροχαίων, ω τμήμα των στόχων βιώσιμη ανάπτυξη, λύγει φέτο. Και δυστυχώ δεν καταφέραμε, ούτε πρόκειται να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα υποβαθμίσουμε τι φιλοδοξίε μα. Θα πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι στην υλοποίηση του στόχου μείωση παγκοσμίω ε, των θανατηφόρων τροχαίων. Και αυτό θα το διατρανώσω και στη Στοχόλμη. Ο Σουηδός Υπουργό Υποδομών θα υποβάλει στη Στοκχόλμη την ε, διακήρυξη της Στοκχόλμης που θα ζητήσει ανανέωση των προσπαθειών και νέους παγκόσμιους στόχους. Είμαι υπέρ της διακήρυξης αυτής και ευελπιστώ ότι θα υιοθετηθεί όπως έχει προγραμματιστεί. Το επόμενο θα, βήμα θα είναι ένα ψήφισμα στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και εκεί θα στηρίξουμε τη διαδικασία για την έγκριση ψηφίσματος μέσω και των δύο γραφείων μας, τη Γενέβη και τη Νέα Υόρκη. Και αυτό που μετράει σε τελική ανάλυση είναι τα αποτελέσματα. Στην Ευρώπη εφαρμόζουμε την ε, προσέγγιση του ασφαλού συστήματος. Πρόκειται για μια σφαιρική προσέγγιση, ένα σφαιρικό σύστημα που εδράζεται στη συνεργασία, τη χρηστή διαχείριση και την επιμερισμένη ευθύνη. Επίσης, ε, καλύπτει όλους τους τομεί. Τις υποδομές, τα οχήματα και την ε, φροντίδα μετά το ατύχημα. Φυσικά το ανθρώπινο λάθος πάντα είναι δυνατό. Αυτό προβλέπει το σύστημα και προσπαθεί να το διορθώσει. Και μάλιστα οι οδηγοί και άλλοι χρήστες που θα κάνουν λάθη ε, στο δρόμο, όπως γίνεται και παντού, γιατί ε, το λάθος είναι ανθρώπινο, ανθρώπινο και σίγουρα η χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών αυξάνει το βαθμό λάθους, αλλά κανένας χρήστης δεν θα πρέπει να χάνει τη ζωή του λόγω αυτών των λαθών. Και μάλιστα υποστηρίξαμε αυτούς τους παγκόσμιους στόχους για τη μείωση κατά το ίμιση των, ε, ε, μέχρι το 2030 των θανατηφόρων ε, ατυχημάτων και των σοβαρών τραυματισμών και μάλιστα έχουμε υποβάλει ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης. Έχουμε ήδη λάβει και τις πρώτες αποφάσεις και έμπρακτες αντιδράσεις. Χάρη στη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενισχύσαμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και για την διαχείριση, ασφαλή διαχείριση των υποδομών και για την ασφάλεια των οχημάτων. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε φιλόδοξες νομοθετικές διατάξεις στη διάρκεια της θητείας μας και προσβλέπω σε ενδελεχή συζήτηση στο μέλλον των επιμέρους προτάσεων. Στο μεταξύ θα πρέπει να συνεργαστούμε, γιατί η συνεργασία είναι η πεμπτουσία του συστήματος ασφαλούς προσέγγισης για την οδική ασφάλεια. Και έτσι ε, πιστεύω ότι έχουμε τα εφόδια ώστε στη συνεργασία με τα κράτη-μέλη, τη βιομηχανία, τη ΜΚΟ, την κοινωνία των πολιτών να καταλήξουμε σε πιο φιλόδοξους στόχους και να προωθήσουμε φυσικά τις δράσεις και στις εκλογικές μας περιφέρειες. Σίγουρα η κινητικότητα αλλάζει ριζικά. Ε, οι κλιματικές αλλαγές μας υποχρεώνουν να μειώσουμε τις εκπομπές, ενώ η ψηφιοποίηση προβλέπει νέες ευκαιρίες για ασφαλέστερη και πιο καθαρή και οικολογική κινητικότητα αλλάζει η κοινωνία και θα αλλάξει και η εστίασή μας στην οδική ασφάλεια. Θέλουμε, έχουμε νέες ε, τάσεις ε, μεταφοράς στις πόλεις. Και τι σημαίνει αυτό για τους πιο ευάλωτους χρήστες. Θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι και οι συνέπειες των αυτόνομων οχημάτων. Θα πρέπει να ηγηθούμε της αλλαγή, αλλά η αλλαγή δεν θα πρέπει να παρεμποδίσει το στόχο μας για πλήρη εξάλληψη των θανατηφόρων τροχέων. Αυτό και προσβλέπω σε πολύ καρποφόρο συζήτηση. Σας ευχαριστώ και πάλι που θέσατε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εκ μέρους τώρα των πολιτικών ομάδων και πρώτα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για δύο λεπτά το λόγο έχει η κυρία Τούν. Σήμερα άνοιξα μια εφημερίδα και κοιτάξτε τι διάβασα. Τις πρώτες 40 ημέρες του έτους 100, 100 πεζοί σκοτώθηκαν από αυτοκίνητα και 60% 60% των ε, πεζών αυτών σε διαβάσεις. Ε, αγαπητέ Επιτροπέ και αγαπητέ Πρόεδρε, χαίρομαι που το βάλαμε το θέμα αυτό στη σημερινή συνεδρίαση, γιατί η ασφάλεια στον δρόμο είναι ένα θέμα ζωής και θανάτου, κυριολεκτικά. Και η κατάσταση στους ευρωπαϊκού δρόμους είναι δραματική. Πέρσι, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε Τι πιο αυστηρέ προδιαγραφέ για οχήματα, τον κανονισμό για τη γενική ασφάλεια. Θα το θυμάστε. Θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2022 και σκοπό έχει να μειώσει σημαντικά τον αριθμό θανάτων στους δρόμους. Αλλά πολλοί διατείνονται ότι ακόμα και πιο καλές τεχνικές λύσεις δεν πρόκειται να βελτιώσουν την κατάσταση στους δρόμους μας αν οι χρήστες, οι οδηγοί, συμπεριφέρονται με ανεύθυνο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να εκπαιδεύσει του οδηγού ακούμε συχνά, αλλά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δυστυχώ δεν έχουν αρμοδιότητα σε τέτοια εκπαιδευτικά συστήματα, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στην διοργάνωση α, μαθημάτων, κύκλων μαθημάτων για του ε, ανθρώπους που μαθαίνουν οδήγηση. Συνάδελφοι, Επιτροπέ, θα πρέπει να συνεργαστούμε πολύ πιο στενά με τα κράτη-μέλη για να πετύχουμε πραγματική, σημαντική μείωση των θάνατων στους δρόμους. Και ναι, Επιτροπέ, είναι στόχος μας να πετύχουμε αυτό το όραμα των μηδενικών ατυχημάτων. Να προετοιμάσουμε λοιπόν έναν οδικό χάρτη για το πώς θα το πετύχουμε αυτό το συντομότερο δυνατόν. Και έχουμε θετικά παραδείγματα από το Λονδίνο, το Ελσίνκι, το Όσλο, τέτοιες πόλεις που κατάφεραν να σταματήσουν τους θανάτους από οδικά ατυχήματα. Ας ε, Εποφεληθούμε λοιπόν όλοι από τις επιτυχίες αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες για τρία λεπτά, μισή λεπτά μάλλον το λόγο έχει ο κύριος Ντάνιελσον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Να ευχαριστήσω και την Επιτρόπο Βάλεαν για την εισαγωγή της. 500 άτομα χάνουν τη ζωή τους στους ευρωπαϊκούς δρόμους κάθε εβδομάδα. Λες και χάνουμε δύο αεροπλάνα τζάμπο κάθε εβδομάδα στην Ευρώπη. Θα ήταν εντελώ απαράδεκτο αυτό υπό άλλε συνθήκε. Αλλά τα αριθμητικά στοιχεία αυτά πραγματικά είναι απαράδεκτα και σε παγκόσμιο επίπεδο τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. 6.000 άτομα χάνουν τη ζωή τους, νέοι ε, κυρίω, αλλά και ε, κυρίω άτομα από χώρε ε, χαμηλόμιστες και παρά το γεγονό ότι έχουμε βελτιώσει την κατάσταση, τα αριθμητικά στοιχεία παραμένουν πολύ υψηλά ακόμα και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να μπει σε υψηλότερο σημείο στι προτεραιότητέ μα η ασφάλεια στου δρόμου. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να πετύχουμε ακριβώ αυτό το μηδενικό στόχο, τον οποίο ανέφερε η κυρία Βαλεάν, και να συνεχίσουμε να δίνουμε σημασία στο θέμα αυτό. Και επίση ε, οι βιώσιμοι στόχοι του ΟΗΕ θα πρέπει να επιτευχθούν. Αν κινηθούμε πιο γρήγορα, ίσως πετύχουμε κάτι παραπάνω. Και αν καταφέρουμε να μειώσουμε στο ίμιση τα οδικά ατυχήματα, ας το κάνουμε. Ο Τόμας Ένρου, το Υπουργό Συγκοινωνιών Μεταφορών στην ε, Σουηδία, θα διοργανώσει το συνέδριο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν ε, να βελτιώσουμε την ασφάλεια στους δρόμους για όλους, για τους οδηγούς, για τους πεζούς και για όλους όσου χρησιμοποιούν του δρόμου. ακόμα και για αυτούς που αναλαμβάνουν έργα στο δρόμο. Και όπως είπε και η Επιτροπή, πολλά από τα δικαιώματα αυτά μπορούν να προληφθούν. Θα πρέπει να φροντίσουμε να λαμβάνονται υπόψη πιο πολύ και οι αθώοι, οι πεζοί, οι ποδηλάτες. Όλοι θα πρέπει να αισθάνονται την ασφάλεια που τους αξίζει. Αν βελτιώσουμε λοιπόν και την ανάλυση της ταχύτητας, των ορίων ταχύτητας, θα βελτιώσουμε την ασφάλεια. Θα βελτιώσουμε και τις εκπομπές. Και έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε μέσω της οδικής ασφάλειας τους στόχους για το κλίμα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των υποδομών. Πάντα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πτυχή της ασφάλειας στους δρόμους και θα πρέπει να είναι πιο αυστηροί οι κανόνες και οι προδιαγραφές μας. Και αυτό το τελευταίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, παρά το γεγονό ότι το ίμιση του κόσμου στον πλανήτη μας είναι γυναίκες, φαίνεται ότι οι γυναίκες έχουν 70% πιο πολλές πιθανότητες να είναι θύματα αμα, ατυχημάτων, δυστυχημάτων. Πολύ απλά γιατί στα crash test δεν χρησιμοποιούμε προδιαγραφές που αφορούν γυναίκες. Χρησιμοποιούμε μοντέλα για άντρες. Να το βελτιώσουμε λοιπόν αυτό το στοιχείο, τα crash test, για να υπάρχει ασφάλεια εξίσου και για γυναίκες και για άνδρες. Άρα και στην οδική ασφάλεια τίφεται θέμα ισότητας. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η σημερινή συζήτηση θα στείλει ένα χειρό μήνυμα και στο συνέδριο που θα λάβει η χώρα την επόμενη εβδομάδα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε όμως για να πετύχουμε τους παγκόσμιους στόχους και για να διατηρήσουμε τα δικαιώματα των πολιτών. Και τέλος, να σας πω ότι όση ώρα μιλούσα σήμερα, εννέα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε δυστυχήματα στον δρόμο. Είναι πολύ υψηλό αυτό το τμήμα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να το μειώσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα εξ ονόματος της ομάδας Renew Europe για τέσσερα λεπτά ο κύριος Φλέγκο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Κάθε μέρα χάνουν ε, το δρόμ το, τη ζωή τους στις ευρωπαϊκούς δρόμους ε, ε, εκατοντάδες άνθρωποι. Και μάλιστα όλοι έχουμε κάποιον εκεί ο, η συγγενή μας που έχει χάσει τη ζωή του, μια οικογένεια που έχει μείνει ε, χωρίς κάποιο μέλος της. Είναι περιττή όλη αυτή οι θάνατοι. Έχουμε επίγνωση λοιπόν ότι θα πρέπει ε, και οφείλουμε είτε να μειώσουμε δραστικά τους θανάτους αυτούς είτε να τους εξαλείψουμε. Γιατί ε, παγκοσμίω, ε, ε, μάλλον στην Ευρώπη, λέει ο μιλητή, 1,35 εκατομμύρια άνθρωποι το χρόνο χάνουν τη ζωή του, μάλλον παγκοσμίω εννοεί. Και ε, είναι πολύ μεγάλος αριθμός των νέων που χάνουν τη ζωή του. Ήδη το 2018 5.000 έχασαν τη ζωή τους ε, στους δρόμους ε, το χρόνο και 135.000 έμειναν βαριά τραυματισμένοι. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε δράσεις. Βέβαια, ο μεσοπρόθεσμος ε, στόχος τη Ευρώπης είναι εκμηδανισμό των θανατηφόρων τροχαίων. Και ε, δυστυχώς έχουμε αναγνωρίσει πια ότι δεν πρόκειται να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Ίσως ήταν ε, υπερβολικές οι φιλοδοξίες μας και οι στόχοι μας και δεν πρόκειται να τους υλοποιήσουμε. Σίγουρα οι στόχοι θα πρέπει να δίνουν κίνητρα για την υλοποίησή τους, αλλά δεν θα πρέπει να είναι εξωπραγματικοί ή ουτοπικοί. Θα πρέπει να έχουμε πιο ρεαλιστικούς στόχους. Η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Κροατία είναι από τις χώρες που έχουμε διπλάσιο αριθμό θανατηφόρων ατυχημάτων σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο. Δεν σημαίνει ότι οι οδηγοί ε, στις χώρες αυτές δεν οδηγούν καλά ή δεν οδηγούν τόσο καλά όσο οι Σκανδιναβοί. Η αλήθεια είναι όμως ότι ε, στην Ρουμανία, Βουλγαρία και Κροατία έχουμε πολύ παλιότερα αυτοκίνητα σε πολύ χειρότερη κατάσταση και πολύ χειρότερες υποδομές αυτοκινητοδρόμων και δρόμων. Οπότε δεν πρόκειται να έχουμε επανάσταση στην ασφάλεια, στην οδική κυκλοφορία, αν δεν αξιοποιήσουμε καλύτερα την τεχνολογία στα οχήματα και αν δεν επενδύσουμε περισσότερο στις οδικές υποδομές. Γιατί η τεχνολογία υπάρχει, η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και εξαρτάται από όλους εμάς πόσο γρήγορα θα εφαρμόσουμε αυτές τις νέες τεχνολογίες. Οι νέες τεχνολογίες, η επιμερισμένη οικονομία, η συνεργατική οικονομία, η ε, οδήγηση ε, με αλληλέγγυα. Νομίζω ότι είναι τρόπος ε, για να μειώσουμε και τα θανατηφόρα τριχεία, αλλά κυρίως να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να βελτιώσουμε την υγεία των πολιτών. Και με τη ρομποτική και τις νέες τεχνολογίες μπορούμε να μειώσουμε το ανθρώπινο λάθος, που είναι η αιτία του 90% περίπου των τροχαίων ατυχημάτων. Μπορούμε λοιπόν ε, στο όραμά μας ε, για μηδενικά θανατηφόρα τυχαία μέχρι το 2030 ε, να προβλέψουμε τα απαραίτητα κονδύλια στα κράτη-μέλη, να βελτιώσουμε τις υποδομές και να βελτιώσουμε την τεχνολογία και την ασφάλεια των οχημάτων. Έτσι θα μειώσουμε στο έπακρο ή όσο είναι δυνατό τον αριθμό των ατυχημάτων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να μειώσουμε και τη φορολογία στα πιο οικολογικά ατυχήματα και να βελτιώσουμε το τεχνολογικό έλεγχο και την ε, κατάσταση των οχημάτων. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ένα σημαντικό τμήμα τη αγώνα μας για τη βελτίωση της ασφάλειας. Θα πρέπει φυσικά να λάβουμε υπόψη τις υποδομές και τις νέες τεχνολογίες, αλλά ας μην ξεχνούμε ότι η μεγαλύτερη, ο μεγαλύτερος κίνδυνος στους δρόμους είναι μερικές φορές οι νέοι οδηγοί, οι νέοι οδηγοί που δεν έχουν ε, αντιληφθεί πόσο σημαντική είναι η υπεύθυνη οδήγηση. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω κύριε Επίτροπε να θέσετε την οδική ασφάλεια και δική σας προτεραιότητα και στην οδική κυκλοφορία και στην κυκλοφορία όχι μόνο των γεωταχειοχημάτων αλλά και των φορτηγών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματο των Πρασίνων, Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, για 2,5 λεπτά η κυρία Μέτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Επιτροπέ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε εβδομάδα 500 άνθρωποι χάνουν τη ζωή του στους δρόμου μας. Δύο γεμάτα λοιπόν αεροπλάνα τα οποία χάνονται. Ποτέ λοιπόν ε, δεν θα αποδεχόμαστε τόσου πολλού νεκρού ε, σε αεροπορικά δυστυχήματα. Γιατί τα δεχόμαστε λοιπόν στα οδικά δυστυχήματα. Κάθε χρόνο εκτιμάται ότι χάνουμε 280 δις ευρώ σε τέτοιε ε, δυστυχήματα. Πέραν από την ανθρώπινη τραγωδία. Γι' αυτό λοιπόν καλωσορίζω τι υποσχέσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπει η οδική ασφάλεια στο πλαίσιο αυτό ε, να μειωθούν στο ίμιση οι θάνατες στους δρόμους. Θα είναι αυτό κλειδί για το Vision Zero, για το μηδενικό αριθμό τέτοιων ατυχημάτων μέχρι το 2050. Με τις τεχνολογικές λοιπόν εξελίξεις και την ε, τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά η ασφάλεια στους δρόμους. Γιατί 94% των ατυχημάτων έχουν να κάνουν με ανθρώπινο σφάλμα. Ένα αυτοματοποιημένο λοιπόν σύστημα οδικής κυκλοφορίας θα φέρει νέες προκλήσεις και νέα προβλήματα και θα κληθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Νέες υποδομές, για παράδειγμα, για τα ε, οχήματα αυτόνομης οδήγησης και αυτό θα, θα συνεπάγεται με τη σειρά του και άλλες συνέπειες ότι αφορά το περιβάλλον, το κλίμα. Σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τους πεζούς, οι οποίοι είναι ε, άτομα τα οποία είναι στο μεγαλύτερο κίνδυνο. Ένα τρίτο των θυμάτων. Για να αυξήσουμε λοιπόν την ασφάλεια στους δρόμους χρειαζόμαστε ένα νέο ε, πολυαδομικό σχεδιασμό για να υπάρχει πραγματικά προτεραιότητα για τους πεζούς και χρειαζόμαστε λοιπόν μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη κινητικότητα και μεταφορές. Όπως ε, λέτε κυρία, Επιτρόπε και χαίρομαι, έχετε μια στρατηγική, αλλά η στρατηγική πρέπει να συνοδεύεται και από μέτρα και ελπίζω να τηρήσετε το λόγο σας και η οδική ασφάλεια τα επόμενα χρόνια να καταστεί πραγματικά σημαντική προτεραιότητα για σας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ και εξ ονόματος των Ευρωπαϊκών Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών για 1,5 λεπτό το λόγο έχει ο κ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Επίτροπε. Η ενίσχυση του επίπεδου ασφάλειας των χρηστών της οδικής κυκλοφορίας, δηλαδή των οδηγών, των πεζών ή των ποδηλατών, είναι τεράστια πρόκληση και για τα κράτη-μέλη και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξετάζοντας τις στρατηγικές, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τη γεωγραφία και οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές είναι αυτές που έχουν τις χειρότερες επιδόσεις. Περίπου 55% των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων λαμβάνει η χώρα στις επαρχιακές οδούς. Και νομίζω ότι αυτό ίσω είναι το καλύτερο επιχείρημα υπέρ τη συνέχιση μια φιλόδοξη πολιτική συνοχή που θα επιτρέπει στην τοπική αυτοδιοίκηση να επενδύει σε ασφαλείς ε, υποδομέ και σε δημόσιες συγκοινωνίες. Ε, τεράστιο στήριγμα για του οδηγού είναι και η τεχνολογία για τα προηγμένα συστήματα ασφάλεια στα οχήματα. Επόμενο βήμα θα είναι σίγουρα τα οχήματα που θα είναι πλήρως αυτόνομα. Βέβαια αυτό το θέμα αφορά περισσότερο το μέλλον. Θα πρέπει όμως να ενθαρρύνουμε τους οδηγούς και κυρίως τους νέους να οδηγούν με υπεύθυνο τρόπο και θα πρέπει στις δράσεις αυτές να εμπλέξουμε και τις ασφαλιστικές εταιρείε που έχουν τρόπους να επιβραβεύουν την ασφαλή συμπεριφορά στο δρόμο. Είμαι πεπισμένο ότι σε ό,τι δράση αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ενισχύσει την οδική ασφάλεια και να εξαλείψει μέχρι το 2050 τα θανατηφόρα τροχαία οχήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υπολογίζει στην αμέριστη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Νοτικής Αριστεράς. Για τρία λεπτά, κυρία Κουντουρά. Πολύ, κυρία Πρόεδρε βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το οφείλουμε στα θύματα να σχεδιάσουμε φιλόδοξες πολιτικές και να υπενθυμίζουμε σε κάθε ευκαιρία ότι για το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο η οδική ασφάλεια είναι μέγιστη προτεραιότητα. στην ευρώπη έχουμε σήμερα 500 νεκρούς την εβδομάδα παρόλο που οι δρόμοι μας είναι οι ασφαλέστεροι στον κόσμο ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε δύο αεροπορικά δυστυχήματα την εβδομάδα στην ευρώπη ή στον αφανισμό μιας μικρής πόλης 26.000 κατοίκων το χρόνο. δυστυχώς όμως τα θύματα στους αυτοκινητόδρομους δεν ενεργοποιούν ανάλογα τα αντανακλαστικά ούτε των μέσων μαζικής ενημέρωσης ούτε της κοινωνίας μας και των πολιτικών μας. η κατάσταση αυτή πρέπει να ανατραπεί ακόμα και αν δεχτούμε ότι τα ανθρώπινα λάθη δεν θα εκλείψουν ποτέ οραματιζόμαστε τη μείωση των ατυχημάτων και κυρίως μηδενικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. το κλειδί είναι να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. ακούσαμε και από τις άλλες πολιτικές ομάδες ότι θέλουν και αυτές φιλόδοξες πολιτικές αλλά αναρωτιέμαι αν οι προθέσεις τους είναι ειλικρινείς γιατί δεν στήριξαν το αίτημά μας για τη σύνταξη ενός ψηφίσματος για την οδική ασφάλεια θα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να τοποθετηθεί το νέο κοινοβούλιο για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα και να το φέρει στην επικαιρότητα εν ώψη μάλιστα της τρίτης παγκόσμιας υπουργικής διάσκεψης στη στοκχόλμη. πρέπει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο να είναι πρωτοπόρο στην οδική ασφάλεια στην πράξη και σας καλώ ως πρώτο βήμα να αναθεωρήσετε τη στάση σας και να στηρίξετε συγκεκριμένες προτάσεις όπως να επαναλάβουμε τη δέσμευσή μας στο ευρωπαϊκό στόχο για τη μείωση στο μισό του αριθμού θανάτων και σοβαρών τραυματισμών από το 2020 χιλιάδες έως το δύο και το μηδενισμό των θανάτων έως το. 2050 να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκά προγράμματα στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο με στόχο την προώθηση πολιτικών που αποδεδειγμένα έχουν θετικά αποτελέσματα ειδικά προγράμματα που στοχεύουν στη μείωση των μεγάλων ανισοτήτων ανάμεσα στα κράτη μέλη σε επιδόσεις οδικής ασφάλειας εκεί δηλαδή που υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης να αξιοποιήσουμε τις τελευταίες καινοτομίες της αυτοκινητοβιομηχανίας σε συστήματα ασφαλείας σε νέα αλλά και παλαιά οχήματα όπου αυτό είναι δυνατό να θέσουμε στόχους για τη μείωση των θανάτων ευάλωτων χρηστών του δικτύου στο πλαίσιο της αστικής κινητικότητας να θεσπίσουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τα οχήματα με αυτοματοποιημένα συστήματα οδήγησης να ενισχύσουμε την εφαρμογή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και διασυνοριακά. η επίτροπος ε, Βάλεαν έχει εκφράσει ήδη δύο φορές στην επιτροπή μεταφορών τη δέσμευσή της όπως και σήμερα εδώ στο κοινοβούλιο να εργαστεί ενεργά για πιο ασφαλείς δρόμους στην ευρώπη και την ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου γι' αυτό πρέπει και εμείς λοιπόν στο κοινοβούλιο να ξεκαθαρίσουμε τις προτεραιότητές μας και να συνεργαστούμε με επιτροπή και κράτη μέλη ώστε τα επόμενα χρόνια να μπουν τα θεμέλια για μια επιτυχημένη στρατηγική και ένα φιλόδοξο νομοθετικό πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να πετύχουμε το στόχο μείωσης κατά το ίμιση των θανάτων και σοβαρών τραυματισμών το. 2030. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής για δύο λεπτά, ο κύριος ε, Λούτκεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τη δήλωσή σας. Η στρατηγική που εγκρίθηκε τον περασμένο Ιούνιο έχει στόχο να μειώσει κατά το ίμιση τα θανάσιμα τροχαία ατυχήματα στους δρόμους. Ένας ε, συγκεκριμένος στόχος ε, ανθρώπινος και δυστυχώς όλοι γνωρίζουμε τραγικές περιπτώσεις οικογενειών που καταστράφηκαν λόγω ε, της πραγματικότητας της οδικής ασφάλειας και των δρόμων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε μια σειρά επιλογών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει και το ε, επιθυμό μια αναθεώρηση της άδεια οδήγησης, επίσης ε, αναθεώρηση της διασυνοριακής συνεργασίας, κυρίως σε περίπτωση Απόσυρση τη άδεια οδήγηση, ε, περιορισμό επίσης κατανάλωση αλκοόλ, ε, ναρκωτικών ή ακόμα και τις ε, ταχύτητε. Πρόκειται για τρεις διαδικασίες που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές, οι οποίες ίσως πέρα το στόχο θα μπορέσουν να επιφέρουν και συγκεκριμένα μέτρα για να βελτιώσουμε την κατάσταση τη οδικής ασφάλεια στην Ευρώπη. Αν δούμε λίγο καλά τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια στασιμότητα στα στοιχεία για την οδική ασφάλεια και αυτό είναι λυπηρό. Υπήρξε μια βελτίωση τα τελευταία χρόνια και τώρα έχουμε μια καθίζηση και φυσικά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η καθίζηση γιατί έχουμε συγκεκριμένου ε, στόχους για τη μείωση των ε, θανατηφόρων ε, ατοχημάτων και των τραυματιών. Ε, χρειαζόμαστε επίση συγκεκριμένε καλέ πρακτικέ ε, ανακράτο μέλο. Ε, πρέπει μαζί να θέσουμε τα κατάλληλα ερωτήματα. Φυσικά δεν είναι παντού τα μέτρα ίδια στη κράτη-μέλη. Πρέπει σε κάποια κράτη-μέλη να εφαρμοστούν και συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση Τη ε, πραγματικότητα τη οδικής ασφάλειας και φυσικά των στατιστικών στοιχείων. Υπάρχουν πολλά ε, στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και πολύ μεγάλε διαφορέ μεταξύ κρατών μελών και πραγματικά επιθυμώ, κυρία Επίτροπε, να μπορέσουμε να εργαστούμε από αυτόν και να πιέσετε κι εσείς και να πιέσουμε κι εμεί ώστε να κάνουμε συστάσεις, να καθορίσουμε συστάσεις αναχώρα, ώστε να εφαρμόζονται καλέ πρακτικέ παντού και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη μοίρα τη οδική ασφάλεια παντού στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια για 1,5 λεπτό η κυρία Μαλτονάδο Λόπεθ. Παρακαλώ. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε που έχετε φέρει εδώ στην Ολομέλεια μια συζήτηση η οποία θεωρώ ότι είναι θεμελιώδης. Ε, πολύ συχνά μιλάμε για πάρα πολλά πράγματα και θέματα όπως είναι η οδική ασφάλεια που είναι θεμελιώδες θέμου στην καθημερινότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά και με τους συμπολίτες μας. Όπως πολύ σωστά είπε η Επίτροπος, πάνω από 500.000 ε, άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο στην Ευρώπη. Το 90 100 των τροχιών ατυχημάτων στην Ισπανία είναι από ανθρώπινο σφάλμα. Και εκεί θα πρέπει να επικεντρώσουμε τι προσπάθειέ μα ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ω ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα πρέπει να ενώσουμε τι δυνάμει μα ε, στα θεσμικά όργανα, αλλά και φυσικά και μεταξύ κρατών. Εγώ πιστεύω ότι οι νέε τεχνολογίε θα διαδραματίσουν και ένα ουσιαστικό ρόλο. Ένα ρόλο κλειδί, γιατί πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ήδη δημιουργούνται νέα μοντέλα αυτόνομων οχημάτων. Ο ανθρώπινο κίνδυνο βλέπουμε ότι είναι ο βασικό παράγων στα τροχαία ατυχήματα και πρέπει να προσπαθήσουμε να το μειώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και πρέπει να είμαστε και έξυπνοι και να εκμεταλλευτούμε τι νέε τεχνολογίε, όπω για παράδειγμα την τεχνητή νοημοσύνη, ώστε αυτό ο ανθρώπινο κίνδυνο να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο στα τροχαία ατυχήματα. Διότι πρόκειται για τη ζωή ε, πάρα πολλών ανθρώπων. Και φυσικά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την ψηφιοποίηση για να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό το μεγάλο αριθμό θυμάτων. Πιστεύω ότι πρόκειται για πραγματική πρόκληση για την ε, ε, ενιαία αγορά. Πρέπει να είμαστε, για παράδειγμα, σε θέση να δημιουργήσουμε και να εγγυηθούμε ασφάλεια δικαίου, να γίνουν επενδύσεις στις αντίστοιχες τεχνολογίες και επίσης να προστατεύσουμε και τους ε, πολίτες και τους καταναλωτές από τις προκλήσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η ψηφιοποίηση είναι μια πολύ καλή λύση ώστε να καταφέρουμε να έχουμε ε, μια καλή αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό, ο κύριος Τζαμπάσκι. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σήμερα βλέπουμε ότι έχουμε περισσότερους ε, ευρωβουλευτές στην αίθουσα της Ολομέλειας τέτοια ώρα. Αυτό είναι πολύ θετικό και δείχνει πόσο σημαντικό είναι για μας το θέμα. Μάλιστα έχω και προσωπική πείρα και μπορώ να αναλύσω το θέμα αυτό, γιατί για πολλούς το ζήτημα της οθικής ασφάλειας είναι κάτι απομακρυσμένο. Γιατί η οθική ασφάλεια δεν σημαίνει μόνο να φοράμε ζώνες ασφαλείας ή να μην χρησιμοποιούμε το κινητό μας όσο οδηγούμε. Έχουμε ανάγκη και από προληπτικά μέτρα. Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη του οδηγού και όλων των χρηστών των οδικών αποδομών. Στην πατρίδα μου, τη Βουλγαρία, πάνω από 682 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε τροχέα. Και μάλιστα θεωρώ ότι δεν είναι ακριβή αυτά τα νούμερα. Εδώ μιλούμε για θανάτους μόνο, όχι για τραυματισμούς που μπορεί στη συνέχεια να άλλαξαν τη ζωή των θυμάτων. Και στη Βουλγαρία έχουμε πολύ περισσότερα τροχαία ατυχήματα από ότι ε, θανάτου σε χώρε που έχουν ένοπλε σειράξει. Αυτό είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό και λέω ότι η οδική ασφάλεια είναι πολύ πιο σημαντικό θέμα από άλλα που συζητούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως είναι η καμπύλη των αγκουριών ή άλλε λεπτομέρειε. Θα πρέπει να εναρμονίσουμε επίση τα οδικά σήματα. Αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Κύριε Επίτροπε, κύριε Βαλεάν, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και εσείς ε, είστε αρμόδια επίτροπος για πολλά από τα θέματα αυτά. Επίσης, θα πρέπει να μην ε, επιμείνουμε σε αυτή την αλλοπρόσελη ιδέα να επιστρέφουν τα φορτηγά άδεια στη χώρα καταγραφής. Πριν από λίγο άκουσα ε, ότι τα crash test δεν είναι προσαρμοσμένα στις γυναικείες προδιαγραφές. Δεν νομίζω ότι οι γυναίκε είναι καλύτεροι ή χειρότεροι για του άντρε. Θα έχουμε αυστηρότερου κανόνε για όλου. Κύριε Τζαμπάσκε, δέχεστε μια ερώτηση με τη διαδικασία τη μπλε κάρτα από την κυρία Τούν. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τζαμπάσκη. Πότε τελευταία συζητήσαμε για τις καμπύλες των αγκουριών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί εγώ είμαι 11 χρόνια ευρωβουλευτής και ουδέποτε δεν συμμετείχα σε τέτοια συζήτηση πότε τελευταία ασχοληθήκατε με το θέμα αυτό, πώς είναι η ειδικότητα του ECR, εσείς πότε τα συζητήσατε αυτά. αδελφέ. να σας υπενθυμίσω ότι την προηγούμενη θητεία εδώ στην αίθουσα αυτή, στην Ολομέλεια, ψηφίσαμε τα συστατικά για τις σάλτσες ντόνερ. Το θυμάστε? Ε, ναι ή όχι. Δεν είναι σημαντικό ζήτημα αυτό. Το ζήτημα που συζητάμε σήμερα είναι πολύ πιο σημαντικό. Και να σας υπενθυμίσω επίσης σε ό,τι αφορά την καμπύλη και του αγκουριού και τις σάλτσες ε, ντόνερ, γιατί μπορεί να τα έχετε ξεχάσει όλα αυτά, αλλά δεν έχουν να κάνουν τίποτα όλα αυτά με τη σημερινή μας συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής για 1,5 λεπτό, η κυρία Λουκατσιεύσκα. Ευχαριστώ. Αναφίβολα, το θέμα της οδικής ασφάλειας είναι σημαντικό ε, θέμα για την κοινωνία. 200, εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν άδεια οδήγησης και όλοι οι πολίτες χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους για να πάνε στη δουλειά τους και την τελευταία δεκαετία τριπλασιάστηκε η οδική κυκλοφορία Αυξήθηκαν βέβαια και οι δαπάνε στις υποδομές, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούμε να έχουμε υψηλό βαθμό θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη το οικονομικό αυτό και κοινωνικό πρόβλημα και να ενισχύσουμε την οδική μας ασφάλεια. Χαίρομαι ιδιαίτερω που η οδική ασφάλεια αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσβλέπω στην ε, μεγάλη στράτευση της ε, Επιτρόπου υπέρ της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας. Και επίσης χαίρομαι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε και τις νέες τεχνολογίες για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Η ε, επιρροή των ε, νέων τεχνολογιών θα είναι τόσο σημαντική αντίστοιχη με την τεράστια θετική επίπτωση που έχει χρήση των ζωνών ασφαλείας στο παρελθόν. Επίσης, ε, πιο φτωχές χώρες ή λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές με κακές οδικές υποδομές έχουν και τα περισσότερα θανατηφόρα τροχέα. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και επίσης είναι πολύ σημαντική επιμόρφωση, η σωστή παιδεία ε, είναι απαράδεκτο κάποιος μετά από χρήση ινοπνεύματος, αλκοόλ ή ναρκωτικών να παίρνει το αυτοκίνητό του και να οδηγεί. Είναι απαράδεκτο, θα πρέπει να λάβουμε πιο αυστηρά μέτρα και να περιορίσουμε τέτοιες τραγωδίες όπως είναι τα τροχαία ατυχήματα. Και μπορείτε να, έχετε την εμπιστοσύνη ε, να είστε σίγουροι ότι θα έχετε την αμέριστη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και έχω ένα αίτημα για τη διαδικασία Catch the Eye. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Ζούντσα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως η οδική ασφάλεια είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μακρύ δρόμο μπροστά της για να ενισχύσει την οδική ασφάλεια, γιατί έχουμε πολλά θανατηφόρα τροχέα και έχουμε ε, πολιετή συνέπειες από τραυματισμούς σε τροχέα, ε, τεράστια έξοδα και ιατρικά και μεγάλη επίδραση στη ζωή του τραυματία. Έχουμε πολλά λοιπόν μπροστά μας να κάνουμε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω μία έκθεση που είναι, κάνει μία συγκριτική ανάλυση των χωρών μελών σε ό,τι αφορά το επίπεδο των θανατηφόρων τροχαίων. Και σίγουρα το μεγαλύτερο ρυθμό τροχαίων έχουμε στις χώρες ε, τις μετακομμουνιστικές, γιατί εκεί λόγω κακών υποδομών είναι πολύ περισσότερα τα τροχαία ατυχήματα. Οπότε δεν θα πρέπει να αφιστούμε προσπαθειών ούτε επενδύσεων για να βελτιώσουμε τις υποδομές. Το, την οδό των Καρπαθίων. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τι υποδομέ χώρε τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. γιατί στους δρόμους αυτούς, Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη έχουμε τα περισσότερα τροχέα, δυστυχώς. Έχετε πολύ δύσκολο δρόμο μπροστά σα και δύσκολη αποστολή. Καλή σα τύχη. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή. Έχετε το λόγο, Επιτροπή Βαλεάνα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτέ. Ε, Εκτιμώ ιδιαίτερα τα σχόλιά σα και το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται για το θέμα αυτό. Όπω είπα εξ αρχή, συνεργαζόμαστε και ασκούμε επαρκή ε, πίεση σε όλου του εμπλεκόμενου φορεί από του οποίου ε, εξαρτάται το κατά πόσον η ασφάλεια στους δρόμους θα έχει τα αποτέλεσματα που επιθυμούμε. Για παράδειγμα, αναφέρατε τους στόχους. Τους στόχους ε, οι οποίοι εκπνέουν, όπως σας είπα, φέτος και ενδεχομένως θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί γιατί έχουμε αυτούς τους στόχους αφού δεν τους πετυχαίνουμε. Είναι σημαντικό όμως εργαλείο η στόχη αυτή για να μπορέσουμε να καταρτήσουμε τις πολιτικές μας και να ξεκινήσουμε τον διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να πετύχουμε ε, συγκεκριμένο όραμα για το μέλλον στους διάφορους τομείς. Και εγώ λοιπόν ε, είμαι υπέρ του να διατηρήσουμε ένα σαφή στόχο βάσει του οποίου θα μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε τις ε, δράσεις μας για το μέλλον δεν ε, χρειάζεται και όλοι σας αναφερθήκατε στα αριθμητικά στοιχεία όπως και εγώ άλλωστε στην αρχή να επαναλάβω ότι οποιαδήποτε αριθμός δεν είναι αποδεκτός όπως είπατε Α, επίσης δεν είναι αποδεκτό το, το γεγονός ότι είναι κάτι τετριμένο και συνηθισμένο το να ακούμε αριθμούς θυμάτων στους δρόμους χρειάζονται κατεπηγόντω δράση και θα πρέπει να δεσμευτούμε προ την κατεύθυνση αυτή. Αναφέρατε πολύ από εσά το πόσο ευάλωτη είναι η πεζή και άλλες κατηγορίες πολιτών στην κυκλοφορία. Όταν μιλάμε λοιπόν για θέματα ασφάλειας, ε, στο επίκεντρο θα πρέπει να είναι ο άνθρωπος, ο πολίτης. Και έχουμε διάφορες κατηγορίες ε, ευάλωτων χρήστων του δρόμου. Και οι πεζοί, αλλά και οι ποδηλάτες. Οι μοτοσυκλετιστές. Πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε τρόπους για τη βελτίωση της ασφάλειας και μέσα στις πόλεις μας. Το πρόβλημα είναι, και το ξέρουμε όλοι μας, εκεί που συναντιόνται όλες οι κατηγορίες. Και τώρα με την εξέλιξη της τεχνολογίας βλέπουμε και ένα νέο κύμα κινητικότητας μέσα στις πόλεις και βλέπουμε λοιπόν ότι τέτοιου είδους κίνδυνοι είναι ακόμα πιο υψηλοί. Θα πρέπει λοιπόν ε, να βρούμε τη σωστή πολιτική εγκαίρως για να προστατεύσουμε αυτές τις κατηγορίες οι οποίες θα συναντηθούν όλες στον ίδιο χώρο ουσιαστικά. Και μιας και συζητάμε τα θέματα αυτά, να αναφερθώ και σε ένα θέμα το οποίο το ακούσαμε από πολλούς σας. Ε, η αυτοματοποίηση και η ψηφιοποίηση μπορούν να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την ασφάλεια στους δρόμους και πολλοί αναφέρατε το θέμα των αυτόνομων οχημάτων στο μέλλον. Το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης αυτό συνεπάγεται και τεράστιες προκλήσεις όμως, γιατί ομολογούμε ότι η αρχή της ε, χρήσης των οχημάτων αυτών με την σταδιακή ε, εξέλιξη της υποδομής θα πρέπει να συνάδει με τις συμβατικές μεθόδους ε, μεταφοράς. Αυτό λοιπόν στην αρχή θα αποτελέσει ένα νέο κίνδυνο για την ασφάλεια στους δρόμους. Αυτό αποτελεί λοιπόν ένα νέο στοιχείο το οποίο το εξετάζουμε και αυτό. Το σύστημα ασφάλειας πιστεύω ότι θα πρέπει να το κοιτάξουμε συστηματικά. Γιατί ακριβώς έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία που καθιστούν την ασφάλεια στους δρόμους, ε, μεγάλη πρόκληση. Και πολλοί από, από εσά αναφερθήκατε και στο θέμα της ε, έκδοσης ε, διπλωμάτων οδήγηση. Κάποιοι αναφερθήκατε στα θέματα ταχύτητας. Όλα αυτά τα κοιτάμε μέχρι το 2022. Για το θέμα της ταχύτητας να σας δείξω ένα άλλο αριθμητικό στοιχείο από το EDSC, ένα αριθμητικό στοιχείο. Ένα χιλιόμετρο το χρόνο μείωση στην μέση ταχύτητα, μόνο ένα χιλιόμετρο μείωση της μέσης ταχύτητας, θα μείωνε τους θανάτους κατά 2.000 το έτος. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικός παράγοντας είναι η ταχύτητα. Αναλύουμε λοιπόν τα στοιχεία αυτά και κοιτάμε πώς μπορούμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν για να δράσουμε όλοι μαζί από κοινού προς την κατεύθυνση αυτή. Το 2017 είχαμε τη δήλωση, την διακήρυξη της Βαλέτας για την ασφάλεια στους δρόμους και τη δέσμευση των ε, Υπουργών για τη δυνατότητα μείωσης των ορίων ταχύτητας. Να δούμε λοιπόν πού έχουμε φτάσει στο θέμα αυτό. Μία μεμονωμένη ανάλυση που γίνεται ένα κράτος μέλος είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Κράτο μέλο, ένα κράτο μέλο, λοιπόν. Να την κοιτάξετε και να συζητήσουμε τα θέματα αυτά μετά την ετήσια έκθεση και τα στατιστικά στοιχεία τα οποία θα δημοσιευτούν τον Απρίλιο. Και επίσης να σας υπενθυμίσω ότι μετά τη διάσκεψη της Στοκχόλμης, δεσμεύομαι γι' αυτό, την επόμενη μέρα νομίζω θα μεταβώ στην Επιτροπή Μεταφορών και θα σας ενημερώσω για το τι δεσμεύσεις αναλήφθηκαν στη Στοκχόλμη και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε στο μέλλον για να αυξήσουμε την ασφάλεια στους δρόμους της Ευρώπης γιατί όχι να μην μπούμε στην ηγεσία στο θέμα αυτό και να ηγηθούμε όλων των άλλων υπήρων, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα project για την Ασία και την ε, Αφρική, προκειμένου τελικά να μειωθούν οι θανατηφόρες, ε, θανατηφόρα δυστυχήματα σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για τη σημερινή συζήτηση και πάντα είμαι στη διάθεσή σας και για το θέμα αυτό και για άλλα θέματα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα ενθαρρυντικά σας λόγια και με αυτό θα ήθελα να κλείσω τη συζήτηση. Τα πρακτικά της συνεδρίασης θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο προς έγκριση στις αρχές της επόμενης ε, ε, συνόδου και αν δεν υπάρχουν ενστάσεις ε, μαζί με τα ψηφίσματα τα οποία εγκρίθηκαν στη συγκεκριμένη σύνοδο η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται και κλείνει η συνεδρίαση. Καλό σας απόγευμα.